So, ladies and gentlemen and dear colleagues, uh, let's Ξεκινάμε την επόμενη συνεδρίαση της ε, Επιτροπής ΙΝΤΑ. Λόγω του ότι έχουμε την Δικούς Επιτροπή του ΠΟΕ σήμερα, έχουμε καλεσμένους μαζί μας εδώ. Ε, θέλω συγκεκριμένα να καλωσορίσω τον κύριο Γέλμαν, τον οποίο όμως δεν βλέπω. Είναι, είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποσχέσεων της Βουλής των, του Καζακστάν. Το Καζακστάν θα ε, φιλοξενήσει την Υπουργική του ΠΟΕ και την ε, Κοινοβουλευτική του ΠΟΕ. Θέλω λοιπόν να, τους να τον καλωσορίσω. Επίσης, το πρώτο θέμα της ημερήσιας ε, διάταξης είναι το 16. Η επιβολή, ο κανονισμός για την εφαρμογή. Σημαντικό ζήτημα, κυρίως δεδομένης της κατάστασης του ΠΟΕ, όπου δεν έχει αυτή τη στιγμή ε, όργανο προσφυγών το οποίο να λειτουργεί και ως εκ τούτου πρέπει να αποφασιστεί πώς θα αντιδράσουμε. Η συγγήτρια είναι η, ε, η Μαριπιέρ Της δίνω το λόγο. Πέρυσι, πέρυσι έκανε μια αναθεώρηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους κανόνες ε, του ε, διεθνούς εμπορίου μετά από το μπλοκάρισμα του οργάνου προσφυγών του ΠΟΕ. Αυτό αποτελεί το 2014 τον, ε, τη νομική βάση που επιτρέπει την προσφυγή μιας χώρας ε, ε, στον ΠΟΕ. Ως εκ τούτου η κατάσταση έχει οδηγήσει την, την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια κατάσταση που είναι νομικού κενού. Η πρόταση λοιπόν αποτελεί νομική βάση και επιπλέον μας επιτρέπει να υπενθυμίσουμε τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ΠΟΕ και στο πολυμερές σύστημα. Γι' αυτό την ευχαριστούμε. Επίσης, αφορά τις κανόνες ελεύθερων συναλλαγών της Ένωσης σε περίπτωση διευθέτηση διαφορών. Πρόκειται για μια καλή θετική πρόοδο που επιτρέπει την ουσιαστική υλοποίηση της εμπορικής πολιτικής και της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών. Θα ήθελα σήμερα να γίνει μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για να ακούσω τις απόψεις των συναδέλφων επί των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να συμπληρώσουμε και να κάνουμε πιο αποτελεσματικό το όργανο εμπορικής πολιτικής. Είναι καλή αυτή η πρόταση, την οποία μπορούμε να τροποποιήσουμε για να συμπεριλάβουμε και την πνευματική διοκτησία και τις υπηρεσίες στο πεδίο εφαρμογή. Είναι η πρόταση ήδη των βουλευτών από την προηγούμενη θητεία πνευματική ιδιοκτησία είναι αναπόσπαστο μέρος της οικονομίας μας και αν ε, συμπεριληφθούν αυτά θα μπορέσουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί με αποτρεπτικά μέτρα. Λοιπόν, θα ήθελα να ακούσω τις παρεμβάσεις των συναδέλφων και ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που, βρίσκεται, που επιτρέπει αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Γιάμανδε. Δέα. στην Επιτροπή μας καλή τύχη για την ε, προετοιμασία του, της διάσκεψης ε, του ΠΟΕ. Καλώς ορίσατε. Οπότε, δίνω το λόγο τώρα στους σκιώδεις εισηγητές. ΕΛΚ δεν παρίσταται. Σοσιαλιστές και Δημοκράτες ε, θα φορέσω το άλλο μου καπέλο και θα γίνω εγώ ο σκιώδης ομιλητής μπορώ να συμφωνήσω με την εισηγήτρια η οποία υποστηρίζει τον κανονισμό. Πράγματι είναι σημαντικό να είναι ξεκάθαρη η θέση μας ε, σε, μια, σε ένα χώρο που έχει κλιμακωθεί. Κατά την άποψή μου, ο, το πεδίο εφαρμογή του κανονισμού είναι υπερβολικά περιορισμένο, γιατί ουσιαστικά συζητά την περίπτωση που δεν θα υπάρξει απόφαση του ε, οργάνου προσφυγών. Όμως υπάρχουν φήμες ότι ένας μεγάλος εμπορικός εταίρος δεν έχει ε, τηρήσει τους κανόνες των δασμών του 95. Και αν υπάρξει πρόβλημα στο διεθνές σύστημα εμπορίου βάση κανόνων, θα πρέπει να αντιδράσουμε και σε κατώτερο, ας πούμε, επίπεδο. Δηλαδή, θα πρέπει να ε, δούμε και το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού εφαρμογής, επιβολής των κανόνων. Αυτή είναι η άποψή μας. Τώρα, η εκπρόσωπος των, ε, ο, ο εκπρόσωπος των Πρασίνων έχει το λόγο. Ο κύριος Μπουτικόφερ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τον εισηγητή. Πρέπει να πω ότι είναι πάρα πολύ περίπλοκο το θέμα αυτό. Και δεν έχω καταλήξει στην τελική μου τοποθέτηση σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό. αν προχωρήσουμε προ την κατεύθυνση την οποία προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι ακούσει αλλά ουσιαστικά θα τερματίσουμε οποιαδήποτε φιλοδοξία για να δώσουμε νέα πνοή στο όργανο αυτό προσφυγής. Γιατί η πραγματικότητα στη είπα σε ό,τι αφορά την τρέχουσα κυβέρνηση. Δεν υπάρχει καμία διάθεση να δοθεί τέτοια, να επιστρέφουμε στα πλαίσια του ΠΟΕ. Ούτε οι Κινέζοι, γιατί οποιαδήποτε μεταρρύθμιση θα σημαίνει α, βάρος για τους Κινέζους. Άρα το μοναδικό μεγάλο εμπορικό σκέλος που θέλει να μεταρρυθμιστεί ο ΠΟΕ από αυτήν την άποψη, είμαστε εμείς. Αν βρούμε μία λειτουργική εναλλακτική προς το όργανο πρόσφυγης, ε, δεν θα έχουμε οποιαδήποτε κίνητρο πλέον και οποιαδήποτε συμφέρον. Να κάνουμε όλες τις διαπραγματεύσεις με εταίρους που δεν έχουν καμία διάθεση να κάνουν διαπραγματεύσεις για το όργανο προσφυγής. Και θα μπει μία τελεία και παύλα στην όλη διαδικασία αυτή. Και έτσι λοιπόν θα υπάρξει ένα άλλο τμήμα ουσιαστικά στην πολυμερή, αυτή, την πολυμερή αυτή διαπραγμάτευση. Άρα ουσιαστικά και μη θελημένα θα το θάψουμε το θέμα αυτό. Και δεν είμαι σίγουρη όμω ότι αυτό είναι το σωστό συμπέρασμα και πόρισμα. Για δύο λόγου, καταρχά. δεν ε, υπάρχει κάποιος λόγος που να μας ξαναγκάζει άμεσα να εφαρμόσουμε τον νέο κανονισμό για να εξετάσουμε τα θέματα αυτά όπως ανακύπτουν. Εξ όσων γνωρίζω, θα ανακύψουν κάποιες τέτοιες υποθέσεις ε, το 2021, όχι φέτος όμως. Δεύτερο στοιχείο. Έχουμε, μία... Έχουμε σημαντικές εκλογές την 1η Τρίτη του Νοεμβρίου στη ΣΥΠΑ. Και δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση αυτή. Ενδεχομένω και να πάρουν τα πράγματα μια τροπή η οποία δεν θα μα αρέσει σε πολλού από εμά. Αλλά ενδεχομένω να υπάρξει και νέο πρόεδρο μετά τι εκλογέ αυτέ εκείνη την Τρίτη του Νοεμβρίου. Αν έχουμε δημοκρατικό πρόεδρο στον Λευκό Οίκο, εγώ δεν θα ήθελα να ξεχάσουμε οποιαδήποτε ελπίδα να συμφωνήσουμε με τους Αμερικανούς ε, για ένα σωστό αποτέλεσμα. Γιατί ξέρω από τους δημοκρατικούς Αμερικανούς ότι θα ήθελαν και θα ήταν πρόθυμοι να κάνουν μια σωστή μεταρρύθμιση για το όργανο προσφυγής. Η Τζένιφερ Χίλτον είναι μία από αυτούς και έχει μόχλευση στους δημοκράτες. Γιατί λοιπόν να προκαταλάβουμε τα αποτελέσματα αυτά ενώ μπορεί να υπάρχει κάποια ελπίδα ακόμα να συμφωνήσουμε με τους Αμερικανούς μετά τις εκλογές. Αν μας αν πιεζόμαστε αν πιεζόμασταν μάλλον να επιλύσουμε το ζήτημα γιατί είχαμε δικά μας συμφέροντα, εντάξει. Αλλά δεν φαίνεται να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Πρόεδρε, αναφέρατε ένα μεγάλο εμπορικό εταίρο, ο οποίος ενδεχομένω να δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα. Αλλά να τα πούμε τα πράγματα όπως έχουν. Ακόμα και αν υπάρχει νέος κανονισμός, δεν θα μπορούσαμε να τον επιβάλλουμε στη ΣΥΠΑ, δεν θα συμφωνούσαν και απλά θα το απέρριπταν, Θα κήρυταν πόλεμο εμπορικό, αν προσπαθούσαμε να επιβάλλουμε τέτοιο κανονισμό. Άρα, ακόμα και αν υλοποιηθούν οι φόβοι σας, ο κανονισμός αυτός δεν θα βοηθούσε σε τίποτα. Τελευταίο στοιχείο που θέλω να αναφέρω. Δεν θέλω να δώσω στον Ντόναλντ Τραμπ και στους πιστούς του τα επιχειρήματα που χρειάζονται για την προεκλογική εκστρατεία. Κοιτάξτε τι κάνουν οι Ευρωπαίοι. Προτιμούν την Κίνα και τη Ρωσία παρά να κάνουν διαπραγματεύσει με τη ΣΥΠΑ. Αυτό θα πούν. Και αυτό θα φανεί κιόλας. Όσο μιλούσαμε για τον Καναδά και την Νορβηγία, είχαμε κάποια αξιοπρεπή παρέα. Αλλά τώρα θα μπούμε σε ένα. Καζάνι. Με δύο από τις πιο δύσκολες χώρες εταίρους. Και θα ακυρώνουμε οποιαδήποτε ελπίδα να πετυχαίναμε συμφωνία με τους Αμερικανούς. Ξέρω ότι έτσι κι αλλιώς αν ξαναβγεί ο Τραμπ δεν πρόκειται να υπάρχει ελπίδα για αυτό που ελπίζω να πετύχω. Και στην περίπτωση αυτή, εντάξει, θα χρειαστεί αναγκαστικά να κάνουμε το βήμα αυτό. Αλλά μήπως θα έπρεπε αντί να προωθήσουμε αυτή την ατζέντα εδώ και τώρα να προετοιμαστούμε και να τους δείξουμε ότι είμαστε έτοιμοι να τα υλοποιήσουμε όλα αυτά όποτε χρειαστεί, χωρίς να προκαταβάλουμε όμως, ε, επαναλαμβάνω, την κατάσταση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα η ε, από το ΕΛΚ. Η κυρία Σμακοπούλου. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι πρωταθλήτρια εμπορικού συστήματο βάσει πολυμερία. Και αυτό σημαίνει να προασπιστεί τον ΠΟΕ και να προωθήσει τη μεταρρύθμιση του. Όχι μια επιφανειακή μεταρρύθμιση, μια ουσιαστική μεταρρύθμιση και ένα από τα στοιχεία τα οποία παρατηρούμε στον ΠΟΕ ότι δεν λειτουργεί αυτός ο πυλώνας για την επίλυση των διαφορών. Και καταλαβαίνω όλα όσα είπατε, όλα τα επιχειρήματα που ακούσαμε, αλλά πιστεύω ότι πραγματικά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προχωρήσει παρόλα αυτά. Θα πρέπει να προετοιμαστεί και να τοποθετηθεί. Και πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να γίνει εγκαίρος, αλλά και με εντελεχή τρόπο. Καλώς ορίζω λοιπόν το γεγονός ότι ακούσαμε ότι θα πρέπει να τοποθετηθούμε, να συζητήσουμε, να ακούσουμε όλες τις πλευρές. Δεν έχω κάτι να προσθέσω στην παρούσα φάση. Θα το εξετάσουμε το θέμα αυτό πιο εκτενώς όσο προχωράμε με το φάκελο αυτό. Ο κύριος Σόλτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και θα συμφωνούσα με κάποια από τα στοιχεία που ανέφερε ο κ. Μπουτικόφερ. Ανέφερε κάποιες προκλήσεις σε ό,τι αφορά ε, την τοποθετησή μας, σε ό,τι αφορά το πολυμερές αυτό σύστημα. Και αυτό προφανώς και συνδέεται με τις φιλοδοξίες μας ε, σε ό,τι αφορά την ε, εισφορά μας, δικό μας κομμάτι που μας αναλογεί για τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ και θα πρέπει να είμαστε φιλοδόξοι εδώ. Ε, εκ παραλλήλου, για ένα πολυμερές σύστημα εμπορικό σε παγκόσμιο επίπεδο, θα πρέπει να κοιτάξουμε τι θα γίνει και τι άλλα γεγονότα έχουμε για σήμερα. Έχουμε την ΑΚΤΑΤ 15 τον Οκτώβριο. σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη των στρατηγικών ανάπτυξη, θα πρέπει να καλυφθεί στο σκέλος αυτό και οι προκλήσεις ε, εθνικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Αν δεν γίνει λοιπόν σύνδεση ΠΟΕ και ΑΚΤΑΤ με τρόπο προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να σταθεροποιήσει την παγκόσμια οικονομία και να πετύχει αποτελέσματα για τους πολίτες, για να υπάρχει εμπιστοσύνη, δεν θα υπάρχει εμπιστοσύνη στην κατάρτιση της πολιτικής. Και αυτό νομίζω ότι θα έχει ως αποτέλεσμα τελείως διαφορετικές εξελίξεις. Εδώ λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση φέρει μεγάλη ευθύνη. Να επιδείξει λοιπόν φιλοδοξία και τόλμη. Δεν ξέρω αν καλά θα κάναμε να περιμένουμε τα αποτελέσματα των εκλογών στις ΕΠΑ. Όποιος και να βγει, οι γενικές γραμμές στο πολυμερές εμπορικό σύστημα δεν πρόκειται να αλλάξουν κατά πάσα πιθανότητα. Εμείς λοιπόν θα πρέπει να οδεύσουμε προς την σταθεροποίηση των εμπορικών κανόνων για να πλαισιώσουμε τις, Ευρωπα... τις εκλογές στην Αμερική. Hey, and now it's a turn from the Commission. It's, uh... τώρα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τον ειδικό για θέματα ΠΟΕ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχει το λόγο. Very much, Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να συμβάλλω στη συζήτησή σα σε αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων σήμερα. Θα ήθελα σε σχέση με τους προλαλήσαντες να θίξω δύο-τρία ζητήματα. Καταρχάς να καταστήσω σαφές ότι η πρόταση της Κομισιόν έχει ένα πολύ απλό στόχο, ξεκάθαρο, να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να προστατεύσει τα συμφέροντά της μπροστά σε μια ε, ε, πολύ ιδιαίτερη κατάσταση το μπλοκάρισμα των μηχανισμών επίλυσης συγκρούσεων. Έτσι, και αυτό θέλει να το κάνει με, την, ε, με το mainstreaming του εφαρμοστικού κανονισμού από το Δεκέμβριο. Είναι γεγονός, γεγονός αναμφισβήτητο, ότι Πρέπει να είμαστε σε θέση να ρυθμίζουμε καταστάσεις όπου επικρατεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια επιθετική διαμάχη σε σχέση με μια άλλη χώρα εντός του ΠΟΕ, χωρίς όμως να είναι σε θέση να αποκτήσει εντολή απαγόρευσης γιατί η άλλη χώρα προσφεύγει και παρακολύει τη διαδικασία. Δεν συμφωνεί με οποιαδήποτε ρύθμιση για την ε, επίλυση της διαφωνίας ή προσφεύγει ε, εν κενό γιατί το σώμα προσφυγών απουσιάζει και έτσι η διαδικασία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί και άρα κολλησιεργεί. Δυστυχώς σήμερα ε, ε, όποιο μέλος το επιθυμεί μπορεί να πράξει κάτι τέτοιο. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να, να δημιουργήσει κατάλληλη θεσμική αντίδραση. Και αυτό ισχύει και με τις άλλες διεθνείς εμπορικές συμφωνίες, το είπε και ο εισηγητής, όπου έχουμε καταστάσεις μπλοκαρίσματος του μηχανισμού επίλυσης διαφωνιών, το έτερο μέρος μπορεί να μπλοκάρει το διορισμό αυτών που θα αποφασίσουν και θα είναι υπεύθυνοι για την επίλυση της διαφωνίας, των adjudicators. Ένα τρίτο που θα ήθελα να σας πω είναι το εξής. Η πρόταση που έχετε μπροστά σας ευθυγραμμίζεται πλήρως με το Διεθνές Δίκαιο για τα Αντίμετρα και με τις ε, κανονιστικές διατάξεις του ΠΟΕ που είναι πολύ σημαντικές κατά τη γνώμη μας διότι βασίζονται στη πολυμερή προσέγγιση σε επίπεδο πάνελ, στο στάδιο του πάνελ. Και τέλος, αυτή η πρόταση και αυτή η προσπάθεια σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις λοιπές δράσεις και προσπάθειες για ε, μηχανισμό συλλογικής επίλυσης συγκρούσεων για να λυθεί, να λυθεί σωστά ε, το πρόβλημα αυτό με τη διαφωνία για το μηχανισμό της επίλυσης των διαφωνιών εντός του ΠΟΕ. Αυτό που προτείνουμε είναι το μέσο τελευταίας διαφυγής. Όταν το σώμα προσφυγών δεν δουλεύει και δεν λειτουργεί και όταν δεν θα έχουμε ε, μπορέσει να έχουμε θεσπίσει μια προσωρινή ε, συμφωνία για την επίλυση συγκρούσεων με το έτερο μέλος. Υπάρχει δυνατότητα να έχουμε προσωρινές μεταβατικές ρυθμίσεις με άλλες χώρες και αν αυτό καταστεί ανέφικτο, ε, να έχουμε τη δυνατότητα να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας σωστά με βάση το διεθνές δίκαιο. Δεν είναι μια πρόταση μεταρρύθμισης εκβάθρων των ε, ε, εργαλείων που έχουμε για τον κανονισμό τον εφαρμοστικό, ούτε θέλει να είναι κάτι τέτοιο και, και δεν είναι η μεταβατική και προσωρινή ε, συμφωνία την οποία συνάπτουμε ε, με διάφορες χώρες εν κίνδυνο. Δεν είναι επίσης μια μεταρρυθμιστική πρόταση εκβάθρων του ΠΟΕ. Θέλουμε να συνεχίσουμε με τη μεταρρύθμιση του μηχανισμού επίλυσης συγκρούσεων με τη συνεργασία όλων των μερών, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή η προσήλωσή μας παραμένει αταλάντευτη το έχει επαναλάβει ο Επίτροπος Χόγκαν αυτό, άρα προτείνουμε αυτόν εδώ τον εφαρμοστικό κανονισμό διότι θέλουμε να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε όλα αυτά τα εργαλεία και προτείνουμε αυτή την τροποποίηση ως μία από αυτές τις προσπάθειες στο πλαίσιο μιας ευρύτερης δουλειάς που γίνεται για να μεταρρυθμιστεί ο ΠΟΕ ε, με πιο ουσιώδη τρόπο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος και εγώ σας ευχαριστώ. Η Μαρή, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για την παρέμβασή τους, αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις διευκρινήσεις της. Όλοι οι προλαλήσαντες έδειξαν ότι στόχος είναι να στηριχθεί η πολυμερής προσέγγιση και να υπερασπιστούμε τον ΠΟΕ. Λαμβάνω υπόψη το σύνολο των παρεμβάσεων και θα προσπαθήσω να τις προσεγγίσω. Θα συνεργαστώ στενά με τους κοιόδης εισηγητές, θα καταρτήσουμε ένα πρώτο και στη συνέχεια θα γίνει μια επόμενη ανταλλαγή απόψεων στην Επιτροπή μας τον Απρίλιο, όπου και θα παρουσιάσουμε το προσχέδιο της έκθεσης. Πρέπει να προχωρήσουμε για να ακουστεί η φωνή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πολυμερές πλαίσιο. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος και εγώ σας ευχαριστώ. Η έκθεση λοιπόν θα είναι έτοιμη στις 21 Απριλίου, οπότε θα γίνει και η επόμενη ανταλλαγή απόψεων για το θέμα αυτό. Καλώς. Ολοκληρώνεται το σημείο, η εξέταση του σημείου 16 της ημερήσιας διάταξης και πριν μπούμε στο σημείο 17 θα ήθελα να καλωσορίσω μία αντιπροσωπεία από τη θαυμάσια πόλη του Γκέτεμπορκ στη Σουηδία. Μία πόλη την οποία έχω επισκεφθεί επανειλημμένως, την πόλη της Βόλβο. Καλώς ήλθατε Ερχόμαστε τώρα στο σημείο 17 της ημερησίας διάταξης. Ίσως έχει σχέση με τον Γκέτεμπορ και τη Βόλβο. Μιλούμε για την κατάσταση με το Χάλιβα και τις ασφαλιστικές δικλείδες safeguard measures με δεδομένο ότι ο, ετέ, ο εταίρος μας στην άλλη μεριά του Ατλαντικού έχει επιβάλει δασμούς στο χάλιβα και σε κάποια προϊόντα της χαλιβουργικής. Απ' την άλλη υπάρχει ε, με πολύ μεγάλη ικανότητα παραγωγή, χαλιβοπαραγωγής ε, στην Κίνα και σε άλλες χώρες και εισάγονται αυτά τα προϊόντα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε κάποιες ασφαλιστικές δικλίδες, κάποιες ρήτρες προφύλαξης για το θέμα αυτό υπήρξαν κάποιες εξελίξεις το 2019. Πιστεύω ακραδάντως ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε αυτούς τους σχετικούς κανονισμούς, διότι έχει αλλάξει δραματικά η κατάσταση το δεύτερο εξάμεινο του 2019. Στην αρχή του 2019 είχαμε κατά μέσο όρο περισσότερες εισαγωγές χάλιβα κατά 165.000 τόνους περισσότερους το μήνα ε, κάναμε εισαγωγή από ό,τι εξάγαμε. Στο δεύτερο μισό μας του 19 τριπλασιάστηκε αυτό. Μιλούμε για 1,2 εκατομμύρια ε, τόνοι χάλιβα που έμπαιναν στην ευρωπαϊκή αγορά περισσότερο από την ποσότητα που ήμασταν σε θέση να εξάγουμε. Γι' αυτό πρέπει να αναθεωρήσουμε τον κανονισμό για τις ασφαλιστικές δικλείδες, το safeguard measures, ως Ευρωπαίοι. Και πρέπει να δούμε και τι θα γίνει γενικότερα με την επιρβολική ικανότητα παραγωγής χάλιβα και χαλιβουργικών προϊόντων. Υπάρχει μια ελαφρά μείωση στην Κίνα κατά 120 δισεκατομμύρια τόνους. Παρ' όλα αυτά παραμένει το πρόβλημα του overcapacity. Επίσης, πολλή χάλιβας έρχεται από την Τουρκία μετά από τις πιέσεις των δασμών που έχουν επιβάλει οι το στο προϊόν αυτό και πρέπει και αυτό το θέμα να το δούμε. Επομένως, καλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας κάνει μια επισκόπηση των ε, θέσεων της ο Λεοπόλδο Ρουμπινάτσι είναι ο εμπειρογνώμων από πλευρά Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με πολύ μεγάλη χαρά σας δίνω το λόγο. Καλημέρα σας. Σκέφτηκα να κάνω μια σύντομη παρουσίαση για να έχετε υπόψη σας κάποια στοιχεία. Με την άδειά σας λοιπόν θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω και την προέλευση αυτών των μέτρων για να, ε, παρότι είπατε πολλά στην, ε, στην εισαγωγή σας. Θα πρέπει αυτά τα μέτρα να τα θεωρήσουμε ως τη βάση της σοβαρής κρίσης για την υπερπαραγωγή, υπερ, υπερβολική δυναμικότητα του τομέα του Χάλιβα. Ε, πολλές από, πολλοί από τους εμπορικούς μας εταίρους επέβαλαν αυστηρά μέτρα και μετά εισήχθησαν το Μάρτιο 2018 ε, μέτρα από τις ΗΠΑ με βάση το, ε, την πράξη 232 που υπέβαλε, επέβαλε φο, δασμούς 25%. Η... Υπήρξε τριπλή αντίδραση. Πρώτον ήταν η μια έρευνα διασφάλισης η οποία ξεκίνησε από την Επιτροπή Ιδία Πρωτοβουλία γιατί θεώρησε ότι υπήρξε φόβος υπερβολικής προσφοράς και ε, από τα, ότι τα αμερικανικά μέτρα κινδύνευαν να βλάψουν σοβαρά και ε, κινδύνευαν να βλάψουν σοβαρά δηλαδή η Κομισιόν κινήθηκε πριν ε, υποστεί τη βλάβη ε, ο κλάδος. Ε, κατά την άποψή μας κινηθήκαμε γρήγορα, επιβάλαμε τα μέτρα τον Ιούλιο του 2018, τα οριστικά μέτρα, την 1η Φεβρουαρίου πέρυσι, με διάρκεια τριών ετών. Επίσης, αφορούσαν όλες τις εισαγωγές εκτός από τον ΕΟΧ και την Νότια Αφρική λόγω μιας ρήτρα της εμπορικής συμφωνίας με την Νότια Αφρική και ε, αποκλείσαμε και τις αναπτυσσόμενες χώρες που εξάγουν κάτω από το επίπεδο de minimis. Ε, ε, καλύπτονται 26 κατηγορίες προϊόντων, αποτελεί τον, το ακριβό, ακρι, το ε, πεδίο ακριβώς των αμερικανικών μέτρων ε, από διάφορους σωλήνες και επίσης ε, για να συνάδουμε με τις ε, απαιτήσει εισάγαμε και ένα μέτρο αφελευθέρωσης. Επίσης, θέλαμε να προστατεύσουμε την χαλιβουργία και δεύτερον να εξασφαλιστεί επαρκής προμήθεια στην, Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν είναι αυτάρκη στον τομέα αυτό η Ένωση. Θεωρούμε ότι η κατάσταση ήταν κειμενόμενη και γι' αυτό ε, εισάγαμε μία ρήτρα ετήσιας αναθεώρησης. Έχουμε λάβαμε ε, μέτρα του τύπου των δασμολικών ποσοστώσεων και 25% εκτός ποσόστοσης για να ε, διαφυλάξουμε τις παραδοσιακές, τους παραδοσιακούς εμπορικούς δεσμούς. υπήρξαν συγκεκριμένες ποσοστώσεις ανά, χώρα, ανάλογα με, την, ε, με τα προϊόντα. Οι ποσοστώσεις μετρώνται από την ημέρα επιβολής των προσωρινών μέτρων. Δεν είναι όμως η Ιανουάριο στο Μάρτιο, αλλά είναι Ιούλιος προς Σεπτέμβριο. Η, ιδιαιτερο, οι συγκεκριμένες κατηγορία 1, 60% των εισαγωγών της Ένωσης καλύπτονται από μέτρα αντι-dumping και κατά των επιδοτήσεων και άρα θεωρήσαμε ότι οι ποσοστώσει των παραδοσιακών ε, εξαγωγέων δεν θα λειτουργούσαν και γι' αυτό ε, δημιουργήσαμε μία παγκόσμια, μία γενική ποσόστοση. Αυτά πριν επιβουληθούν τα μέτρα διασφάλισης και πραγματικά υπήρξε τεράστια αύξηση εισαγωγών ε, με κόκκινο βλέπετε το μέσο όρο της, της περίοδου 14 με 17 και ήταν τα επίπεδα των ποσοστώσεων και βλέπετε ότι αυτά είναι περίπου ίδια με τις εισαγωγές του 16 όταν εξακολουθούσε να είναι κερδοφόρα η Ευρωπαϊκή Χαλιβουργία. Ξεκινήσαμε μια πρώτη αναθεώρηση τα μέσα Μαΐου του 19, δύο μήνες μόνο μετά την θέση ενισχύ των μέτρων και είδαμε ότι τα μέτρα λειτουργούσαν σχετικά καλά αλλά ότι χρειαζόταν κάποιες προσαρμογές. Έτσι μειώσαμε το ε, ρυθμό απελευθέρωσης από το 5% στο 3%, το 30%, είχαμε 30% μέγεθος στην πρώτη κατηγορία. Η, επίσης, ε, ε, ενημερώσαμε τις, τους, τους αποκλεισμούς των αναπτυσσόμενων χωρών και επίσης το μέγιστο όριο των κατηγοριών 2 και 16 για να αντισταθμιστεί το crowding out και οι προσαρμογές ε, ε, τέθηκαν ενισχύ την 1η Οκτωβρίου του 2019. Τώρα, αυτά θα σας τα εξηγήσω λίγο καλύτερα. Αν βλέπετε καλά, θα δείτε ότι ε, ε, ε, ποια είναι η κατάσταση με τις διάφορες χώρες. Η, Τουρκία πήρε το μερίδιο του λέοντος και γι' αυτό βάλαμε ένα μέγιστο όριο ώστε καμία χώρα να μην μπορεί να εξάγει πάνω από το 30% της συνολικής διαθέσιμης ποσόστοσης. αυτό είναι το λεγόμενο crowding out. Αριστερά βλέπετε τι γίνεται στο τρίτο ε, τρίμηνο όταν οι χώρες εξάγουν με βάση τις ε, ειδικέ ποσοστό σε ένα χώρα και βλέπετε μετά τους παραδοσιακούς ε, προμηθευτές όπως η Λευκορωσία η οποία μπορεί να εξάγει στην Ένωση. Ενώ δεξιά βλέπετε <clears throat> τι συνέβη το τέταρτο τρίμηνο όταν χώρες που είχαν εξαντλήσει τις ε, ε, ποσοστώσεις της χώρας τους μπορούσαν να εκμεταλλευτούν την υπολοιματική ποσόστοση. Και βλέπετε εδώ εισαγωγές από την Τουρκία οι οποίες ε, αφαιρούν όλες τις δυνατότητες εξαγωγών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση από άλλους παραδοσιακούς προμηθευτές μας. Έτσι λοιπόν λειτουργούν τα μέτρα διασφάλισης. Αν συγκρίνεται την ε, εφαρμογή του 19 σε αιτήσια βάση σε σχέση με την κορύφωση των εισαγωγών του 18 έχουμε μία μείωση ε, πάνω από 4 εκατομμύρια τόνους και επιστρέφουμε στα 28-29 εκατομμύρια τόνους που θεωρούμε ότι δεν είναι επιβλαβές επίπεδο. Αυτό δείχνει ότι οι διασφαλίσεις πέτυχαν το στόχο τους, δηλαδή ε, μας προστάτευσαν από, την ε, μεγάλη ε, εισαγω... από τις μεγάλες εισαγωγές. Εδώ βλέπετε την εξέλιξη των εισαγωγών. Το κίτρινο σημειώνει τις εισαγωγές του 19 πάντοτε είναι χαμηλότερα από τα επίπεδα του 18 και σε περισσότερες περιπτώσεις χαμηλότερα και από τα επίπεδα του 17. Και κατόπιν, πέραν της ε, του περιορισμού του συνόλου των εισαγωγών βλέπουμε ότι είδαμε ότι υπάρχουν και πάνω από 3 εκατομμύρια τόνοι των, από τις ποσοστώσεις που δεν χρησιμοποιήθηκαν, δηλαδή δεν υπήρξε ε, στε, ε, έλλειψη στην προμήθεια. Ε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ε, ξεκινήσαμε την δεύτερη αναθεώρηση την περασμένη Παρασκευή σκοπός εδώ δεν είναι να αμφισβητηθούν οι διασφαλίσεις, αλλά εάν υπάρχει ε, πεδίο περαιτέρω βελτίωσης. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα. Ε, η, η, η ανακοίνωση έναρξης της ε, διασφάλισης περιλαμβάνει δεσμεύσεις, οπωσδήποτε δε πριν τις 30 Ιουνίου, ε, για την ολοκλήρωση. Βεβαίω, αν λάβετε υπόψη σα. πόσο χρόνο χρειάζεται για όλε αυτές τις διαδικασίες, στην ουσία δύο εβδομάδες μένουν για έρευνα. Στο σημείο αυτό θα ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε, αλλά με, τα χαρά να απαντήσω σε ερωτήσεις. Um, Ευχαριστώ πολύ, ο Σούστερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μία ερώτηση έχω να κάνω η οποία όμως είναι σημαντική για την εξέλιξη που παρατηρούμε στην χαλιβό βιομηχανία. Πώς υπολογίζετε τι γίνεται στον ε, χαλιβουργικό ε, τομέα μέσα στην κρίση. Μειώνεται δηλαδή η παραγωγή, αλλά αυξάνονται οι εξαγωγές και η παραγωγή. Αυτό θεωρώ ότι σημαίνει περισσότερη πίεση. Και γι' αυτό λοιπόν τά τά συνυπολογίζουμε τα συνυπολογίζουμε ή κάνουμε λες και είναι ίδια ε, η παραγωγή χάλβα στην Ευρώπη. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να υπολογίσουμε, να δούμε πώς υπολογίζονται όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σκάνας. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είδαμε σημαντική αλλαγή στις συνθήκες και στις περιστάσεις από την τελευταία αναθεώρηση των μέτρων το καλοκαίρι του 2019. Το 2019 η παραγωγική ικανότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μειώθηκε σε σχέση με το 2018, ειδικότερα στην αυτοκινητοβιομηχανία, όπου είχαμε πτώσει τις τάξεις του 7%. Αυτό σημαίνει ότι η ζήτηση στην Ευρώπη είναι πιο ασθενής Έχουμε πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, έχουμε ύφεση στην τουρκική οικονομία και γι' αυτό έχουμε περισσότερες εισαγωγές, δυσανάλογα περισσότερες, παρότι υπάρχει πτώση της ζήτησης. Και αυτό οδήγησε σε περικοπές παραγωγής ε, ύψους 3,4 εκατομμυρίων τόνων από πλευράς παραγωγών. Διατηρούμε πολύ ψηλά επίπεδα εισαγωγών οι ποσοστώσει εισαγωγών ε, χρησιμοποιήθηκαν στο δεύτερο εξάμεινο του 19 παρά την πτώση της ζήτησης. Έχουμε τις ανάλογα υψηλές ποσοστώσεις. Η Επιτροπή θα εξετάσει το ενδεχόμενο να διαγράψει την αυτόματη μεταφορά των ποσοστώσεων, τον αυτόματο μηχανισμό επιβολής ποσοστώσεων από τη στιγμή που η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική. Είχαμε ποσόστοση 5% όταν είχαμε τα τελικά μέτρα το Φεβρουάριο, ε, γιατί περιμέναμε αύξηση. Δεν έγινε αυτή η αύξηση. Θα το διαγράψει η Κομισιόν αυτό το 5%, θα προσαρμόσει τις ποσοστώσεις στην πραγματική ζήτηση της αγοράς. Ευχαριστώ. Και εγώ το ίδιο ερώτημα ήθελα να θέσω δεν θέλω τίποτα άλλο να προσθέσω, λέει ο κύριος Μορέλ. Um, Κύριε Σασίνη. Σαλίνη. Διορθώνει ο βουλευτής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κι εγώ συμφωνώ με τα σχόλια του κυρίου Κάνια πολύ εύστοχα. Θέλω να προσθέσω όμως και κάτι, γιατί έχω λίγο μπερδευτεί. Για να μπορέσουμε να δούμε τα αποτελέσματα των διασφαλίσεων, θα πρέπει να δούμε όχι το, τον υπολογι... να μην υπολογίζουμε τη διαφορά σε τόνους, αλλά το μερίδιο της αγοράς. Αυτό ίσως αποτελεί καλύτερο δείκτη και ενδεχομένως αυτό να είναι ενδιαφέρον κριτήριο. Υπόθηκε ότι δεν θα γίνει αποδεκτό από τον ΠΟΕ. Νομίζω όμως ότι δεν ισχύει αυτό. Παρά τα αυτά, εξακολουθεί να ισχύει το εξής. Πώς θα περιοριστούν οι ζημιές με τη χρήση των διασφαλίσεων οι προσπάθειες να αντιμετωπιστεί αυτό έχουν αποτύχει μέχρι τώρα. Και συμφωνώ με τις ανησυχίες που έχουν διατυπωθεί. Δεν μπορούν όλα να μεταφερθούν. όλοι όχι όλη η ποσόστοση που δεν έχει χρησιμοποιηθεί δεν μπορεί να μεταφερθεί. Πρέπει να δούμε μια συνολική μείωση της ποσόστοσης που χορηγείται στις μεγάλες χώρες, ας πούμε την Τουρκία. Θα πρέπει να περιορίσουμε την χρήση της υπολοιματικής ποσόστοσης, αλλά να εξετάσουμε και τις ε, εθνικές ποσοστώσεις που χορηγήθηκαν είναι ο μόνος τρόπος, θεωρώ, που θα μπορέσουμε να, έχουμε, να αντιμετωπίσουμε την αγορά η οποία βρίσκεται σε κρίση. Η ευρωπαϊκή αγορά είναι σε κρίση και ο κίνδυνος είναι να χάσουμε ένα πολύ μεγάλο ε, κομμάτι της ε, εφοδιαστικής ε, αλυσίδας αξίας και ο χρόνος πιέζει. Υπάρχει εν γέννη υποστήριξη ακούγοντας, ε, μπορώ να πω ακούγοντας τους προηγούμενους ομιλητές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σόλτς. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις εξηγήσεις που μας έδωσε. Νομίζω ότι χρειάζεται σημαντικές αλλαγές ε, σε ό,τι αφορά ασφαλιστικά μέτρα. Αυτό δεν χωράει εμφιβολία. Το θέμα είναι πώς θα το πετύχουμε, τι θα κάνουμε. Αυτό ενδεχομένως να μην το έχουμε εξετάσει επαρκώς στη συζήτηση ως τώρα. Έχουμε καταρχάς ε, τη μεταφορά ποσοστώσεων. Ε, είναι ένα εργαλείο που έχει σημαντικό κίνδυνο. Γιατί όταν αλλάζουν οι οικονομικές καταστάσεις, προφανώς βρισκόμαστε σε μια κατάσταση χωρίς προστασία για την ε, ευρωπαϊκή χαλιβουργία. Γιατί θα ήταν Άδικέ οι ε, ποσοστώσει. Άρα να σκεφτούμε το ανώτατο όριο και πάλι. Τα οριζόμενα ανώτατα όρια δεν είναι τα κατάλληλα. Και η δεύτερη μεταρρύθμιση των ε, δεσφαλιστικών μέτρων θα πρέπει να επικεντρωθεί στο 30% σε ό,τι αφορά τα ποσοστό για τις ε, χώρες εξαγωγών. Ενδεχομένω λοιπόν και να μπορέσουμε να ξανακοιτάξουμε το μηχανισμό στο σύνολό του. σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, τις ε, διαρκείς ε, αλλαγές ε, που υπάρχουν στις αγορές εξαγωγών, θα πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτό, να μην έχουμε μια εφάπαξ λύση, να υπάρχει ένας ρευστός μηχανισμός. Ένα δεύτερο σημείο το οποίο δεν άκουσα επίσης είναι το θέμα της διαρροής άνθρακα. Αυτός ο κίνδυνος. Λοιπόν, ρωτιέμαι, η όλη αλλαγή της ε, γερμανικής ή της ευρωπαϊκής χαλιβουργίας σε ό,τι αφορά το διοξείδιο του άνθρακα, πώς θα ε, επιδράσει αυτή η προσαρμογή στα σύνορα. Αναρωτιέμαι. Θα ληφθεί υπόψη σε ό,τι αφορά το διοξείδιο του άνθρακα. Αυτό θα ληφθεί υπόψη και στον μηχανισμό για τις ποσοστώσεις. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε κίνητρα προκειμένου να γίνει αυτή η αλλαγή που χρειάζεται στο διεθνές προσκήνιο και στο αλουμίνιο φαντάζομαι, όχι μόνο στο χάλβα. Θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα έσοδα από την διασυνοριακή προσαρμογή και να χρησιμοποιηθούν αυτά τα χρήματα για την μεταρρύθμιση που χρειάζεται. Για να υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού, οι οποίοι δεν υπάρχουν στην παρούσα φάση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σμπιτικόφερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και το δεν είμαι εμπειρογνώμονα στα θέματα χάλιβα, γι' αυτό θέλω να τα κοιτάξουμε σε πιο απλό επίπεδο τα πράγματα το κατά πόσον χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Χαλιβουργία μία επιπρόσθετη προστασία. Θεωρώ ότι το, η απάντηση είναι θετική και μόνο. Χρειάζεται. Θα πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε τις προτάσεις της Eurofair. Και θα συμφωνούσαμε με αυτά που είπε ο κ. Σόλτς σε ό,τι αφορά το όριο του 30%. Κατά δεύτερον, να παρακαλέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πιο προσεκτικά πώς αυτή η μεταρρύθμιση και μεταμόρφωση της χαλιβουργίας μπορεί να κινηθεί προς την κατεύθυνση του πράσινου χάλιβα, αν μου επιτρέπετε να το πω έτσι. Πώς, λοιπόν, αυτή η μεταμόρφωση θα ληφθεί υπόψη στα μέτρα τα οποία θα λάβουμε. Άκουσα προσεκτικά αυτά που μας είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά αυτό δεν ε, επισημάνθηκε. Είναι όμως αφές, ευθύς εξ αρχής, ότι θα μπορούσαμε να εντάξουμε και το σκέλος αυτό. Θα πρέπει να το κοιτάξουμε λοιπόν πιο προσεκτικά. Γιατί, ωραία, δεν ε, μπορούμε να αναβάλουμε αυτή την ε, μεταμόρφωση, αν θέλετε, της αγοράς μέχρι ότου βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση. Ο Πρόεδρος, κοιτάξτε, είναι σοβαρά τα θέματα. Και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια υπήρξε μία μείωση στην παραγωγή χάλιβα 8 ε, δις τόνους στην Ευρώπη. 15.000 θέσεις. Αυτό προφανώς θα πρέπει να υπόψη και στην όλη φάση, στην όλη διαδικασία μεταρρύθμισης του κλάδου. Ε, το ακούσατε ερωτήσει των συναδέλφων και ίσω θα μπορούσατε να κάνετε και κάποια σχόλια για τη γενικότερη παγκόσμια κατάσταση στον κλάδο αυτό. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ και σα ευχαριστώ για τα σχόλια που κάνατε. Ευχαριστώ. Θα απαντήσω κατευθείαν. Θα απαντήσω κατευθείαν στην ερώτησή σας. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι η κατάσταση με την υπερπαραγωγή ε, στο χάλβα είναι κακή εξακολουθεί να υπάρχει εκτεταμένη υπερπροσφορά στον τομέα και υπάρχουν ε, εμπορικοί εταίροι που συνεχίζουν να ασκούν πρακτικές που στρεβλώνουν την αγορά, κυρίως μέσω επιδοτήσεων. Άρα εμείς είμαστε δεσμευμένοι να βελτιώσουμε τους κανόνες για, την, ε, για τις επιδοτήσεις, επιμένουμε, εξετάζουμε τα στοιχεία αυτά πολύ προσεκτικά. Πιθανότητα αυτό είναι ο λόγος, το γεγονός ότι παραμένει μια εξαιρετικά στρεβλή κατάσταση στο διεθνές εμπόριο. Αυτός είναι ο λόγος που ε, η Ευρωπαϊκή Χαλιβουργία είναι αυτή που είναι περισσότερο προστατευόμενη από τα εμπορικά μέτρα η Ευρωπαϊκή Χαλικουργία προστατεύεται από περίπου 25 μέτρα κατά του ντάμπινγκ και των επιδοτήσεων. Έχει καταγράψει η Επιτροπή, ε, αντιδρά, έχουν καταγραφεί ε, ε, κάθε φορά αντιδράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όταν, υπάρχουν, όταν υπάρχει και ντάμπινγκ και επιδοτήσεις. Γίνονται αυτή τη στιγμή διάφορες έρευνες Είμαι βέβαιος ότι οποτεδήποτε η Ευρωπαϊκή Χαλιβουργία διαπιστώνει επιζήμια πρακτική, δεν θα διστάσει να ε, υποβάλει ε, προσφυγές. Ξεκίνησαν λοιπόν οι ευρωπαϊκές διασφαλίσεις, έχουμε σημειώσει με προσοχή τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις των μελών Θέλω όμως να είμαι σαφής σχετικά με το τι είναι εφικτό και τι δεν είναι. Οι διασφαλίσεις δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ε, επιτύχουν μείωση της εσωτερικής ζήτησης. Μόνο για να ε, αντιμετωπίσουν την ευνίδια αύξηση των εισαγωγών που είναι επιβλαβής. Αλλιώς πρέπει να χρησιμοποιηθούν άλλα μέτρα. Το ίδιο ισχύει και για την διαρροή άνθρακα carbon leakage. Αυτό που μπορούν να κάνουν όμως είναι να να φροντίσουν, να εξασφαλίσουν ότι το επίπεδο εισαγωγών δεν θα ξεπερνά ένα επίπεδο πέρα από το οποίο θα προκληθεί ζημιά. Άρα η ποσοστός, η σημείωση του 30%, οι δυνατότητες ε, των εξαγωγών να εκμεταλλευτούν ε, την πολυματική ποσόσταση. Όλα αυτά είναι εφικτά στο πλαίσιο της αναθεώρησης και είμαι βέβαιος ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη θα ε, μας ε, απασχολήσουμε αυτά τα θέματα. Αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε είναι να μειώσουμε ε, τα επίπεδα ποσόστοσης ε, κάτω από το ε, ιστορικό εμπόριο της περίοδου 15-18. Επίσης δεν μπορούμε να έχουμε οποιοδήποτε στοιχείο προοδευτικής απελευθέρωσης. Αυτά δεν είναι επιτρεπτά. Πέραν αυτού όμως πολλά μπορούν να γίνουν και έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε ότι οι διασφαλίσεις θα λειτουργήσουν καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, παρακαλώ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι οι απαντήσεις που μας δόθηκαν σήμερα ήταν ξεκάθαρες. Και φαίνεται ότι εμείς είμαστε οι μόνοι στους οποίους μπορεί κανείς να έχει εμπιστοσύνη. Ότι δηλαδή είμαστε οι μόνοι που τηρούμε τους κανόνες του ΠΟΕ. Οι μόνοι είμαστε που φαίνεται να τους τηρούμε και κανείς άλλος. Όταν μιλούμε όμως για το μέλλον της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, πρέπει κανείς να δει τα θετικά του ΠΟΕ. Αν είναι τώρα να λέμε τι καλό για την Ευρωπαϊκή Βιομηχανία είναι να είναι μέλο του ΠΟΕ, ε, ας το κάνουν αυτό οι οικονομολόγοι οι πανεπιστημιακοί, να γράφουν ε, μελέτες και ούτω σε θεωρητικό επίπεδο. Θα πρέπει όμως στην πράξη να δούμε την αλήθεια κατάματα και αυτό είναι πιο σημαντικό. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος κ. Κάνιας. Συμφωνώ με τον συνάδελφο. Οι απαντήσει είναι επίσημε. Αλλά μόνο εμεί οι Ευρωπαίοι τηρούμε του κανόνε. Κανεί άλλο δεν του τηρεί. Πηγαίνετε εσεί να εξηγήσετε σε 15.000 ανθρώπου που έχουν χάσει τη δουλειά του ότι τα κάναμε όλα σωστά και παίζουμε με του κανόνε. Τι θα του πούμε δηλαδή. Δηλαδή θα πάμε στου 15.000 ανθρώπου που έχουν χάσει τη δουλειά του να του πούμε ότι εμεί τηρούμε του κανόνε και άλλοι όχι και τι να κάνουμε. Ξέρουμε ποιε χώρε εφαρμόζουν όλα αυτά. Ξέρουμε τι σημαίνουν όλα αυτά για τις χώρες μας για τους παραγωγούς μας και για τους εργαζομένους μας. Δεν είναι τίποτα καινούριο αυτό, δεν είναι κενό υπό το φως του ηλίου. Είχαμε κάνει και παρεμφερή συζήτηση, να υπάρχει level playing field. Αυτό είναι, είναι λέξη της μόδας, ένα αυτές οι νέες λέξεις που πρέπει όλοι να ε, υιοθετούμε στο λεξιλόγιο μας. Όχι, πρέπει να έχουμε ίσους κανόνες για όλους, για να μην μετακινούνται τα τέρματα να είναι ίσοι οι κανόνες για όλους και ισορροπημένοι. Αυτό πρέπει να απαιτήσουμε. Ιδαλλιώ χάνουμε θέσει απασχόληση, χάνουμε βιομηχανία, χάνουμε παραγωγική δραστηριότητα, γιατί έχουμε ανταγωνιστέ οι οποίοι μα βάζουν συνεχώ παγίδε και οι οποίοι στρεβλώνουν την αγορά. Και δεν είναι μόνο αριθμητικά στοιχεία, γραφικέ παραστάσει, ε, τυράκια, καμπύλε. Αριθμητικά στοιχεία είναι άνθρωποι, αληθινοί άνθρωποι που χάνουν τη δουλειά του. Ναι, ναι, να έχουμε ισότιμους κανόνες, αλλά για όλους. Και όταν υπάρχουν παίκτες οι οποίοι δεν τηρούν τους κανόνες και μάλιστα συστηματικά, το να πηγαίνει κανείς με το σταυρό στο χέρι και να λέει ότι εμείς θα κάνουμε όλα σωστά, ε, δεν φτάνει. Πρέπει να το εξηγήσετε αυτό και να το πείτε πιο ξεκάθαρα. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ, κύριο Σούστερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω κι εγώ μια μικρή παρατήρηση με τη σειρά μου. Δεν είναι πολύ αποτελεσματικό να μην βασίζεται κανείς στη ζήτηση, διότι δεν θα εκπληρώσει το στόχο της δημιουργίας των ε, βέλτιστων συνθήκων ανταγωνισμού, των ευίωνων συνθήκων ανταγωνισμού. Δεν προστατεύει έτσι τη βιομηχανία, και θα υπάρξει μεγάλη αναταραχή στους κόλπους των βιομηχανικών και παραγωγικών κλάδων. Και αυτό είναι πολύ προβληματικό, διότι η Ευρώπη είναι σημαντική είναι πολύ οι κρίκοι της αλυσίδας που επηρεάζονται ο ένας από τον άλλον και αν δεν μπορούμε να εφοδιαστούμε και να προμηθεύουμε τους εαυτούς μας με τα αγαθά που μας χρειάζονται, όντως πρέπει να κάνουμε εισαγωγές, αλλά όχι εισαγωγές ε, άκρητα χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τη ζήτηση. Επιμένω λοιπόν να λαμβάνεται υπόψη η ζήτηση και να υπάρχει ε, ισορροπημένη προσέγγιση. Ο κύριος Σόλτς παρακαλώ. Και εγώ έχω να κάνω ένα σχόλιο ε, σε σχέση με τις προηγούμενες παρατηρήσεις, οι οποίες ήταν πολύ σαφείς και θέλησαν να εκπέμψουν ένα στοιχειώδες μήνυμα, α, σαφέστατο. Δεν πρόκειται περί ε, προστασίας απλά των θέσεων απασχόλησης στην ευρωπαϊκή παραγωγική αλυσίδα. Δεν μιλούμε μόνο γι' αυτό. Είναι παγκόσμια η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε. Πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα της ζήτησης και της προσφοράς. Πώς θα καταλήξουμε σε ένα σημείο ισορροπίας. Γι' αυτό επιστρέφω σε αυτό το θέμα του φόρουμ του Χάλιβα. Εάν το φόρουμ του Χάλιβα δεν λειτουργεί πλέον, γιατί είναι αποκλίνουσες οι απόψεις των μεν και των δε ορισμένων, ε τότε θα πρέπει να μεταρρυθμιστεί δομικά, διαρθρωτικά το φόρουμ αυτό. Και περιμένω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Διπουργική Διάσκεψη να είναι σε θέση να καταθέσει πρόταση επιτάπητος, ώστε το φόρουμ της Χαλιβουργίας στο πλαίσιο του ΠΟΕ να αναδιοργανωθεί καλύτερα. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μια σύντομη παρατήρηση ε, προς τον ε, εκπρόσωπο της Κομισιόν τώρα που προσέχετε, ε, αν προσέξατε, η συζήτηση ξεκίνησε ε, την στιγμή που έπρεπε να έχει τελειώσει. Πριν από λίγα χρόνια η, απάντησή σας ήταν τέλεια, μια ωραία παρουσίαση και θα είχαμε... Ε, εγώ είμαι Ρουμάνος και έχουμε πληρώσει το τίμημα της προς, ε, τη ένταξής μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλους τομείς και στη χαλιβουργία μας. Έτσι λοιπόν, αφού οι συνέπειες είναι και κοινωνικές, αφού η ευθύνη είναι πολιτική ευθύνη, πιστεύω ότι έφτασε η στιγμή της αλλαγής και δεν υπάρχει θέμα Green Deal ή τήρηση των κανόνων του ΠΟΕ που φαίνεται ότι είμαστε οι μόνοι που ε, τηρούμε, δεδομένου ότι και αυτό θα φανεί στην συζήτηση που θα ακολουθήσει, νομίζω ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά από μια καινούρια ε, σκοπιά. Έχει ζητήσει το λόγο ο, ε, ε, ο προσκεκλημένος από τον ΠΟΕ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λυπάμαι έφτασα με καθυστέρηση, ενδεχομένως ε, τα λόγια μου να μην είναι απολύτως σχετικά, αλλά επ' αυτού. Θεωρώ ότι όταν οι χώρες δεν τηρούν τους κανόνες του ΠΟΕ, τότε ε, έχουμε πρόβλημα δραστηριότητας. Έχουμε καταδίκες στο παρελθόν Εν τω μεταξύ όμως οι αποφάσεις ε, φτάνουν χρόνια αργότερα. Εν τω μεταξύ όμως μπορούν να ληφθούν συντηρητικά ασφαλιστικά μέτρα, ώστε για να, ε, γίνουν πιο σωστές αυτού του είδους οι συναλλαγές. Στην περίπτωση του αλουμινίου ας πούμε υπήρξαν χώρες που κάνουν ε, μεταφορά ε, παραγωγής σε, άλλες, σε σχέση με άλλες χώρες τις οποίες στόγευαν τα μέτρα. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο, με αυτά τα ασφαλιστικά μέτρα μπορούμε να, φέρουμε, να κάνουμε ορθότερο το διεθνές εμπόριο. Ε, ευχαριστώ. Τι να πω, λέει ο πρόσωπος της Κομισιόν. Θέλω να είμαι σαφής σχετικά με δύο ζητήματα. Πρώτον, ακούσαμε αυτά που υπόθηκαν. Και δεύτερον, είπα ότι τα περισσότερα πόσα έθεσαν τα μέλη σχετικά με την πιθανή βελτίωση των διασφαλίσεων είναι εφικτά. Απλώς πρέπει να κάνουμε έρευνα. Ταυτόχρονα, ο κύριος Σούστερ έχει απόλυτο δίκιο. Υφίσταται σχέση μεταξύ ε, ανάμεσα στο τι γίνεται στην εσωτερική αγορά και στις εισαγωγές. Άρα η απάντηση πρέπει να είναι πολύπλευρη. Δεν μπορούμε τα πάντα να τα βάλουμε σε σχέση με τις διασφαλίσεις. Πρέπει να υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Γιατί οι διασφαλίσεις εκφύσεως είναι προσωρινό εργαλείο. Εργαλείο που μόνο με το επίπεδο των εισαγωγών μπορεί να ασχοληθεί. Υπάρχουν και πολλά άλλα με τα οποία πρέπει να ασχοληθούμε. Ας πούμε, η Κομισιόν προσπαθεί να εκπονήσει βιομηχανική στρατηγική. Δεν είχα λοιπόν καθόλου σκοπό να απαντήσω τυπικά και επίσημα. Ήθελα να είμαι όσο το δυνατόν σαφέστερος σχετικά με το τι είναι εφικτό στο πλαίσιο των διασφαλίσεων και αυτά τα οποία δεν είναι εφικτά στο πλαίσιο των διασφαλίσεων θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με άλλα μέτρα και δεν είπα ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλλα μέτρα. Ευχαριστώ. Οπότε, λέει ο πρόεδρος, θα εξετάσουμε τις 15 ημέρες της αναθεώρησης των ε, διασφαλίσεων και είμαστε πεπισμένοι ότι θα συνεχιστεί η συζήτηση για να στηρίξει η Ευρωπαϊκή Χαλιβουργία σε σχέση με τα αιτήματα, την ψηφιοποίηση και την μετατροπή ε, της παραγωγής χάλιβα χωρίς ε, διοξίδιο του άνθρακα. Γιατί θέλουμε η Ευρώπη να, είναι βασικό, να έχει βασικό στοιχείο το χάλιβα στην αλυσίδα αξίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τα μέλη και τους συμμετέχοντες και τώρα περνάμε στο σημείο 18. um, Οπότε φτάσαμε σε μια σειρά θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που αφορούν τον ΠΟΕ. Παρατάφτα και σε δύο από τα προηγούμενα θέματα που συζητήσαμε έπαιξε σημαντικό ρόλο ο ΠΟΕ. Εξακολουθεί λοιπόν να είναι ο ΠΟΕ ένα θέμα που ε, αφορά πολλά από τα ζητήματα που απασχολούν την ε, Επιτροπή μας. Και πρέπει να επιμείνουμε στο σύστημα εμπορίου με βάση τους κανόνες, παρότι μερικές φορές δεν είναι και τόσο εύκολο. Θέλουμε όμως να βελτιώσουμε τις δυνατότητες του ΠΟΕ. Λόγω της συνάντησης της δικού σας επιτροπής, στις ε, κοινοβουλευτικής ε, συνάντησης που γίνεται σήμερα στις Βρυξέλλες, εμείς εδώ στην Επιτροπή επικεντρωνόμαστε στον ΠΟΕ. Και ε, καλωσορίζω τα μέλη της ε, δικού σας επιτροπής, της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του ΠΟΕ. Πολλοί από αυτούς παρίστανται στη συνεδρίασή μας. Σας καλωσορίζω θερμότατα. Έχετε έρθει από την Βραζιλία, Ινδία, Καζακστάν, Σενεγάλη και πολλές άλλες χώρες. Καλώς ορίσατε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ίντα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Από το 2002, μαζί με την Διεθνή Κοινοβουλευτική Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχουμε αναλάβει την Διοικούσα Επιτροπή της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΠΟΕ, η οποία συνεδριάζει τακτικά. την προκειμένη συνάντηση στο πλαίσιο της προετοιμασίας της ε, υπουργικής συνάντησης που θα γίνει στο Νουρ Σουλτάν φέτος τον Ιούνιο. Είναι πολύ καλή αυτή η παράδοση ε, για που επιβάλλει δύο συμπροέδρους. Ο συμπρόεδρός μου βρίσκεται εδώ, δίπλα μου, είναι ο δόκτωρ Φαλίτ Τσόν, μέλος του Κοινοβουλίου της Ινδονησίας. Θα του δώσω το λόγο για να ε, μιλήσει στα μέλη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λάγκα. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ εκ μέρους ε, του Προέδρου της Διακοινοβουλευτικής ε, Ένωσης. Το θέμα που θα συζητηθεί είναι πολύ σημαντικό. Η προετοιμασία για το Καζακστάν, την Υπουργική του Καζακστάν και την ε, διακοινοβουλευτική διάσκεψη του ΠΟΕ, καθώς πλησιάζουμε την ημερομηνία δεξιαγωγής της η αντιπροσωπεία της δικού σας επιτροπής θα συζητήσει την ουσία και την προετοιμασία του ΠΟΕ. Σήμερα το απόγευμα ενδεχομένω. Είμαστε ευγνώμονες που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φιλοξενεί τη συνάντηση Νομίζω ότι το θέμα αυτό θα συζητηθεί ε, μετά την μεσημεριανή διακοπή. Ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ζών ε, για την παρουσία σας εδώ και για την ομιλία σας. Βεβαίως, η συνεδρίαση της Διοικού σας Επιτροπής θα ξεκινήσει το απόγευμα. Ένα θέμα της διάσκεψης που θα γίνει στο Νουρ Σουλτάν είναι το θέμα της μεταρρύθμισης του ΠΟΕ που έχει επίσης συζητηθεί και από τα κράτη-μέλη του ΠΟΕ. Χαίρομαι ιδιαίτερα λοιπόν που έχουμε τον, τον ε, πρέσβη του Καναδά, τον Στέφεν Ντεμπόρ, ο οποίος θα μας μιλήσει. Δεδομένου ότι ο Καναδάς είναι, ανήκει στην λεγόμενη ομάδα της ΟΤΑΒΑ, η Όταβα Group του ΠΟΕ, η οποία προσπαθεί να επιτύχει την μεταρρύθμιση του ΠΟΕ. Η ομάδα της Οτάβας, λοιπόν, στην οποία συμμετέχουν μέλη του ΠΟΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες, έχουν συνεδριάσει τρεις φορές σε μια μικρουπουργική βάση τελευταία φορά συναντήθηκαν στο Νταβός. Βεβαίως, πέρα το γενικό ζήτημα της μεταρρύθμισης του ΠΟΕ, υπάρχει και το θέμα της μεταρρύθμισης του μηχανισμού επίλυσης διαφορών και του οργάνου προσφυγών, όπως επίσης και θέματα της εξέλιξης της ε, ατζέντας ατζέντα όπως τους κανόνες Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκεται εδώ ο κύριος Ντεμπόρ. Έχετε το λόγο. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία να ενημερώσω την Επιτροπή σας για τις απόψεις και τις προτεραιότητες του Καναδά για τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ. Ελπίζω να έχουμε μια καλή συζήτηση μετά. Θα ήθελα να ξεκινήσω αναφέροντας κάτι το βασικό. Παρότι μπορεί να έχετε ακούσει κάτι διαφορετικό, ο ΠΟΕ δεν βρίσκεται καθόλου στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Γίνονται διαπραγματεύσεις, οι επιτροπές συνεδριάζουν, τα ζητήματα συζητώνται, οι ιδέες προωθούνται, προχωρούν και ακόμα και οι διαφωνίες προβάλλονται για να επιληθούν. Ναι, πράγματι υπάρχουν σοβαρές προκλήσεις και θα έρθω σε αυτές εντός ολίγου. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε όμως ότι αυτός ο οργανισμός συνεχίζει να λειτουργεί και να προσθέτει αξία στη δουλειά μας. Πρέπει να να καταρρύψω το μύθο ότι έχουν αποχωρήσει οι από τον ΠΟΕ. Πράγματι, οι έχουν ε, υιοθετήσει μια διαφορετική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των ζητημάτων εντός του ΠΟΕ και παρόλο που η προσέγγιση τους είναι διαφορετική με τον τρόπο με τον οποίο παραδοσιακά οι ΗΠΑ ε, δούλευαν και λειτουργούσαν εντός του ΠΟΕ, παραμένουν οι ΗΠΑ Πολιτείες εξαιρετικά δραστήριες στο έργο του οργανισμού αυτού. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η φυστάμενη κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο ΠΟΕ δεν είναι ε, λόγω λάθους ή δράσεων ενός μέλους Όλοι έχουμε ευθύνε γι' αυτό. Επομένως, είναι λογική η παραδοχή ότι ο μόνος τρόπος να επέλθουν αληθινές αλλαγές στον ΠΟΕ είναι μέσα από τη συλλογική δράση, εξού και η πρόκληση. Νομίζω ότι με ασφάλεια μπορούμε να πούμε ότι είναι ομόφωνη συμφωνία βάσει της οποίας ο ΠΟΕ πρέπει να μεταρρυθμιστεί για να διασφαλίσει ότι θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του με έναν τρόπο που να ταιριάζει στις ανάγκες και στις προκλήσεις του 21ου αιώνα. Όμως η συλλογική συμφωνία και αυτά που πρέπει να επιληθούν και το πώς θα γίνουν όλα αυτά για να πετύχουν πετύχουμε τους στόχους μας είναι κάτι που μας διαφεύγει. Το διακύβευμα, η επίλυση των διαφωνιών, οι βιομηχανικές ενισχύσεις, η αντιμετώπιση των αναπτυσσόμενων χωρών μεταξύ άλλων. Όλα αυτά είναι περίπλοκα ζητήματα. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να προχωρήσουμε προς τα εμπρό σε σχέση με αυτά τα ζητήματα. Αυτό απαιτεί χρόνο. Είναι δύσκολο. Και η πρόοδος θα, θα υπάρξει με αθρηστικό, με σορευτικό τρόπο, σιγά σιγά, λίγο λίγο. Αυτό δεν σημαίνει ότι καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια και περιμένουμε να συμβούν τα πράγματα από μόνα τους. Το Σώμα Προσφυγών ένα καλό παράδειγμα. Ο Καναδάς είναι δεσμευμένος να συνεργαστεί με όλους για βιώσιμη λύση. Δεν θα καθίσει με οκνηρό τρόπο να παρατηρεί τι εξελίξεις και να προστατεύει μόνο τα συμφέροντά του. Έχουμε μια διμερή συμφωνία μεταβατική προσωρινή για την επίλυση συγκρούσεων μεταξύ ε, Καναδά και ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περασμένο φθινόπωρο έγινε αυτό και δουλεύουμε με κάτι αντίστοιχο με υπόλοιπες 15 χώρες για να διασφαλίσουμε τα δικαιώματά μας μέχρι ότου ξαναρχίσει να λειτουργεί το Σώμα Προσφυγών το επίσημο. Τα μέλη ήλπιζαν ότι γρήγορα θα λυθούν τα προβλήματα. Η μόνιμη λύση για το σώμα προσφυγών ε, απέχει ακόμα, είναι μακριά. Για να την πετύχουμε χρειάζεται να καταβάλουμε επιβρόσθετες προσπάθειες και για εξού και έχουμε καταλήξει αυτή την προσωρινή ρύθμιση και ελπίζουμε να την επεκτείνουμε και με άλλες χώρες. Ε, ένα ψήφισμα από το MC12 δεν είναι ρεαλιστικό. Πρέπει να μην έχουμε ε, υπερβολικές φιλοδοξίες για, για το εφικτό ε, σε σχέση με την Υπουργική Διάσκεψη των 12. Η Υπουργική Διάσκεψη Ministerial Conference είναι πολύ σημαντικό όργανο γιατί μπορεί να διαπιστώσει την κατάσταση και να ανοίξει κάποιους δρόμους για τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ. Όπως γνωρίζετε και όπως είπε και ο Πρόεδρος, ο Καναδός έχει αναλάβει τα ενία σε αυτή τη μεταρρυθμιστική ε, προσπάθεια. Έχουμε συγκαλέσει την ομάδα της ΟΤΑΒΑ, θέλουμε ενεργή συμμετοχή και ε, θέλουμε να επιδείξουμε πνεύμα ηγεσίας. Σκοπός της ομάδας της ΟΤΑΒΑ δεν είναι να καταλήξει σε προτάσεις και ιδέες για τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ. Θέλουμε να είναι ένα φόρουμ για να υπάρξει ανταλλαγή απόψεων και ιδεών μεταξύ μελών που φρονούν το ίδιο για το πώς μπορούν να ε, στηρίξουν αυτή τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια, υπ' αυτή την έννοια. Έχουμε καλέσει όσους έχουν ιδέες να έρθουν να μιλήσουν στα μέλη της ομάδας της ΟΤΑΒΑ, να δώσουν ε, απαντήσεις στα ερωτήματα, να προτείνουν ιδέες για το πώς θα προχωρήσουμε. Νομίζουμε ότι είναι συζητήσεις που κομίζουν με επιπρόσθετη αξία σε αυτή την προσπάθεια της μεταρρύθμισης του ΠΟΕ και θα συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Οι Υπουργοί θα συναντηθούν στα μέσα Μαρτίου στη ΝΟΤΑΒΑ για άλλη μια φορά για να συνεχιστούν οι συζητήσεις και να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε θετική έκβαση στην Υπουργική Διάσκεψη των 12 και ε, ε, ε, έτσι ώστε να λάβουμε καλύτερα υπόψη μας στη δουλειά μας την άποψη της βιομηχανίας και των παραγωγικών κλάδων. Δεν έχουμε αυταπάτες ότι η ομάδα της ΟΤΑΒΑΣ θα μπορέσει να λειτουργήσει ως τομή στις εξελίξεις, όμως είμαστε αισιόδοξοι. Πιστεύουμε ότι τα μέλη του ΠΟΕ θα μπορέσουν να προχωρήσουν τη δουλειά σε διάφορα πεδία και θα υπενθυμίσουν στην κοινή γνώμη πόσο σημαντικό είναι το όργανο αυτό τον 21ο αιώνα. Ο Καναδάς ε, είναι στοχοπροφυλωμένο στο η θετική έκβαση των διαπραγματεύσεων για τον αλλιευτικό κλάδο. Θέλουμε να διατηρήσουμε τα αποθέματα για τις μελλοντικέ γενιές. Πρέπει να πετύχουμε θετική έκβαση στις αλληλευτικές ενισχύσεις σε επίπεδο υπουργικής διάσκεψης 12 και αν τα καταφέρουμε θα αυξήσουμε την ε, αξιοπιστία του ΠΟΕ. Θα είναι ένα όργανο που θα έχει αποδείξει ότι χρειάζεται, ότι μας είναι απαραίτητο τον 21ο αιώνα. Είναι ευκαιρία να δείξουμε πρόοδο ε, και για την κοινή δήλωση ε, πρωτοβουλίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο αλλά και για την παροχή υπηρεσιών. Και τις εγχώριες διατάξεις. Πιστεύουμε επίσης ότι θα προτεύσουμε ε, στη δουλειά που πρέπει να γίνει για τις πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, με τις κοινέ πρωτοβουλίες για τη διευκόλυνση των ε, επενδύσεων. Θέλουμε να συνεργαστούμε με άλλες χώρες που φρονούν το ίδιο όπως εμείς στο επίπεδο της Υπουργικής Διάσκεψης 12 για να αντιμετωπίσουμε το θέμα της γεωργικής στήριξης σε εγχώρικο επίπεδο. Ο Καναδάς δουλεύει με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να έχουμε υπουργική δήλωση για το εμπόριο και την περιβαλλοντική αηφορία. Ε, νομίζω ότι είναι απολύτως απαραίτητο τα μέλη του ΠΟΕ να στείλουν ένα τέτοιο μήνυμα στην κοινή γνώμη με στην υπόλοιπη κοινωνία ε, στους καιρούς που ζούμε. Θεωρούμε ότι είναι ένα εφαλτήριο αυτό για να ενισχύσουμε το εμπόριο και τη γυναικεία δραστηριότητα και την περαιτέρω ανάπτυξη και απόκτηση δεξιοτήτων και ε, ικανοτήτων των γυναικών δεν θα είναι μια συνάντηση στην οποία θα σταυρώσουμε τα χέρια και δεν θα κάνουμε τίποτα. Ο Καναδάς πρέπει να συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση με διάφορα σχήματα για να υπερασπιστεί και να προστατεύσει το πολυμερές σύστημα είναι μακρόπνο εγχείρημα, εγχείρημα μακράς πνοής αυτής. Πρέπει να εργαστούμε προς κοινού στόχους και πιστεύω ότι τελικά θα σημειώσουμε επιτυχία. Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας. Με μεγάλη χαρά θα απαντήσω στις ερωτήσεις σας. So, uh, Σας ευχαριστώ. Είσαστε αισιόδοξο. Βλέπετε το ποτέρι μισογεμάτο. Όχι μισοάδιο. να δώσω το λόγο στον κύριο Σίμων, ο οποίο και είναι ο συμπρόεδρο από τη δική μα πλευρά τη Διευθυντική Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σα ευχαριστώ για την εισαγωγή αυτή. Ήταν πάρα πολύ αφηρημένη. Είπατε ο Καναδάς θα αγηθεί. Σας ρωτώ, έχετε μια πιο συγκεκριμένη ιδέα για το πώς θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα σε ό,τι αφορά το μηχανισμό επίλυσης διαφορών για το σώμα προσφυγής. Μιλάτε για την προετοιμασία του ΠΟΕ για τον 21ο αιώνα. Ίσως έχετε πιο συγκεκριμένες απαντήσεις όμως σε ό,τι αφορά τις κριτικές που ασκούνται προς τις πέρα από αυτά που μας παρουσιάσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Φαμπρέμπτ. Ευχαριστώ. Κύριε Ντεμπούρ. Ολλανδικής προέλευσης ε, το όνομά σας. Και συμβαίνει αυτό συχνά με τους Καναδούς φίλους μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισαγωγή σας και νομίζω ότι από τη μία μας δίνετε μια μας δινεται ρεαλιστική εικόνα σε ό,τι αφορά αυτή την 12η ε, ε, υπουργική συνδιάσκεψη, να μην είμαστε υπερβολικά φιλόδοξοι ότι θα ξεκινήσει μόνο η μεταρρύθμιση, αλλά παράλληλα μας δίνεται και κάποια ελπίδα ότι υπάρχει κάποια πλατφόρμα, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως μια πλατφόρμα για να προχωρήσουμε. Ας επιδείξουμε, αισιοδοξία είναι απαραίτητο άλλωστε τέτοιου καιρού. Πέρα από τα θέματα για το σώμα προσφυγής, αναφερθήκατε στην ομάδα της ΟΤΑΒΑ, τι κάνει και τι πρέπει να κάνει. Υπάρχουν και άλλες πρωτοβουλίες όμως. Η πρωτοβουλία, για παράδειγμα, της Νέας Ιλανδίας, ε, που συμμετέχει στην ομάδα της ΟΤΑΒΑ. η σύνδεση μεταξύ της μεταρρύθμισης του ΠΟΕ και των ε, κλιματικών ε, ζητημάτων. Αυτό το λέω και ως μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν θέλουμε να είμαστε ελπιδεφόροι και να έχουμε και ελπίδα για το μέλλον, θα πρέπει να προετοιμαστούμε για το μέλλον αυτό. Είναι λοιπόν πολύ ενδιαφέρον ότι στην υπουργική συνδιάσκεψη μπορούμε να προετοιμαστούμε εδώ και να υποστηρίξουμε τη Νέα Ζηλανδία που καθίσταται πρωτοπόρος δύναμη στον κόσμο σε ό,τι αφορά τον ΠΟΕ και σε ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος. Άλλες ρωτήσεις κανείς. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και τους πρέσβεις που μας παρουσίασαν τις απόψεις τους. Ο κύριος Βίνκλερ, το θέμα των βιομηχανικών επιδοτήσεων. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έγινε και μια συζήτηση προηγουμένως ε, για το θέμα αυτό. Ο τρέχον κατάλογος των επιδοτήσεων που απαγορεύονται σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ ε, είναι ανεπαρκής, θεωρείται, σε ό,τι αφορά τις τρευλώσεις που προκαλεί. Αυτό το διαπιστώνουμε και λειτουργεί βέβαια σε κάποιες ε, επικράτειες. Χρειαζόμαστε όμως παρόλα αυτά κάποιες νέες ε, απαγορεύσεις για επιδοτήσεις και κάποια καινούργια στοιχεία στη συμφωνία με τον ΠΟΕ. Ίσως και όπως τα βίντεο παιχνίδια, όπου καλείται κανείς ε, να διαλέξει όπλο και να ξεκινήσει τον πόλεμο. Ε, όλοι τώρα λοιπόν προσπαθούν να πάρουν το μεγαλύτερο όπλο. Έχουμε λοιπόν την εργαλειοθήκη, αλλά προφανώς θα πρέπει να προσθέσουμε στην εργαλειοθήκη αυτή κάποια καινούργια στοιχεία. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό. Πώς πιστεύετε ότι πρέπει να εξελιχθεί το θέμα των βιομηχανικών επιδοτήσεων σε ό,τι αφορά τα πλαίσια του ΠΟΕ. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος, ο επόμενος ομιλητής, ο κύριος Μπουρζουά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίασή σας και για το γεγονός ότι αναλαμβάνετε ηγεσία και ηγετικό ρόλο στο πολύ σημαντικό αυτό θέμα. Είπατε ότι ο ΠΟΕ δεν είναι στα πρόθυρα της κατάρρευσης αισιόδοξε κουβέντε. Γιατί νομίζω ότι ο πρώτος και βασικός μας στόχος είναι να σώσουμε τον ΠΟΕ. Για την ε, δήλωση ο πλευρά του Καζακστάν υπέρ του ΠΟΕ, υπέρ της πολυμερίας, θα ήταν πάρα πολύ προσδεκτή και υπέρ της βιωσιμότητας, υπέρ του εμπορίου βάσει κανόνων. Πιστεύετε ότι δεν υπάρχει αμφιβολία για τις αρχές αυτές. Οι συζητήσεις δηλαδή είναι πιο πολύ για τα πρακτικά ζητήματα, τα τεχνικά ζητήματα. Δεν αμφισβητείται η αρχή της πολυμέρειας στον ΠΟΕ. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά το σώμα προσφυγών. Ξέρουμε ότι είπα διατείνονται ότι υπάρχει α, υπερβολικά ευρύ πεδίο έχει αλλάξει η οικονομία από το 1995 όμως. Έχουμε το ηλεκτρονικό εμπόριο, έχουμε τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Αυτές οι λύσεις ε, για το σώμα προσφυγών, για την αλλαγή των κανόνων του ΠΟΕ και τη συμπερίληψη νέων κανόνων, πιστεύετε ότι δεν θα έπρεπε να είναι τμήμα αυτής της ε, υπερβολικά μεγάλης εντολής ε, σε ό,τι αφορά το τομέα για τον οποίο είναι αρμόδιο το Σώμα Προσφυγών. Και τρίτον, νομίζω ότι όλοι ανησυχούμε για το πώς πάνε οι αναπτυσσόμενες χώρες, ε, κρατικέ επιδοτήσει, ε, ενισχύσει κτλ. Πιστεύετε ότι θα πετύχετε πρόοδο στο θέμα αυτό. Η ε, κυρία Μπάρ, ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και τον πρέσβη που μας παρουσίασε η κυρία Ήμπνερ. Μας παρουσίασατε λοιπόν με διπλωματικό τρόπο ότι γίνεται και τις προσπάθειές σας. Είναι σαφές ότι προστίθεται μεγάλη αξία χάρη σε εσά στη συζήτηση για τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ. Θα συμφωνήσω όμως με τον Σβέν Σάιμον Μπορείτε να είστε λίγο πιο συγκεκριμένος σε ό,τι αφορά την συμμετοχή των ήπα και την κριτική που ασκείται εκεί. Και πώς μπορούν να βρεθούν απαντήσεις σε ό,τι αφορά τις προκλήσεις του ΠΟΕ, λαμβάνοντας υπόψη και την ήπα Σε ό,τι αφορά τη Βραζιλία τώρα και την ε, Νότια Κορέα, σε ό,τι αφορά το καθεστώς αναπτυσσόμενων χωρών το οποίο έχουν ε, παραχωρήσει οι ίδιοι στον εαυτό τους. Πιστεύετε ότι με τις αποφάσεις αυτές ε, φτάνουμε σε ένα σημείο όπου θα μπορούσε να συζητηθεί και το θέμα αυτό στην, ε, στον ΠΟΕ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Καβατσένη. Ευχαριστώ κύριε Πρέσβη και χαίρομαι και που βλέπω τόσους πολλούς προσκεκλημένους στις Βρυξέλλες. Η, η κλιματική αλλαγή και ήταν ε, στο επίκεντρο της ομάδας της ΟΤΑΒΑ. Θα ήθελα να ακούσω τη σκέψη σας ε, λόγω του Green Deal, αλλά επίσης και με το θέμα των δεσμεύσεων του Παρισιού θα ήταν πολύ σημαντικό να αντιμετωπιστεί και το θέμα της ε, κλιματικής αλλαγής σε σχέση με οποιαδήποτε μεταρρύθμιση του ΠΟΕ. Έχετε κάποιες ιδέες, ποιες θα ήταν οι συγκεκριμένες προτάσεις που ξεπερνούν τα εμπορικά και περιβαλλοντικά αγαθά θα με ενδιαφέρει να ακούσω τις απόψεις από αυτού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Πρέσβη για την ολοκληρωμένη ενημέρωση. Όλοι συμφωνούμε κατά πάσα πιθανότητα ότι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο ΠΟΕ απαιτεί ε, και έχει προκαλέσει την προσοχή των πολιτών των χωρών μας. Ο ΠΟΕ δεν έχει δημιουργηθεί απλώς για να υπάρχει ένας οργανισμός για το εμπόριο, αλλά επειδή ε, γίνεται εμπόριο μεταξύ των χωρών με σκοπό το όφελος των πολιτών. Οικονομικό, οικολογικό και κοινωνικό όφελος και ανάπτυξη. Οπότε, ρωτάω, έχει ήδη συζητηθεί η ομάδα της Οτάβα, στην ομάδα της Οτάβα το το άνοιγμα του ΠΟΕ και της μεταρρύθμισης της προκλήσης του 21ου αιώνα. Οποιαδήποτε χώρα μπορεί να πει ότι κυρίως με ενδιαφέρουν η αλληλεία ή η συνέχιση του γύρου της Ντόχα ή οτιδήποτε. Μια νέα αντίληψη όμως της εξέλιξης του ΠΟΕ. Πώς θα βρεθούν και οι κανόνες για όλα αυτά. Γιατί έχουμε συμφωνήσει ότι μόνο αν προχωρήσουμε βάσει κανόνων θα μπορούμε να εγγυηθούμε τη συμμετοχή όλων σε αυτό το εμπορικό σύστημα σε ισότιμη βάση. Πρέπει το σύστημα να μην έχει αποκλεισμού και να είναι δίκαιο. Μόνο λοιπόν το ελεύθερο εμπόριο συζητείται. Όπως είπε και η Ανακαβατσίνη, η κλιματική αλλαγή είναι πρόβλημα η κοινωνική και πολιτική και πολιτική απασχόληση είναι θέμα του ΠΟΕ. τουλάχιστον στην ομάδα της ΟΤΑΒΑ. Και τι θα γίνει με αυτούς που δεν έχουν ακόμα φτάσει εκεί. Ελπίζω ότι η Υπουργική του Νουρ Σουλτάν θα μπορέσει να προχωρήσει τα πράγματα και να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα με τρόπο που να ε, ενδιαφέρει και να ικανοποιεί την κοινή γνώμη. Να είμαστε πέρα από το αισιοδοξία ή αισιοδοξία. Πρόσωπος του, της Γαλλικής Γερουσίας. Μια παρατήρηση και μια ερώτηση προς τον ε, πρέσβη παρατήρηση. Δεν έχω την εντύπωση ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε σκοπεύουν την πλήρη καταστροφή του ΠΟΕ απλώ να μπλοκάρουν επειδή ποτέ δεν αντιλήφθηκαν, αντιλήφθηκε ο οργανισμός τις παρατηρήσεις των, των σε σχέση με τις υπερβολικές απαιτήσεις επί αρκετά χρόνια των δικαστών του. Μπόρεσα να το πω στον κύριο Ντενισές αυτό στη Γενέβη. Υπάρχει μια <coughs> στάση, ε, αλλά όχι επιθυμία καταστροφής. Επίσης, ε, ενδεχομένως θα μπορούσε να μας διευκρινίσει ο πρέσβης σε περίπτωση υποκατάστασης, σε περίπτωση ε, αποτυχίας του ΠΟΕ μπορεί να διευκρινίσει αν υπάρχει ε, πρόθεση να καταργηθούν όλες οι διαδικασίες μέχρι ότου επιστρέψουν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Χάνσεν. Ευχαριστώ τον κύριο Ντεμπέρ, με τον οποίο είχα συναντηθεί και στις αρχές Δεκεμβρίου στη Γενέβη μαζί με άλλους ε, εκπροσώπους ε, πρέσβης τρίτων χωρών μελών του Είχαμε συζητήσει το θέμα της αλίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, προετοιμάζεται για την μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλίας και Θάλασσας και αυτό έχει επικριθεί στη Γενέβη από πολλές τρίτες χώρες αλλά και από ε, καθώς και η ανακοίνωση της Προέδρου Βάντερ Λάιν για τον μηχανισμό προσαρμογής ε, μεθοριακό, στη μεθόριο του άνθρακα. Αυτό είναι ε, βασικά θέματα που απασχολούν την Ένωση στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του ΠΟΕ. Υπάρχουν, είναι αυτά εμπόδια. Ακούσαμε πολλά από τη πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών μπορείτε να μας μιλήσετε για αυτά και αν είναι δυνατόν να υπάρξει ένας μηχανισμός προσαρμογής του άνθρακα στα σύνορα που να συνάδει με τον ΠΟΕ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Θα κάνω κι εγώ μια ερώτηση. G33. Έκαναν δήλωση για τις ε, ενεξελίξεις διαπραγματεύσεις στην Διευπουργική, που κυρίως στηρίζεται στην τόχα στο γύρο της Ντόχα και το αίτημα να ολοκληρωθούν δύο από τα εκρεμή θέματα του κύκλου αυτού, το θέμα των ζωοτροφών συγκεκριμένα. Τι πιστεύετε, μπορεί να υπάρξει κάποιο συμβιβασμός για τον εξυγχρονισμό ή βρισκόμαστε σε κατάσταση όπου αυτό θα σταματήσει, θα μπλοκαριστεί. Γιατί αυτά είναι τα εκρεμή θέματα της Ντόχα. Πριν σας δώσω το λόγο, σκεφτείτε λίγο εσείς τις απαντήσεις και θα ζητήσω από τον Ντένις, τον ε, εμπειρογνώμονα της, του ΠΟΕ, από την Κομισιόν, να σχολιάσει λίγο όσα ακούσαμε από τον πρέσβη. Ευχαριστώ. Είμαστε στην ανταλλαγή απόψεων με τους αρμοδίους, γι' αυτό θέλω λίγες αντιδράσεις να παρουσιάσω και να τονίσω τα σημεία στα οποία θεωρούμε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι υπάρχει η σύγκληση με, με μας και με τον Καναδά. Ο Καναδάς όντως έχει επιδείξει πολύ ηγετικό πνεύμα εντός του οργανισμού. Έχουμε συνεργαστεί στενά. Άποψή μας είναι ότι πράγματι δεν καταραίει ο ΠΟΕ. Αυτό είναι ορθό. Συνεχίζει να λειτουργεί το σύστημα στη Γενέβη. Παρ' όλα αυτά, οι απειλές ε, είναι σημαντικές κατά τη γνώμη μας. Και είχαμε την ευκαιρία να το παρουσιάσουμε αυτό επανειλημμένο στην Επιτροπή σας. Και γι' αυτό θεωρούμε ότι η μεταρρύθμιση του ΠΟΕ είναι κάτι πολύ σημαντικό και πρέπει να αγγίξει όλους τους πυλώνες του οργανισμού, να μην περιοριστεί στο μηχανισμό επίλυσης διαφωνιών, πρέπει να επικταθεί και στον κλάδο της διαπραγμάτευσης και ε, στο, στις λειτουργίες που έχουν να κάνουν με τους κανόνες, με τη διαφάνεια. Όλα αυτά πρέπει να αναβαθμιστούν για να επιβιώσει το εμπορικό σύστημα που θα βασίζεται σε κανόνες. Σε ορισμένου τομεί έχουμε αναλάβει πρωτοβουλίε, έχουμε καταθέσει προτάσει. Σε άλλου τομεί ε, καταθέτουμε κοινέ προτάσει με τον Καναδά, ειδικά για το δεύτερο πυλώνα που έχει να κάνει με τη διαφάνεια για την παρακολούθηση και την επιπτία. Προσυπογράφουμε από κοινού προτάσεις για το πώς θα βελτιωθεί ε, το track record των notifications και έχουμε και μία νέα πρόταση που έχει να κάνει με τη λειτουργία των τακτικών επιτροπών του ΠΟΕ που ε, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο για την εύρυθμη καθημερινή λειτουργία του οργανισμού. Το ηγετικό πνεύμα του Καναδά μας έχει βοηθήσει ιδιαίτερως και στο πλαίσιο της ομάδας της ΟΤΑΒΑ υπενθυμίζω ότι στον Ταβός συναντηθήκαμε και μπορέσαμε και με τον Καναδά και με άλλα μέλη να να κηρύξουμε την έναρξη της πολιτικής διαδικασίας και έχουμε και αυτό το stop gap mechanism για την επίλυση των συγκρούσεων. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό το χρονικό σημείο στον Ταβός και η ομάδα της ΟΤΑΒΑ μπόρεσε να συναντηθεί και μετά άλλη μέλη για να συζητήσει το θέμα αυτό. Τώρα για τις προσωπτικές. Νομίζω ότι ο πρέσβης Τεμπούρ του Καναδά μας έδωσε μια πολύ συγκεκριμένη άποψη και ρεαλιστική πραγματική για το ποιε είναι οι προοπτικές της διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο της Υπουργικής Διάσκεψης 12. Ο κατάλογος του όντως μας ταιριάζει είναι τα θέματα, τα 12 είναι τα θέματα που πρέπει η Υπουργική Διάσκεψη των 12 να ε, ε, επεξεργαστεί, να δουλέψει. Είναι βασικά βήματα για να προχωρήσουν κάποια θέματα που είναι υποδιαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή. Και ελπίζουμε ότι ο Καναδάς συμφωνεί μαζί μας στο εξής. Η Υπουργική Διάσκεψη τον 12 δεν μπορεί μόνο να έχει θετική έκβαση για τα χ 10 σημεία, καλό είναι αυτό, αλλά πρέπει να λειτουργήσει και ως εφαλτήριο για να πάμε παραπέρα, να προχωρήσουμε πιο πολύ. Να αφουγκραστούμε τις ανησυχίες των μελών εδώ οι οποίοι πιστεύουν ότι ορισμένοι τομείς πρέπει να τύχουν περισσότερο μεταρρυθμίσεων. Δηλαδή, στον τομέα ε, του level playing field, να, έχουμε, ε, να μην έχουμε πια κενά στο βιβλίο με τους κανόνες και θα μιλήσουμε και το θέμα των βιομηχανικών ενισχύσεων αργότερα ε, ότι υπάρχει ένα ολόκληρο θεματολόγιο πέραν των εμπορικών αγαθών η δυνατότητα να διευκολυνθεί το παγκόσμιο εμπόριο και στην παροχή υπηρεσιών και στον τομέα των επενδύσεων. Και τέλος και πιο σημαντικό, μιλούμε για την ατζέντα της αηφορίας εντός του ΠΟΕ, η οποία είναι υπανάπτυκτη αυτή τη στιγμή, είναι πολύ λίγο ανεπτυγμένη, δεν έχει δοθεί ιδέουσα προσοχή από τα περισσότερα μέλη. Εμείς πιστεύουμε ότι λειτουργεί ως αγκίστρωση, ως βαρύδι που αξισορροπεί αυτή τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια. Πρέπει να δούμε πώς ε, ε, λειτουργεί συνιστόσα η διαπραγματευτική του ΠΟΕ. Πρέπει να ορίσουμε ε, καλύτερη προσέγγιση στο θέμα το, της ειδική και προτιμησιακής μεταχείρισης και στο θέμα των benefits που δεν επιβαρύνουν τα άλλα κράτη, τα άλλα μέλη. Είναι ένα εγχείρημα μακράς πνοής και ελπίζουμε να συνεργαστούμε με τον Καναδά και με άλλες χώρες και πριν και μετά και πέριξ της Υπουργικής Διάσκεψης 12, αλλά και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και εντός αυτής βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε ένα ερώτημα εσείς στο πίσω μέρος της αίθουσας, παρακαλώ. Από τη Σενεγάλη. Ε, έχετε το λόγο εσείς κύριε από τη Σενεγάλη. Εκτός μικροφώνου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συμμετάσχω στη συζήτηση διότι εδώ και κάποιες ώρες, εδώ και κάποιες στιγμές παρακολουθώ τις παρεμβάσεις των μεν και των δε. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι για τον ποια Αλλιώς ας, το, πετάξουμε όλο το εγχείρημα στο και Πρέπει όμως να έχει κανείς και την κατάλληλη ενέργεια για να αντέχει στις διαπραγματεύσεις. Το πρόβλημα είναι εξελικτικό. Όταν εξελίσσεται κανείς, πάντοτε πρέπει να αλλάζει να αλλάζει την πορεία του, να αλλάζει το ύφο του και τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσει τα, υψο... τα εμπόδια που υψώνονται μπροστά του. Πρέπει να αλλάξουν και διάφορες κανονιστικές διατάξεις. Καλό είναι να ευχηθούμε στην ομάδα της Οτάβα κάθε επιτυχία και να την πρικοδοτήσουμε με τις απόψεις και τις ιδέες μας. Μιλήσατε για level playing field και για ισορροπημένους κανόνες. στο ΠΟΕ είχαμε level playing field όταν είχαμε τις μεγάλες ε, χώρες, μόνο για αυτές να ισχύει και στο σώμα των προσφυγών το ίδιο. Όμως στι λιγότερο ανεπτυγμένε χώρες, στις υπανάπτυξες, στι αφρικανικές χώρες που έχουν μεγάλες δυνατότητε πλουτισμού, δεν έχει κανείς στρέψει το βλέμμα του προς αυτές τις χώρες. για να, έτσι ώστε να μην είναι ουραγή αλλά ταγή οι χώρες αυτές. Και γι' αυτό τίθεται εν κινδύνο η έννοια των ισορροπημένων κανόνων. Πρέπει η πλουτοπαραγωγική δυνατότητα των χωρών της Αφρικής να γίνει σεβαστή για να μπορέσει να βοηθήσει ε, όλους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Και θα προσπαθήσω να απαντήσω όλες αυτές τις ερωτήσεις, γιατί πολλές μαζέψαμε. Σε ό,τι αφορά το σώμα προσφυγών τώρα και το τι χρειάζεται να γίνει εδώ, να επισημάνω διάφορα στοιχεία. Καταρχάς, να είμαστε πολύ προσεκτικοί το πώς ε, ακούμε αυτά που μας λένε οι Αμερικανοί. Να διακρίνουμε επίσης μεταξύ της τακτικής και των μηνυμάτων που δεχόμαστε. Οι Αμερικοί λοιπόν, οι Αμερικανοί μας λένε διάφορα για το σώμα προσφυγής. Και θα πρέπει να τα ακούσουμε αυτά. Ένα εξ αυτών των στοιχείων το ανέφερε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε τρεις, ε, τρία, τρεις τομείς εργασίας του ΠΟΕ. Η επισέμεναν ότι το σκέλος των διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ δεν έχει λειτουργήσει καλά ως τώρα. Και γι' αυτό λοιπόν ε, καταλήγουμε να χρησιμοποιούμε υπερβολικά το σώμα προσφυγών. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε νέα πνοή σε αυτή τη διαδικασία και το σκέλος της διαπραγματεύσης. Έχουμε 170 σελίδες, 174 σελίδες ε, παραπώνων και ενστάσεων για το σώμα προσφυγών. Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα από τους Αμερικανούς και έχουν πρόσκληση προς την κατεύθυνση αυτή είναι να μας πούν τι πιστεύουν ότι χρειάζεται. Πιο λεπτομερώς. Επίσης να αναγνωρίσουμε ότι έχουν υπάρξει προβλήματα. Ο Καναδάς ε, δεν θεωρεί ότι τα προβλήματα είναι τόσο άσχημα όσο τα προβλήματα τα οποία επισημαίνουν οι Αμερικανοί. Ούτε θεωρούμε ότι είναι σωστό να μπλοκάρουμε τους διορισμούς στο σώμα προσφυγών. Αλλά θα πρέπει να ακούσουμε και τα προβλήματα που υπάρχουν. Και έχουμε δύο ενεργές διαπραγματεύσει, η μία λίγο πιο ενεργή από την άλλη. Η μία για την αλληλεία. Οι ΕΠΑ μιλούν ξεκάθαρα και αναφέρουν ότι υπάρχει ανάγκη να υπάρξει συμφωνία από την 12η Υπουργική Συνδιάσκεψη από αυτού. Άρα εδώ λέμε στους Αμερικανούς ουσιαστικά ότι λειτουργεί το διαπραγματευτικό σκέλος του ΠΟΕ. Επίσης αυτό θα έβαζε τον ΠΟΕ σε ένα καλό δρόμο για να αποδείξει ότι μπορεί να πραγματευτεί και θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. 14,6. Ε, είμαστε προς την κατεύθυνση επίλυσης των διαφορών αυτών. Αυτό λοιπόν θα καταδείκνυε ότι είμαστε σε θέση να ανταπεξελθούμε με θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Θα ήταν επίσης πολύ ενδιαφέρον για το πώς θα μπορούσε και θα έπρεπε να λειτουργήσει το SNDT. Ο Καναδάς θεωρεί ότι το SNDT δεν λειτουργεί σε κενό. χρησιμοποιείται στο, στη φάση σχεδιασμού των κανόνων. Θα πρέπει να πούμε λοιπόν ότι, κοιτάξτε, αυτοί είναι οι κανόνες. Αλλά επειδή είμαι αναπτυσσόμενη χώρα, χρειάζομαι ειδικού κανόνες για να τους εφαρμόσω. Και εδώ η διαφωνία σε σχέση με την αλληλεία θα μπορούσε να αποτελέσει ένα χρήσιμο παράδειγμα. Να μην αφήσουμε λοιπόν κατά μέρος της αντιπραγματεύσει για την Αλία είναι μια χρήσιμη ευκαιρία για να καταλήξουμε σε μια καλύτερη αντιμετώπιση του θέματος στα πλαίσια του ΠΟΕ και αντιμετώπιση του θέματος της βιώσιμη ανάπτυξης. Να κοιτάξουμε τώρα το θέμα της ε, μεταρρύθμιση του σώματος προσφυγών. Και τα δύο αυτά θέματα αλληλοσυνδέονται. Αυτό λοιπόν θα έδειχνε στους Αμερικανούς ότι είμαστε σε θέση να διαπραγματευτούμε και ότι είμαστε σε θέση να καλύψουμε και άλλα σκέλη της εργασίας μας ε, ως ΠΟΕ. Σε ό,τι αφορά το σώμα προσφυγών, είπα, ρωτούν πώς θα ενημερώσουμε τον, ε, τους κανόνες λένε να επανέλθουμε και να επιστρέψουμε στο 95, στους κανόνες του 95. Ενώ ουσιαστικά αυτό που χρειάζεται και αυτό που λένε είναι ότι θα πρέπει να καταστεί πιο κατάλληλος ο όγκος των κανόνων. Δεν είμαστε απαραίτητα αντίθετοι λοιπόν για τις βιομηχανικές επιδοτήσεις τώρα. Ο Καναδάς και νομίζω ότι όλη η ομάδα της ΟΤΑΒΑΣ είναι πολύ αισιόδοξη που η και η Ιαπωνία έχουν καταλήξει σε ένα κείμενο. Θέλουμε λοιπόν να εντάξουμε τους κανόνες εκεί. Δεν είναι σαφές προς τα που θα πάει αυτή η συζήτηση, πόσο γρήγορα θα κινηθεί και πώς θα συμβάλλει ο καθένας. Αλλά αυτός δεν είναι λόγος να μην κάνουμε τη συζήτηση. Από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Και χαιρόμαστε που η ΕΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιαπωνία έχουν ξεκινήσει αυτή τη συζήτηση. Θέλουμε και εμείς να συμμετέχουμε στη συζήτηση αυτή. Θεωρούμε όμως ότι αυτό το έργο θα πάρει χρόνο. Η 12η Υπουργική Συνδιάσκεψη θα είναι σίγουρα ένα σημείο στο οποίο μπορούμε να κάνουμε έναν έλεγχο για το που βρισκόμαστε, αλλά δεν πρόκειται να είναι έτοιμα τα πράγματα μέχρι τότε. Θα εργαστούμε σκληρά όμω για να σημειώσουμε πρόοδο προ την κατεύθυνση αυτή. Γενικά τώρα για το εμπόριο και την βιώσιμη ανάπτυξη. Διάφορες χώρες μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση, κινείται προς μια κατεύθυνση δήλωσης στα πλαίσια του ΠΟΕ για την βιώσιμη ανάπτυξη. Ελπίζουμε να αφιερώσουμε μισή ημέρα, την 8 Ιουνίου, πριν ξεκινήσει η διάσκεψη, για να γίνει καταρχάς μια δήλωση για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη και το πώς αυτά εντάσσονται στα πλαίσια του ΠΟΕ και για να τριγωνωθεί και μια σειρά εκδηλώσεων που θα ακολουθήσουν πάντα ε, την ίδια ημέρα για την ενδεχόμενη μεταρρύθμιση των επιδοτήσεων, για την πρωτοβουλία ε, της Κίνας, για τα πλαστικά, για την κυκλική οικονομία και για το περιβάλλον και την περιβαλλοντική ανταλλαγή. Αλλαγή. Αυτή η συζήτηση χρειάζονται εδώ και καιρό. Δεν πρόκειται να προσυπογράψουν και τα 164 μέλη, αλλά είναι καλό να ξεκινήσουμε από κάπου. Κάτι άλλο που χρειαζόμαστε και δεν υπάρχει ακόμα στα πλαίσια του ΠΟΕ. Είναι επίσημες σχέσεις μεταξύ του ΠΟΕ και των ε, διεθνών ε, περιβαλλοντικών οργανώσεων και συμβάσεων. Θα πρέπει να υπάρχει πιο ε, επίσημη λοιπόν διάτραση με την ICUN, τη UNAP και άλλες οργανώσεις. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον όπου η κατάρτιση των κανόνων δεν θα θεωρηθεί ως κακόβουλη και δεν θα θεωρεί ότι εξυπηρετεί σκοπούς προστατισμού, αλλά ότι θα προωθεί την οικονομική ανάπτυξη. Άρα αυτή η συζήτηση θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνει. Και για να επανέλθω στην Αλία η συμφωνία για τις επιδοτήσεις στην Αλία θα αποτελούσε ένα πάρα πολύ γύρω μήνυμα που θα καταδείκνει ότι είμαστε σε θέση να το πετύχουμε. Είναι σημαντική λοιπόν. Θα πρέπει να φροντίσουμε να πετύχουμε τη συμφωνία αυτή. Κάτι άλλο τώρα που ήθελα να αναφέρω. Το ανέφερα και στην εισαγωγή μου σε ό,τι αφορά την άλλη πλευρά των διαπραγματεύσεων και το γεγονό ότι οι υπα ότι το σκέλο διαπραγμάτευση του ΠΟΕΤΑ λειτουργεί. Σωστά. Η γεωργία αποτελεί το άλλο σκέλο. Όταν, ε, πρόεδρε, αναφέρθηκε το G33, πολλέ χώρε ζητούν κανόνες σε ό,τι αφορά την εγχώρια υποστήριξη και την ενίσχυση, άνωτατα όρια κτλ. Αλλά αν κινηθούμε προς την ε, γεωργία, η γεωργία και η σχετική συμφωνία θα πρέπει να είναι πολύ πιο ευρεία. Και επαναλαμβάνω ότι ούτε αυτό θα επιτευχθεί στην υπουργική διάσκεψη. Ελπίζω όμω στην 10η υπουργική διάσκεψη να κατακτήσουμε έναν δικό χάρτη για το πώ θα διαμορφωθούν οι διαπραγματεύσει, οι οποίε και θα αγγίξουν διάφορα θέματα σε σχέση με την ατζέντα την αναπτυξιακή της Δόχα. Και πάλι, επαναλαμβάνω, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα περιβάλλον που όλοι θα προωθήσουν τα συμφέροντά τους στις διαπραγματεύσεις και να μην δοθεί η εντύπωση ότι κάποιες χώρες κάνουν υπερβολικά πολλές υποχωρήσεις και κάποιες άλλες επωφελούνται μόνο. Όλοι θα πρέπει να προχωρήσουμε σε ό,τι αφορά αυτά που ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τη Γεωργία. Είπατε ότι θα πρέπει να εργαστούμε σε τρεις πυλώνες και βασικά και στη διαφάνεια ένας από τους τρεις πυλώνες αυτούς. Η διαφάνεια είναι εξαιρετικά σημαντική για τη λειτουργία του ΠΟΕ. Και εδώ πέρα έχουμε προβλήματα και οι έχουν επισημάνει και η ΙΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιαπωνία έχουν προβεί σε μία πρόταση κοινοποίηση την οποία υποστηρίζει ο Καναδάς. Εδώ λοιπόν αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην Γεωργία. Ελπίζουμε μέχρι την 12η ε, Υπουργική Διάσκεψη να έχουμε κάποιο δικό χάρτη για το πώς θα κινηθούμε στο μέλλον. Άρα, ο ΠΟΕ δεν είναι μόνο το όργανο επίλυσης διαφορών, βασίζεται σε τρεις πυλώνες εργασιών. Και αυτό σημαίνει ότι και εμείς ως μέλη του ΠΟΕ θα πρέπει να κοιτάξουμε τι γίνεται στην επικράτειά μας. Να είμαστε σίγουροι, για παράδειγμα, ότι πληρούμε τους κανόνες κοινοποίησης ότι υποστηρίζουμε όλα τα συστήματα του ΠΟΕ και ότι είμαστε διτεθειμένοι να τα συζητήσουμε. Να συζητήσουμε το θέμα των μεταρρυθμίσεων και στους τρεις πυλώνες. Ένα τελικό στοιχείο για το Σώμα Προσφυγών και τη μεταρρύθμιση του συστήματος επίλυσης διαφορών. Να μην σκεφτόμαστε την μεταρρύθμιση στο πλαίσιο της ε, επίλυσης διαφορών μόνο σε όρους μεταρρύθμισης του σώματος προσφυγής, να κοιτάξουμε πώς αντιμετωπίζουμε και πώς θα έπρεπε να αντιμετωπίζουμε διάφορα ζητήματα σε ό,τι αφορά εμπορικέ ε, διαφωνίες, κατά πόσον μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με άλλο τρόπο τις εμπορικές αυτές διαφωνίες και πάλι ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια πρόταση την οποία υπέβαλε. Μπορεί να βρεθεί ένας άλλος τρόπος ε, ε, επίλυσης χωρίς να φτάσουμε καν στο σώμα προσφυγών. Μπορούμε να ρυθμίσουμε τις διαφορές μας και τις διαφωνίες μας μεταξύ μας και να μειώσουμε την πίεση στην οποία υπόκειται το σώμα προσφυγών. Μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση για τη διαδικασία του πάνελ, αυτό το πρώτο επίπεδο επίλυσης διαφωνιών. Γιατί επικεντρωνόμαστε συνέχεια στο σώμα προσφυγών, γιατί εκεί επιμένει να γίνει μεταρρύθμιση η Αμερική, αλλά υπάρχει ένα γενικότερο σύστημα για την αντιμετώπιση των διαφορών και των διαφωνιών. Ελπίζω να απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις σας, 12 μου κάνατε και ήταν λίγο δύσκολο να απαντήσω σε όλες. Αν κάτι ξέχασα, να μου το επισπάνετε παρακαλώ. Τέλεια, τέλεια κύριε Πρέσβη. Καλή τύχη στις διαπραγματεύσεις. Μια τελευταία ερώτηση. Θα γίνει διακοινοβουλευτική διάσκεψη πριν από την Υπουργική ακριβώς, τον Ουρ Σουλτάν. Υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που επιθυμεί η ομάδα της ΟΤΑΒΑ από την διακοινοβουλευτική. Ίσως αυτή η τελευταία ερώτηση είναι η πιο άδικη Ένα από τα χειρότερα αποτελέσματα, ή μάλλον δύο πράγματα δεν θα ήθελα να προκύψουν από την 12η Υπουργική. Το ένα, να μην υπάρχει συμφωνία για την Αλία και το δεύτερο, ό,τι και αν προκύψει, να πούμε ότι πρόκειται για καταστροφή. Δεν νομίζω ότι θα είναι καταστροφή. Θα προκύψουν από την Υπουργική πολύ χρήσιμα πράγματα και αυτό το οποίο ελπίζω είναι ότι οι πολιτικοί ηγέτε του κόσμου θα πούνε ότι βεβαίως δεν είναι τέλειο, αλλά υπάρχει η βάση για να προχωρήσουμε. Έχουν μπει οι σπόροι στο χώμα. Πολλοί στο παρελθόν είχαν μιλήσει για καταστροφή. Και αν δείτε όλες τις ε, αποφάσεις που ελήφθησαν, που δεν ήταν όλες ε, πολυμερείς, ήταν εξαιρετικέ. Ακόμα και για τις πρωτοβουλίε των κοινών δηλώσεων. Παρά όλα αυτά έχουμε στο μυαλό ότι εκεί υπήρχε πρόβλημα. Κάποιο είπε κάτι νωρίτερα και το θυμήθηκα αυτό. Μια πολιτική δήλωση, υπουργική δήλωση. Δεν υπήρξε τέτοια στην ενδέκατη, ενδεχομένως να μην υπάρξει και στη δωδέκατη υπουργική. Σας καλώ να μην θεωρήσετε την έλλειψη πολιτικής δήλωσης ως αποτυχία της υπουργικής η Υπουργική θα πρέπει να κριθεί από τα επιτεύγματά της. Ας κινηθούμε προς μεταρρύθμιση, ας κάνουμε κάτι. Μια δήλωση που λέει για το ΑΒΓ δεν είναι τόσο σημαντική όσο το να γίνουν αυτά τα ΑΒΓ. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να, να δω κάτι που θα στηρίζει το σύστημα δεν χρειάζεται να είμαστε πολύ και να μιλάμε πάντα με αισιοδοξία, να παίζουμε το παιχνίδι της χαράς, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να έχουμε το θάρρος να συνεχίσουμε τη δουλειά μας. Ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σας. Ε, ελπίζω να σας βοηθήσουμε. Οπότε, στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται το σημείο 18, η συζήτηση για το σημείο 18 και περνάμε στο σημείο 19 που θα υπάρξει μια σύνδεση με βίντεο στις 11. Όπως είπατε λοιπόν και εσείς, το πιο σημαντικό θέμα της Υπουργικής ίσως να είναι το θέμα της αλίας. Οι διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ για τις επιδοτήσεις του, της αλίας ξεκίνησαν το 2001, εδώ και πολλά χρόνια, στην Υπουργική της Ντόχα. Έχουν ε, υπάρξει διάφορες φάσεις στην εξέλιξή τους. Ελπίζουμε, όπως είπε και ο πρέσβης, θα δούμε κάποια αποτελέσματα για το θέμα της αλληλείας στην 12η Υπουργική. Βεβαίως, το θέμα είναι ποια, πώς έχουν σήμερα τα πράγματα, ποια είναι τα εκρεμή ζητήματα και εμείς ως κοινοβουλευτικοί τι μπορούμε να κάνουμε. Χαίρομαι που ο πρέσβης Σανκιάτο Φίλης, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Κολομβίας στον ΠΟΕ, βρίσκεται εδώ μαζί μας μέσω βίντεο διάσκεψης. Είναι ε, ε, πρόεδρος της ομάδας κανόνων του ΠΟΕ, η οποία ασχολείται με το θέμα των ε, επιδοτήσεων στην Αλία. Κατόπιν θα ακούσουμε την κυρία Άλλη Στίπινγκ του Διεθνούς Ινστιτούτου Βιώσιμης Ανάπτυξης της Γενέβης. Είναι ειδική στις διαπραγματεύσεις για τις επιδοτήσεις στην Αλία. Κύριε Ντεβίλης, με ακούτε? Από ό,τι φαίνεται, με ακούτε. Ναι. Τέλεια. Σας δίνω το λόγο απευθείας. Thank you very much, much, Chair. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας απευθύνω το λόγο με τηλεδιάσκεψη. Οι άλλοι Στύπιν και εγώ θα ασχοληθούμε με τις διαπραγματεύσεις για τις ενισχύσεις στον αλληλευτικό κλάδο εντός του ΠΟΕ και από ό,τι μου είπαν θα ήταν πιο χρήσιμο από εμένα να κάνω μια μικρή εισαγωγή στη δουλειά που κάνουμε στο ΠΟΕ και μετά να έχουμε συζήτηση. Όπως ε, αναφέρθηκε, είμαι πρόεδρος της Διαπραγματευτικής Επιτροπής για τους Κανόνες στο ΠΟΕ, όπου ε, εκεί γίνονται οι διαπραγματεύσεις για τις ενισχύσεις στον αλευτικό κλάδο. Μιλώ με την ιδιότητα του Προέδρου, άρα, και δεν θα μιλήσω εξ ονόματος της ομάδας ή και ούτε καν της δικής μου χώρας, της Κολομβίας. Δεν μιλάω ε, ε, εξ ονόματος κάποιου μέλους του ΠΟΕ. Προσωπικές μου απόψεις είναι όλες και πρέπει να σας το πω εξ αρχής δεν δεσμεύουν κανέναν άλλο παρά μόνο εμένα τον ίδιο. Ποια είναι η εντολή μας. Οι διαπραγματεύσεις στον ΠΟΕ για τις ενισχύσεις για τον αλληλευτικό κλάδο εξελίσσονται εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Ξεκίνησαν το 2001, 20 χρόνια διαπραγματευόμαστε για το θέμα αυτό. αν ήταν παιδί που είχε γεννηθεί το 2001, σήμερα θα μπορούσε να ψηφίζει, να οδηγεί, να πίνει αλκοόλ. Θα μπορούσε επίσης να είχε γίνει πατέρας, αν ήταν μικρό αγόρι ε, αυτές οι διαπραγματεύσεις που γεννήθηκαν το 2001. Έχουν ε, αναπτυχθεί πλήρως και έχουν ε, φτάσει να αναπτύξουν δική του ζωή αυτές οι διαπραγματεύσεις. Έχουμε σαφή εντολή με βάση το 14,6 δηλαδή να εξαλειφθούν οι ενισχύσεις για τη λαθρέα, άναρχη, παράνομη αλία και να απαγορεύσουμε ορισμένα είδη ενισχύσεων που συμβάλλουν στην υπερβολική αλευτική δυνατότητα και στην πλεονάζωσα παραγωγή. Επίσης, αφές είναι ότι τα ηχθιαποθέματα παγκοσμίω απειλούνται και η κατάσταση συνεχώς επιδεινώνονται. Σύμφωνα με το ΦΑΟ, το 33% των ηχθιαποθεμάτων παγκοσμίων γίνονται αντικείμενο υπεραλίευση και τα περισσότερα αλλιεύονται πλήρως ούτω ή άλλω. Η αλληλευτική δραστηριότητα είναι μικρό κομμάτι του ΑΕΠ κάθε χώρα, όμω για ορισμένε χώρε και παράκτητε περιοχέ ε, είναι εξέχουσα ε, σημασία στο ζήτημα αυτό. 40 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίω ε, βρίσκουν τα προστοζήν αλλιεύοντα, ψαρεύοντα. Η αλληλευτική δραστηριότητα ανέρχεται στο 20% τη καθημερινή πρόσληψη πρωτενε για 2 δισεκατομμύρια ανθρώπου. Είναι το τρόφιμο που γίνεται αντικείμενο εμπορία στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό δεν συμβάλλει όμως να απασχόληση στο, στο ΑΕΠ και στο εμπόριο ε, αν εξαλειφθεί και τρία δις άνθρωποι πραγματικά θα δουν τη θέση τους να επιδεινώνεται ιδιαιτέρως. Δεν έχουμε ακριβή ιδέα του πόσα δαπανώνται στις ενισχύσεις για την ελευτική δραστηριότητα. Ενισχύσεις για να αλλιεύσει κανείς. Δεν μιλάω στις ενισχύσεις για να μην αλλιεύσει ή ενισχύσεις στις παρακτές κοινότητε για να διαφοροποιήσουν την ε, παραγωγή και τις οικονομική δραστηριότητα και δεν μιλάω και για ενισχύσεις για την ηχθειοκαλλιέργεια. Οι εκτιμήσει ποικίλουν για το πόσο διαμορφώνονται οι ενισχύσεις παγκοσμίω. 35 δι δολάρια το 2018 ήταν το ύψος των ενισχύσεων, 22 δι δολάρια είπα, ε, θεωρήθηκαν επιβλαβή, επιβλαβείς ενισχύσεις. Μπορεί κανείς να διαφωνήσει για τα νούμερα, ε, μπορεί να είναι μικρότερα τα ποσά και το μισό να ήταν είναι πάρα πολλά χρήματα να δαπανώνται για να προωθά κανείς μία μη αηφόρο κατάσταση. Με τη σαφή εντολή λοιπόν και με το πρόβλημα που θα πρέπει να λυθεί και έχοντας συζητήσει τις ενισχύσεις στην αλληλευτική δραστηριότητα για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα αναρωτιέται κανεί μα πού κολλάει το πράγμα, ποιο είναι το πρόβλημα. Καταρχάς δεν είναι τόσο απλές οι διαπραγματεύσεις. Υπάρχουν διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες για την ελίευση και τη διαχείριση της αλλευτική δραστηριότητας. Έχουμε την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της θάλασσας, τη συμφωνία για τα μέτρα για τους λιμένες, διάφορες διεθνείς συμφωνίες, κώδικες διοντολογίες ε, και ο Νουκάς αριθμός. Η απαγόρευση των ενισχύσεων απουσιάζει. Είναι σημαντική. Είναι ένα κομμάτι του παζλ και θα πρέπει να ταιριάξει και με τα υπόλοιπα για να ολοκληρωθεί το παζλ αν δεν είναι κάτι το εμφυλεγόμενο, θα πρέπει να μπορεί να ταιριάξει. Επίσης, απουσιάζουν αξιόπιστα στοιχεία και δεδομένα. Για παράδειγμα, η παράνομη αλληλεία θεωρείται ε, ως σημαντική, δηλαδή ότι είναι πολλά τα ποσάκια οι όγκοι που αλλιεύονται, αλλά κανείς δεν αναφέρει αυτά που ε, αλλιεύσε όταν το έχει κάνει παρανόμος. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, έχουμε 10 έως 23 εκατομμύρια τόνους αλλιευτικής δραστηριότητας παράνομες. Επίσης ε, έχουμε πρόβλημα με τον ορισμό του, τι η ενίσχυση και αντισταθμιστικά μέτρα, αλλά δεν κοινοποιούν τα κράτη-μέλη τις ενισχύσεις τους, δεν το κάνουν όλα τα κράτη-μέλη και όταν το κάνουν δεν παρέχουν στοιχεία για το ύψος των ενισχύσεων. Άλλοι χρησιμοποιούν διαφορετικό ορισμό όπως αυτός του ΟΣΑ ε, για να βαφτίσουν τις ενισχύσεις αλλιώς. Σε κάθε περίπτωση η συμφωνία αυτή θα είναι νομικώς δεσμευτική στο πλαίσιο του ΠΟΕ και γι' αυτό χρειαζόμαστε ακριβείς όρους που να υιοθετηθούν από τα 164 μέλη του ΠΟΕ και να ισχύσουν για όλους. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε άλλου άλλους ορισμούς όπως είναι οι ορισμοί που περιλαμβάνονται στη Συμφωνία για την Ελαθρέα Άναρχη Παράνομη Αλία. Όμως ε, δεν υπάρχει ορισμός για το subsistence, για την επιβίωση, για λόγους επιβίωσης δηλαδή ελευτική δραστηριότητα ή ε, για άλλου είδους όρους, για άλλους τέτοιους όρους. Και πρέπει να βρούμε τρόπους να τους παρακάμψουμε, τους όρους για τους οποίους δεν υπάρχει σαφής νομικός ορισμός. Πρέπει να δούμε και τα θέματα τα εμπορικά. Είναι η πρώτη φορά που διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του ΦΠΟ έχουν να κάνουν με την αηφορία. Δηλαδή, χρειάστηκε να αλλάξουμε κάπως νοοτροπία εντό του ΠΟΕ. Γνωρίζουμε ότι οι ενισχύσει έχουν αντίκτυπο στο εμπόριο και ε, το, το θέμα με τις ενισχύσει είναι πολύ σαφές παρόλο που δεν ξέρουμε ποιο είναι ο ύψο των συναλλαγών. Όμως το να έχουν οι ενισχύσεις αντίκτυπο στην αηφορία, αυτό είναι κάτι το καινοφανέ για μα. Κοιτάξτε, όταν κανείς μελετά ένα θέμα για 20 χρόνια, το καλό είναι ότι όλοι καταλαβαίνουν τα τεχνικά και το υπόβαθρο των θέσεων που υποθετεί κάθε μέλο στην ομάδα. Είναι σαφής η εντολή και σαφέστατη η δέσμευση από όλα ε, τα μέλη να υπάρξει αποτέλεσμα στην επόμενη υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ τον Ιούνιο στο Καζακστάν. Έχουμε μια δομή, μια διάρθρωση που θα ακολουθήσουμε για την επίτευξη συμφωνίας και κάποιες βασικές ιδέες, ε, κυρίως την απαγόρευση των ενισχύσεων για ηχθιαποθέματα που υπεραλλιεύονται και την απαγόρευση των ενισχύσεων για δραστηριότητες λαθρέας άναρχης και παράνομης αλληλεία. Τώρα μένει το θέμα των ενισχύσεων που, σε αλληλευτική δραστηριότητα που οδηγεί σε πλεονάζουσα παραγωγή. Το κάθε μέλος κρατάει Κατηγορεί το άλλο ότι προστατεύει την εγχώρια πολιτική. Δεν λέω ότι φταίει ο ένα ή ο άλλο ή ότι φταίνε όλοι. Μπορώ να πω το προφανέ. Ε, χρειάζεται περισσότερη δουλειά και θα πρέπει να είναι εντατική για να πετύχουμε συμφωνία στην Υπουργική Διάσκεψη στο Καζακστάν τον Ιούνιο. Όμως έχω έξι εργαλεία, έξι ανθρώπους που με διευκολύνουν. Ο καθένας έχει αναλάβει ε, διαφορετικό τομέα. Έναν για την ε, λαθρέα άναρχη παρανομαλία, άλλο για τα είδη που υπεραλλιεύονται και το άλλο για την υπερπλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα. Πέρσι τον Ιούλιο, ξέρετε, οι, αυτοί οι έξι facilitator κατάρτισαν ένα σχέδιο κειμένου, ένα προσχέδιο κειμένου πάνω στο οποίο βασιστήκαμε για να κάνουμε διαπραγματεύσει. Μόλι ανέλαβα την Προεδρία, του ζήτησαν να καταρτήσουν νέο προσχέδιο και το έκαναν στην τελευταία σύσκεψη και συνεδρίαση στα τέλη τη περασμένη χρονιά. Με την έλευση του 2020 δουλεύουν πάνω στο κείμενο, το βελτιώνουν. Και από ένα σημείο και μετά θα πρέπει όλα αυτά τα κομμάτια να αρχίσουμε να τα μαζεύουμε για να φτιάξουμε το puzzle, για να συντάξουμε ένα ολοκληρωμένο κείμενο για να δουν όλοι πώς συνδέονται οι παράγραφοι μεταξύ τους και πώς συνδέονται και οι έννοιες μεταξύ τους. Πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να απεικονίσουμε όλες τις απόψεις με ισορροπημένο τρόπο. Είναι πολύ σημαντικό βέβαια αυτό το κείμενο να μην, τον να μην το υπερφορτώσουμε, να το στολίσουμε και να καταλήξει να είναι χριστουγεννιάτικο δέντρο υπερφορτωμένο με διατάξεις και υποπεριπτώσεις, αλλά ούτε θα πρέπει να το αποδυναμώσουμε ούτως ώστε να καταλήξει να είναι ένα γυμνό ε, δέντρο χωρίς κλαριά. Ε, το σημαντικό είναι να είναι ένα ισορροπημένο κείμενο που να μπορέσει να εγκριθεί τον Ιούνιο στο Καζακστάν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω πάντα, συμβάλλει σε κάθε βήμα αυτή τη διαδικασία. Ε, ε, συνεργάζομαι στενά με τον πρέσβη τη Ευρωπαϊκή Ένωση στη Γενέβη, αλλά και με του συναδέλφου τη Βρυξέλλε. Είναι πολύ σημαντικό μέρο τη διαπραγματεύση η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εξέχοντα ρόλο και η σημασία της ε, επάγεται ευθύνη. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιδείξει ηγετικό πνεύμα, ε, πολιτική βούληση τους επόμενους μήνες. Τους επόμενους μισή μήνες, ούτε καν τέσσερις, για να μπορέσουμε να ε, έχουμε συμφωνία και θετική έκβαση. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει τα μέλη να παραχωρήσουν κάτι το ιδιαίτερο. Χρειάζεται όμως να επιδείξουν ευελιξία. Και αυτό ισχύει για όλα τα μέλη. Και τέλος, η επιτυχία αυτών των νυχτιαποθεμάτων είναι στα χέρια των ε, ε, κρατών μελών. Η αποτυχία θα είναι κάτι το αρνητικό για τα μέλη, για τον ΠΟΕ, για τους, για τους ωκεανούς και για τους λοιπούς στόχους ε, της αηφόρου ανάπτυξης πάνω στους οποίους έχουν συμφωνήσει οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε, έστω και με την μέθοδο της τηλεδιάσκεψης. Θα περιμένω μεγάλο ενδιαφέρον να συμμετάσχω στη συζήτηση και να ακούσω τις ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για την ενημέρωση για το πώς έχουν τα πράγματα για τις επιδοτήσεις και θα ήθελα να καλέσω την κυρία Τίπινγκ να πάρει το λόγο και να παρουσιάσει την δική της απόψη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να περιμένουμε λίγο μέχρι να κατέβει η, η παρουσίαση με τις διαφάνειες PowerPoint για να παρακολουθήσουμε και τις ε, λεπτομέρειες. Ευχαριστώ. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση που βρίσκομαι εδώ. Ε, Alice Tipping, ε, εργάζομαι σε ένα think tank στη Γενέβη, για σε Ίδρυμα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ονομάζεται AISD και παρακολουθούμε το θέμα για τις επιδοτήσεις στον, ε, στην Αλία εδώ και καιρό πολύ στενά. Και σήμερα μου ζητήσατε να σας εξηγήσω εν συντομία τι έχουμε επιτάπητος οι φίλοι μου από την Επιτροπή που παρακολουθούν τις διαπραγματεύσεις αυτές ε, θα καταλάβουν ε, πόσο λίγες λεπτομέρειες θα δώσω στα 10 λεπτά. Αλλά αν θέλετε φυσικά να επισέλθω σε μεγαλύτερο βαθμό λεπτομέρειες μετά. Βλέπετε Νομίζω τα δύο σημεία τα οποία θα ήθελα να επισημάνω σε αυτή την ε, λεπτομερή διαφάνεια. Πόσο παχές είναι οι γραμμές και τα χρώματα. Κοιτάξτε, δείχνουμε λοιπόν που έχουμε επίσημες ε, αξιολογήσει ε, των αποθεμάτων σε ό,τι αφορά την αλληλεία. Άρα, όσο πιο παχιά είναι η γραμμή, είναι πιο, όσο πιο πολλέ είναι οι αξιολογήσει και οι γραμμές, το χρώμα τη γραμμή επισημαίνει που υπάρχουν προβλήματα, που δέχονται πίεση στα εχθρία αποθέματα. Και βλέπουμε λοιπόν κάποιε περιοχέ τι οποίε γνωρίζουμε, στο Βορειοελλαδικό για παράδειγμα, στο Νότιο Ειρηνικό που υπάρχουν προβλήματα και έχουμε και αλληλεία σε κάποιε περιοχέ ε, όπου πραγματικά δεν έχουμε επαρκή στοιχεία. Οι πολύ πολύ λεπτέ γραμμέ για παράδειγμα, στον Ινδικό ωκεανό. Εδώ βλέπουμε ότι αντιμετωπίζουμε επιδοτήσει σε, σε ένα κλάδο που εξαρλεί από θέματα, αλλά δεν γνωρίζουμε απαραίτητα τι γίνεται παντού. Αυτό είναι το πρώτο σημείο, λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα δεδομένα και το πόσο δύσκολο είναι να γίνει προγραμματισμό και σχεδιασμό. Δεύτερο σημείο, το επισήμανε και ο πρεσβή Will, αυτό το θέμα για τις... πόσο δύσκολο είναι να καθορίσουμε πόσες επιδοτήσεις ε, στρέφονται και τελικά καταλήγουν στον κλάδο αυτό. Και εδώ βλέπετε μία ανάλυση που έγινε των ε, εργαλείων που είχαμε το 2009 στο σύνολό τους και το τι υπήρχε ως δεδομένα τότε. Η πλειονότητα λοιπόν των επιδοτήσεων για τις οποίες είχαμε στοιχεία πριν από 10 χρόνια πηγαίνει στην ε, μεγάλη κλίμακα αλληλεία. Και αυτό γιατί πολλέ από τι ε, επιδοτήσει για τι οποίε έχουμε εμ, ε, στοιχεία επιδοτούν λίγε επιχειρήσει. Και βλέπετε λοιπόν ότι όσο πιο πιο πολλά καύσιμα έχει κανείς, πιο πολύ όγκο έχει κανείς, όσο πιο πολύ υποφελείται από τις επιδοτήσεις. Και άρα δεν είναι σαφές και εύκολο να βρούμε τι επιδοτήσεις δίνονται από τον ΠΟΕ και από άλλους φορείς, αλλά κοιτώντα τι διατίθεται ως επιδοτήσεις, αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι πιο πολλές επιδοτήσεις δίνονται σε μεγάλη κλίμακας αλληλευτικές εκμεταλλεύσεις. Να κοιτάξουμε λοιπόν τώρα τον πίνακα. Αναφερθήκατε και εσείς σε κάποια τα θέματα αυτά. Κοιτάμε τρεις διαφορετικούς πυλώνες. Καταρχάς, η ιδέα της απαγόρευσης της επιδοτήσεων για την παρανομιλαθρέα και αναρχιαλία. Αυτό τονίστηκε στον στόχο 14.6. Η δεύτερη, η απαγόρευση των επιδοτήσεων σε ε, θέματα τα οποία είναι ήδη υποποίηση. Ήταν δηλαδή οι κόκκινες γραμμές στην πρώτη μου διαφάνεια. Ο τρίτος πυλώνας κανόνων είναι η γενικότερη ιδέα για την δημιουργία κάποιας ε, απαγόρευσης των επιδοτήσεων σε ό,τι αφορά ε, επιδοτήσεις μάλλον που συμβάλλουν στην ε, υπεραλίευση και την ε, υπερπαραγωγή. Αυτό ήταν στην ε, εντολή του ΠΟΕ. Και πολλά κράτη προσπαθούν να καταρτήσουν και να αποφασίσουν τι θα πρέπει να κάνει αυτή η συμφωνία. Υπάρχει σύμβαση λοιπόν σχετική και υπάρχουν διάφορα ζητήματα εγκάρσια ό,τι αφορά το όργανο επίλυση διαφόρων κτλ. Δεν θα επιδροθώ εδώ πέρα γιατί νομίζω ότι οι πρώτοι τρει κανόνε είναι αυτοί που είναι οι πιο σημαντικοί και ελπίζω να έχετε και να πάρετε αντίτυπο των διαφανειών πιο μετά, για την μικρά τα γράμματα. Γενικότερα λοιπόν ε, προσέγγιση είναι ότι θα πρέπει να απαγορευτεί η παροχή επιδοτήσεων σε σκάφη και σε εταιρείε αν υπάρχει απόφαση για ε, αναρχή και παράνομη ε, λαθρεαλία, αν υπάρχει δηλαδή τέτοια απόφαση από το κράτος που παρέχει την επιδότηση, από το ο κράτος, από το κράτος σημαίας ε, και από τις οργανώσεις ε, διαχείρισης της περιφερειακής αλίευσης. Γιατί μπορεί να εντοπίσουν τέτοια σκάφη στην επικρατεία τους. Μιλάμε λοιπόν για 130 σκάφη. Είναι μικρός ο κατάλογος, αν λάβει κανείς υπόψη, είναι εκατομμύρια σκάφη ο στόλος. Τελευταίο στοιχείο το οποίο υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να υπάρχουν διατάξεις από το κράτος λιμένα. Σε ό,τι αφορά τους προσδιορισμούς αυτούς. Αν λοιπόν προσδιοριστεί από το κράτος ε, λιμένα ότι ένα κράτος, ότι ένα σκάφος ε, κάνει παρανομή αλία, θα πρέπει να ισχύσει αυτός ο προσδιορισμός. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν έχει, από όσο ξέρω, ένα σύστημα το οποίο λίγο πολύ είναι ίδιο και παρόμοιο στην παρούσα φάση. Εδώ θα ήθελα να τονίσω το εξή. Υπάρχει μια γενική συμφωνία στον ΠΟΕ ότι η έκδοση ενό προσδιορισμού είναι δικαίωμα, όχι υποχρέωση. Αν υπάρξει τέτοιο προσδιορισμό, ο οποίο θα α, σήμαινε υποχρέωση επιδότηση. Δύο ερωτήματα τώρα. Θα έπρεπε να υπάρχουν δέουσε διαδικασίε και όροι σε ό,τι αφορά τους προσδιορισμούς αυτούς για να εξασφαλίσουμε ότι γίνεται με δίκαιο τρόπο σε ό,τι αφορά και την υποχρέωση επιδότησης που θα σήμεραν. Και θα πρέπει να υπάρχει κάποια στοιχεία αναλογικότητα σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, κάποιε ε, ίσονο σημασία παραβιάσεις... οι οποίες ενδεχομένω να μην σημαίνουν απαγόρευση πλήρη. Αυτό ήταν ο πρώτο πυλώνα, λοιπόν, σε ό,τι αφορά την ε, λαθρέα αναρχιαλία. Το δεύτερο θέμα, η ιδέα των επιδοτήσεων σε ό,τι αφορά θέματα ήδη υποπίεση. Η γενική προσέγγιση είναι να πούμε ότι θα απαγορεύονται οι επιδοτήσεις όταν υπάρχει θέμα υπεραλίευσης ε, και όταν έχουμε μία από τις δύο αυτές ε, παρακατόρους, όταν δεν υπάρχει σωστή αναπλήρωση των αποθεμάτων και όταν υπάρχει διαρκή μείωση του επίπεδου των αποθεμάτων. σε κάποιε περιπτώσει ενδεχομένω να υπάρχει υπεραλίευση δηλαδή, αλλά υπάρχει μια πορεία ανάκαμψη και θα, μπορέσουν, θα μπορούσε σε αυτήν την περίπτωση αυτή να επιτρέπουν οι επιδοτήσει. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εδώ, στο σχέδιο κειμένου, είναι να πούμε το εξή. Αν υπάρχει υπεραλίευση και μειώνονται τα αποθέματα, απαγορεύονται οι επιδοτήσει. Αλλά θα πρέπει να πληρώνουν και σχετικοί όροι. Οι νομικοί στην αίθουσα θα επισημάνουν κατευθείαν ότι υπάρχει το πρόβλημα του ποιο θα καθορίσει κατά πόσον υπάρχει ε, υπεραλίευση, θα πρέπει να υπάρξει κάποιο ορισμό βάσει των βιολογικών παραγόντων, μέγιστη απόδοση κτλ. ή θα πρέπει να υπάρχουν αρμοδιότητε και να αποφασίζουν οι εθνικέ ή περιφερειακέ αρχέ πότε υπάρχει υπεραλίευση και τι τεκμηρίωση θα πρέπει να υπάρχει για τι αποφάσει αυτέ. Είναι πολυτεχνικά λοιπόν τα θέματα αυτά και τα διέτρεξα γρήγορα-γρήγορα. Αυτό είναι λοιπόν ο δεύτερο πυλώνα, κατά πόσον υπάρχει υπεραλίευση. Και νομίζω ότι υπάρχει ένας, μια σαφή κατεύθυνση. Ξέρουμε πώ θα δημορφωθεί κατά πάσα πιθανότητα ε, ο κανόνα αυτό. Ο τρίτο πυλώνα είναι εντελώ διαφορετικό, ωστόσο. Η ιδέα ενό γενικότερου κανόνα για τι ε, επιδοτήσεις που εντείνουν την υπεραλίευση. Εδώ έχουμε διάφορε προσεγγίσει επιτάπητο. Τα κρατημέλη έχουν διαφορετικέ ιδέε, πολύ διαφορετικέ ιδέε για το πώ θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ο κανόνα αυτό. Μία προσέγγιση λοιπόν είναι η εξή. Να απαγορευτούν οι επιδοτήσει σε ό,τι αφορά το λειτουργικό κόστο και το κεφάλαιο μόνο για μεγάλε κλίματα, βιομηχανικέ αλλιευτικέ εκμεταλλεύσει. Αυτό θα εξαιρούσε λοιπόν και θα κάνει διάκριση μεταξύ μικρή κλίμακα και μεγάλη κλίμακα αλλιεύση. Και αυτό έχει σημασία ιδιαίτερα για τι αναπτυσσόμενε χώρε. Αυτή είναι μια προσέγγιση η οποία βασίζεται στο ότι δεν μπορεί να επιδοτηθεί σε καμία περίπτωση η μεγάλη κλίμακα αλλιεύση γραφτικέ εκμεταλλεύσει ε, εκτό του εθνικού εθνική επικράτηση. Μια δεύτερη ιδέα να υπάρχει μια ευρεία απαγόρευση σε όλε τι εκμεταλλεύσει ε, που συντείνουν και συμβάλλουν στην υπεραλίευση. Εκτό και αν υπάρχει κάποιο σχέδιο αντιμετωπίση τη υπεραλίευση, που πάλι πτύφεται το θέμα του τι σχέδιο θα είναι αυτό ακριβώ. Δεύτερο στοιχείο και υπάρχει το στοιχείο του πράσινου κουτιού. Όσοι παρακολουθούν τι διαπραγματεύσει για την Γεωργία στον ΠΟΕ θα την γνωρίζουν την ιδέα αυτή και την έχουμε δει σε διάφορες προτάσεις την ιδέα αυτή του πράσινου κουτιού. Να υπάρχει μια λίστα επιδοτήσεων που μπορούν να χορηγηθούν υπό όλε τις συνθήκες σε κάθε περίπτωση για την ανάπτυξη, για την ασφάλεια, για ανάκαμψη σε περίπτωση φυσικών καταστροφών, ενδεχομένω και μια ιδέα και σκέψη θα ήταν κατά πόσο θα επιτρέπονταν τέτοιε επιδοτήσει και πώ θα πρέπει να δημορφωθούν. Έχουμε και διάφορα άλλα είδη κανόνων στον πυλώνο αυτό. Μια περιστασιακή αντιμετώπιση και προσέγγιση που απαγορεύει τις επιδοτήσεις ιδιαίτερα όταν υπάρχει πλεονάζουσα ε, η αλίευση. Και πάλι επαφείται στα κρατημέλη, στα, στις περιοχές και στις περιφέρειες να καθορίσουν ε, το επίπεδο αυτό. Έχουμε την ιδέα της ε, απαγόρευσης ε, της αλίευσης εκτός, από την αποκλειστική, οικονομική της αποκλειστικής ζώνης των κρατών. Κάποιοι θα μιλούσαν για το ανοιχτό πέλαγος, κάποιοι θα μιλούσαν για αλλιεύση στο ανοιχτό πέλαγος και σε άλλες ε, οικονομικές, αποκλειστικές οικονομικές ε, ζώνες. Και επίσης τίθεται το θέμα των ε, σκαφών μεταπλοήγησης. Αυτές είναι λοιπόν, αυτή είναι η ποιοτική αν θέλετε κανόνες, ποιοτικούς τους αποκαλώ. Άλλα κράτη προτείνουν ποσοτικούς κανόνες που θα αποτυπώνουν και κάποιες από τις ιδέες που, έχουμε στις ακροτικές συμφωνίες. Μία ιδέα θα ήταν να διατηρηθούν οι επιδοτήσει σε συγκεκριμένο επίπεδο όμως και να γίνει διαπραγμάτευση για μείωση των επίπεδων επιδοτήσεων. Και για παράδειγμα, η εδώ με την Αυστραλία και κάποιε χώρε τη Λατινική Αμερική έχουν προτείνει τέτοιο είδου μοντέλο, να διαιρεθούν δηλαδή όλα τα μέλη για όλων των μελών του ΠΟΕ και όσοι έχουν μεγαλύτερη ποσοστό υπεραλίευσης να υπόκεινται σε πιο αυστηρές κανονισμούς σε ό,τι αφορά τα ανατοτά όρια για τις επιδοτήσεις και σε ό,τι αφορά τις ε, και η Κίνα επίση ε, πρότεινε και είναι ενδιαφέρον αυτό μια ποσοτική προσέγγιση. Είναι ένα από τα λίγα πράγματα στα οποία συμφωνούν η ΕΠΑ και η Κίνα. Εδώ όμω ε, προτείνουν μια πολύ διαφορετική ποσοτική προσέγγιση. Πολύ πιο μεγάλη ευελεξία για τι αναπτυσσόμενε χώρε ε, στη συνέχιση των επιδοτήσεων. Και ένα από τα βασικά θέματα το οποίο προκύπτει εδώ είναι το πώ θα δημορφωθεί ένα τέτοιο σύστημα. Θα πρέπει να υπάρχει μια διαπραγμάτευση μεταξύ των κρατών για το επίπεδο της μείωσης ε, και των επενδύσεων ή θα έπρεπε να υπάρχει μια πιο διαφανής ε, μορφή, ένας πιο διαφανής τύπος για τη διαμορφώση ε, του ύψους των επιδοτήσεων. Και πάλι, όπως βλέπετε στη διαφάνεια, έχουμε την έκτη προσέγγιση στον τομέα αυτό. Και είναι πραγματικά πολύ έντονες οι συζητήσεις για το ποια προσέγγιση θα επικρατήσει, κατά πόσο θα πρέπει να επικρατήσει ένα ευρετικό σύστημα μεικτό και τι συνέπειες θα έχει αυτό Τώρα, τα εγκάρσια θέματα δεν θα θέλαμε να τα κοιτάξουμε πολύ λεπτομερώς, αλλά νομίζω ότι στην παρούσα φάση λίγο πολύ επικρατεί συμφωνία για το γεγονός ότι επικεντρωνόμαστε στις επιδοτήσει σε ό,τι αφορά τις θαλάσσιες δραστηριότητες, όχι για τις καλλιέργειες και σε άλλες τομείς. όπως είπε και ο πρέσβης Ντεμπούρ και ο κύριος ε, Βίλς, αυτό που είναι ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις αυτές είναι ότι αποτελούν ένα μικρό κόσμο της ειδικής ε, και διαφοροποιημένης μεταχείρισης, γιατί πολλοί από τους μεγάλους ε, αλληλείς και τους μεγάλους τις μεγάλε χώρε επιδοτήσεων είναι αναπτυσσόμενε χώρε. Άρα χρειάζεται πιο πολύ ευλεξία για τι αναπτυσσόμενε χώρε διατείνονται. Αλλά αυτό δεν θα λειτουργήσει ω σύστημα στην προκειμένη περίπτωση. Γιατί πολλέ από τι προτάσει που τελικά έχουν κατατεθεί έχουν σκοπό να ισχύσουν σε όλα τα μέλη. Δεν βασίζονται σε ένα κλασικό μοντέλο διάκριση για τι ε, αναπτυσσόμενε χώρε με μια ειδική και διαφοροποιημένη μεταχείριση. Αυτά είναι λοιπόν διαφορετικά στοιχεία, τα οποία θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στην ειδική και διαφοροποιημένη μεταχείριση. Υπάρχουν, ε, θα μπορούσαν να υπάρξουν συγκεκριμένε εξαιρέσει, ε, γεωγραφικέ εξαιρέσει, ανάλογα με την ε, κλίμακα τη αλίευση, θα μπορεί να υπάρχει ταξινική αρρωγή και το καθεξή. Υπάρχουν λοιπόν πολλά εργαλεία στην εργαλειοθήκη για τον σχεδιασμό και την κατάρτιση τελικά μιας, ε, ενός κειμένου συμφωνίας για την αλία και ελπίζουμε όλα αυτά τελικά να αποτυπώνουν και την πραγματικότητα της παγκόσμιας οικονομίας σήμερα και τις πολιτικές ευαισθησίες προφανώς που επικρατούν σε επίπεδο ΠΟΕ. Και να υπογραμμίσω και ένα τελευταίο στοιχείο το οποίο το ακούσαμε ήδη πριν κλείσω. Από πλευρά κοινωνία των πολιτών θεωρούμε ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές αποτελούν κρίσιμο στοιχείο και για τον ΠΟΕ και τα μέλη τα μέλη του είτε οι κυβερνήσει ε, καταφέρουν να βρουν έναν τρόπο αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων με τον. Μάλλον τίθεται το κατά πόσο οι κυβερνήσει του ΠΟΕ μπορούν να βρουν τρόπο αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων που έχουμε σήμερα. Ελπίζουμε ότι η απάντηση είναι φετική και καταφατική. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστούμε πολύ. Είναι απολύτω σαφέ ε, και βεβαίω το πρόβλημα είναι πάντα στι λεπτομέρειε. Το να έχουμε μια σωστή νομικά δεσμευτική συμφωνία είναι ένα σύνθετο εγχείρημα που χρειάζεται συζήτηση σε όλες τις λεπτομέρειες. Δίνουμε το λόγο στις, ε, στα μέλη τώρα. Ευχαριστώ πολύ τους δύο εισηγητές. Πράγματι είναι πολύ περίπλοκο το πρόβλημα αυτό. Το είπε και ο μιλητής ότι διαπραγματευόμαστε από το 2001 Χαιρετίζω τον ΠΟΕ και τις προσπάθειες που καταβάλει, ώστε οι ενισχύσεις να συνάδουν με την αηφόρο αλία. Αυτό που επιθυμούμε εμείς. Η ευρωπαϊκή αγορά είναι η πιο ελκυστική αγορά του κόσμου. Η ευρωπαϊκή αλληλευτική αγορά και ο αλλιευτικός στόλος, ο ευρωπαϊκός πρέπει να πληρεί τα πιο αυστηρά πρότυπα σε επίπεδο εργασιακό, σε επίπεδο περιβαλλοντικό. Και ανταγωνίζεται ο ευρωπαϊκό αλλιευτικό στόλο με άλλου αλληλευτικού στόλου που δεν τηρούν τι ίδιε προποθέσει και που αλλιεύουν προϊόντα τα οποία δεν παρουσιάζουν καμία αηφορία ε, και πλημμυρίζουν τις αγορές μας με τέτοιου είδους αλλιεύματα. Μπορεί κανείς να θέσει σε αμφισβήτηση ορισμένα είδη ενισχύσεων, αλλά δεν μπορεί να δαιμονοποιήσει την αλληλεία. Ούτε μπορεί να αμφισβητήσει κάθε είδους ενισχύσεις και να μην θέλει καμία ποτέ. Προφανώς και συμφωνώ απολύτως. Πρέπει να απογορευτούν και να περιοριστούν οι ενισχύσεις σε αλλιευτικά σκάφη, σε αλλιευτικούς στόλους, τα οποία επιδίδονται στη λαθρέα παράνομη και άναρχη αλία, την αλία IUU. Και η Κομισιόν ε, κάνει πολύ καλή δουλειά. Προς αυτή την κατεύθυνση ψώνει κίτρινη κάρτα σε κάποιες χώρες, κόκκινη κάρτα σε άλλες. Δεν έχει κανένα νόημα να δίδονται ενισχύσει και επιδοτήσεις σε αλλιευτικούς στόλους χωρών που έχουν κίτρινη κάρτα ή κόκκινη. Δεν είναι όμως λογικό να έχουμε προτιμησιακό σύστημα για ορισμένες χώρες όπου υπάρχουν χαμηλοί δασμοί και επιτρέπεται να πουλήσουν τα λευτικά τους προϊόντα ή να τα αγοράσουμε από αυτούς, αλλά από την άλλη δεν μπορούμε να τους ενισχύσουμε γιατί έχουν κόκκινη κάρτα. Υπάρχει κάτι το οξύμορο δηλαδή εκεί. Συμφωνώ επίσης με το γεγονός ότι δεν θα πρέπει να δίδουμε ενισχύσεις που να οδηγούν στην πλεονάζουσα παραγωγή, ε, στην υπεραλίευση. Λογικό είναι αυτό και όλοι συμφωνούμε. Όμως έχουμε στραμμένο το βλέμμα μας στην Ευρώπη και είμαστε εξαιρετικά απαιτητικοί με τον αλευτικό μας στόλο. Όμως οι άλλες χώρες δεν κάνουν το ίδιο με τους δικούς τους στόλους. Ενισχύουν και μάλιστα ευρέως και επιδίδονται σε πολύ επισταμένες και έντονες και μεγάλες ενισχύσεις σε αλευτικούς στόλους που δεν σέβονται σχεδόν τίποτα. Δεν σέβονται τους στόχους του περιβάλλοντος, ούτε τις εκπομπές, τους στόχους για τις εκπομπές του ε, διοξιδίου του άνθρακα, δεν προσαρμόζουν την αλληλευτική δραστηριότητα, παρουσιάζουν καμία εφορία, δεν υιοθετούν προγράμματα συγκέντρωσης ε, ε, στοιχείων. Ε, υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα, ειδικά στις ασιατικές χώρες, όπου χρησιμοποιούν τα χρήματα αυτά για να αυξήσουν εκθετικά τον αλλιευτικό του στόλο και έχουν και ενισχύσεις για, την, για, για το κόστος λειτουργίας, που καλύπτουν το κόστος λειτουργίας. Και είναι άλλη η περίπτωση της η οποία ενισχύει με κρατικό χρήμα για, που καλύπτει το 30% της ναυπήγησης των αλλιευτικών στόλων εφόσον ναυπηγούνται σε ρωσικά ναυπηγεία. Είναι τεράστια εξοικονόμηση αυτή ε, για αυτούς τους επιχειρηματίες. Ε, ο ανταγωνισμός μετά είναι στρεβλός, δεν ανταγωνιζόμαστε με τις ίδιες συνθήκες. ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Πρέπει να συνεχιστεί η δουλειά. Ζητώ να μην δαιμονοποιήσουμε τις ενισχύσεις θεωρητικά για την αλία. Η αλία είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Έχουμε τεράστιο έλλειμμα υπερακμετάλλευση σε ορισμένε περιπτώσεις. Όμως στην Επιτροπή Αλίας προχθές λέγαμε ότι η κατανάλωση ήχθη από θεμάτων είναι πολύ ελληματική από το μέσο άνθρωπο και θα πρέπει να επενδύσουμε σε δραστηριότητες, π.χ. και ηχθειοκαλλιέργεια, η οποία συχνά έχει δαιμονοποιηθεί και αυτή δυστυχώς, ε, έτσι ώστε ο μέσο άνθρωπο να καταλώνει περισσότερο ψάρι. Να στοιχηματίσουμε στην ερασιτεχνική αλία, οι οποίοι βεβαίως οι μικροί αλίοι σέβονται πολύ περισσότερο το περιβάλλον, και να διατηρήσουμε τις ενισχύσεις στην αλληλευτική δραστηριότητα η οποία επιφέρει βελτιώσεις ε, πετυχαίνει εργασιακούς στόχους, περιβαλλοντικούς στόχους που βελτιώνει την κατάσταση στα αλλιευτικά σκάφη και διευκολύνει τη ζωή των αλλιέων. Εγώ επανειλημμένως έχω πει ότι θέλω οι αλλιείς όχι να αλλιεύουν περισσότερο, αλλά να αλλιεύουν καλύτερα και σε καλύτερες συνθήκες και για τους ίδιους. Η αηφορία έχει να κάνει με το περιβάλλον, αλλά όχι μόνο με αυτό. Πρέπει να υπάρχουν περισσότεροι ηχθείες ε, στα ύδατα, αλλά και περισσότεροι άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες που να εργάζονται στην αλλιευτική βιομηχανία. Για να πετύχουμε λοιπόν αυτή την τριπλή αηφορία χρειάζονται ενισχύσεις, ενάρετες ενισχύσεις και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λειτουργεί προς αυτή την κατεύθυνση. Ολοκληρώνω εκπέμποντας το μήνυμα που θέλω ε, να στείλω. Μη δαιμονοποιούμε σύσσωμες όλες τις ενισχύσεις γιατί αυτό είναι πραγματικά πολύ άδικο για τον αλλιευτικό κλάδο. Μόνο τις κακές ενισχύσεις για τη λαθρέα άναρχη παράνομη αλληλεία και ούτω καθεξής. Ευχαριστώ, επόμενο ομιλητή, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα αυτό. που αφορά την κοινοπολιτεία, μια ομάδα 54 χωρών, το συζητούμε συχνά. Ξέρουμε ότι σε ό,τι αφορά στην λαθρέα, άναρχη και παράνομη ε, ε, ε, υπάρχουν μέτρα επίγοντα που πρέπει να ληφθούν. Είναι επίγουσα η κατάσταση και πρέπει να αποκαταστήσουμε ε, τις βλάβες. Οι 54 χώρες της κοινοπολιτείας συμφωνούν με αυτό. Είχαμε την υπουργική διάσκεψη του Buenos Aires στην Αργεντινή το 2017 σε σχέση με το στόχους ε, τους αναπτυξιακούς της χιλιετίας και τους στόχους για την αηφόρο ανάπτυξη. Ε, αποφασίσαμε ότι μέχρι το 2020 ε, θα απαγορεύαμε 30 τόσες ενισχύσεις ε, αλληλευτικής δραστηριότητας που συμβάλλουν στην υπερπαραγωγή, στην πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα και θα πρέπει να εξαλείψουμε ενισχύσεις που ενισχύουν τη λαθρέα παρανομική αναρχιαλία. Όμως, ερωτώ, μετά από 20 χρόνια και διαπραγματεύσεων. Και παρακολουθώ παραθετικά να σας πω με μεγάλη προσοχή τη, τις πολύ σημαντικές ε, παρεμβάσεις σας στη συζήτηση αυτή. Μετά από 20 χρόνια όμως νομίζω ότι πρέπει να συμφιλειωθούμε με κάποιους όρους. Να καταλήξουμε σε μια φόρμουλα, σε μια διατύπωση, εν πάση περιπτώσει, για μια ισορροπημένη ε, αναπαράσταση και ύπαρξη ενισχύσεων. Πρέπει κάποια πρόοδο να σημειώσουμε, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά τα χρόνια. Και η θέση της κοινοπολιτείας σε αυτό το φόρουμ και σε κάθε φόρουμ είναι ότι πρέπει να συνεχίσουμε να πείθουμε περισσότερο με επιστημονικά όπλα, με επιστημονικά εργαλεία ότι πρέπει να βρεθεί μια κάποια ρύθμιση. Ευχαριστώ. τι λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από αυτόν? Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ενημερώσω την Επιτροπή για το αυτό που οποίο κάνουμε στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Εμείς ε, ως Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύουμε σε ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα της υπουργική. Αυτός, χωρίς αμφιβολία, είναι ο στόχος της προσπάθειας την οποία επιχειρούμε, ασχέτως των προκλήσεων που μάθηκαν στην αρχή της συνεδρίας από τον Πρόεδρο. Η θέση μας, καθώς το επιδιώκουμε αυτό, υποκινείται από το βασικό πολιτικ... τη βασική πολιτική ε, εντολή της διαπραγμάτευσης. Ο στόχος 14,6 ε, των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ολοκληρωμένη απαγόρευση επιδοτήσεων στην παράνομη λαθρέα και άναρχη αλληλεία και αυτό πραγματικά πρέπει να είναι απόλυτη απαγόρευση και το αποτέλεσμα θα πρέπει να περιλαμβάνει απαγόρευση των επιδοτήσεων, οι οποίες είναι επιβλαβείς λόγω του ότι ενισχύουν το πλεόνασμα της ικανότητας. Υπάρχουν μορφές υποστήριξης που δεν είναι επιβλαβείς, όπως ακούσατε, και δεν χρειάζεται να απαγορευθούν στο πλαίσιο αυτής της διαπραγμάτευσης. Υπάρχουν και θετικές επιδοτήσεις, προγράμματα επιδοτήσεων που περιλαμβάνουν ε, την στήριξη των ε, αλλιέων να μην αλλιεύουν ή να στηρίζουν τα, ε, τους αλλιευτικούς πόρους και στήριξη της σωστά διαχειριζόμενης αλλίας η αλληλεία ελέγχεται. Οπότε η επιδότηση δεν μπορεί να βλάψει την βιωσιμότητα του ε, αλληλευτικού αποθέματος. Αυτό θα μπορέσει να δημιουργήσει ε, κίνητρα για τα μέλη του ΠΟΕ ώστε να κινηθούν πέρα από τα, από τις επιβλαβείς επιδοτήσεις και να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση και σε αυτό έχει συνεισφέρει ε, βαθμιαία και σε άλλους τομείς στον τομέα της ε, ε, αγροτικής ανάπτυξης παραδείγματος χάρη. Και ταυτόχρονα εδώ δεν θα υπάρξει συμφωνία διακυβέρνησης των ωκεανών. Θα υπάρχει ένα άλλο πλαίσιο το οποίο θα συνεχίσει να λειτουργεί εκτός του ΠΟΕ. Το οποίο έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα ότι λειτουργεί με μηχανισμό που ε, ασχολείται με τις επιδοτήσεις γιατί έχει, ε, το έχει κάνει αυτό σε άλλους τομείς και έχει αν θέλετε το σχετικό λογισμικό. Υπάρχουν προτάσεις εκ μέρους σας στα διάφορα στοιχεία αυτής της διαπραγμάτευσης και επίσης έχουμε πρόσφατα πει στις πιο πρόσφατες φάσεις της διαπραγμάτευσης μέσω της, των πρόσφατων παρεμβάσεων του Επιτρόπου κ. Χόγκαν στις συνεδριάσεις του ΠΟΕ κάποιες ευελιξίες που θα λάβουμε υπόψη μας για να βοηθήσουμε τις διαπραγματεύσεις. Επισημαίνω το ότι, κατά την άποψή μας, ο αποκλεισμό των θετικών επιδοτήσεων μπορεί να είναι υπό, όρων, υπό όρους, δηλαδή το πράσινο κουτί, το green box, θα λάβει υπόψη του την, ε, ε, ένα πραγματικό πράσινο κουτί, το οποίο δεν θα αυξήσει την δυναμικότητα του στόλου. Επίσης, θα στηρίξουμε την απαγόρευση επιδοτήσεων που στηρίζουν την αλία στις ανοιχτές θάλασσες και στε, ε, ε σκάφη που φέρουν σημαίες ευκαιρίας και βεβαίως αυτό χρειάζεται περισσότερη επιτήρηση από ότι όταν η αλληλεία γίνεται εντός των υδάτων της χώρας και βεβαίως θα δούμε και το θέμα της ειδική και διαφοροποιημένης μεταχείρισης. Αυτό παραμένει σοβαρό θέμα στις διαπραγματεύσεις, είναι σύνθετο, επειδή είναι ακόμα πιο σύνθετο από ό,τι είναι σε άλλες εμπορικές διαπραγματεύσεις. Υπάρχει εδώ και ε, το θέμα της βιωσιμότητας στην καρδιά του ζητήματος και το περιπλέκει έτσι περαιτέρω. Και ε, ε, υποστηρίζουμε ότι ο τομέας αυτός δεν έχει ανοιχθεί επαρκώς από τα ε, κράτη-μέλη για να μπορέσουμε να πιστέψουμε ότι πράγματι προχωράμε προς επιτυχία. Πρέπει να είναι σαφές κατά την άποψή μας ότι για κάποια μέλη πρέπει να υπάρξει μεταβατική περίοδο με βάση πραγματικές ανάγκες. Αυτό δεν μπορεί να ισχύσει για μεγάλα λευτικά κράτη. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο και είναι σαφές ότι δεν θα στηρίξουμε αποτέλεσμα ε, για οποιαδήποτε μεταβατική περίοδο σε ε, επιδοτήσεων της παράνομης λαθρέας και άναρχης αλίας. Θα κλείσω λέγοντας ότι όπως δεδομένου ότι η διαπραγματική μας θέση ε, περιορίζεται από τους ε, συνομοθέτες ε, και τους εσωτερικούς περιορισμούς, θέλω να ενθαρρύνω τα μέλη της Επιτροπής να συνεχίσουν το διάλογο με τα μέλη της Επιτροπής για να βρεθούν λύσεις στο πλαίσιο του μελλοντικού πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου που ευθυγραμμίζεται με τον 14-6, ο οποίος πιστεύω πρέπει να αποτελέσει τη βάση της διαπραγματευτικής μας θέσης. Θέλω να ευχαριστήσω εσάς κύριε Πρόεδρε για την προσπάθεια που έχετε κάνει να ευαισθητοποιήσετε το Κοινοβούλιο για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και μία μικρή πρόσθετη ερώτηση επειδή το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι πλέον μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει κάποια αλλαγή στην διαδικασία, στην ε, τοποθέτηση μάλλον, τη διαπραγματευτική του Ηνωμένου Βασιλείου. Όχι. Το Ηνωμένο Βασίλειο άρχισε να εκφέρει γνώμη σε διάφορες συνεδριάσεις του ΠΟΕ σε ό,τι αφορά τον κώδικα κοινών εμπορικών πολιτικών που εποπτεύει το Ενωμένο Βασίλειο στα πλαίσια του ΠΟΕ. Παραμένουμε ε, στο πλαίσιο της ε, Συμφωνίας Αποχώρησης. Δεν αναμένουμε μεγάλες αλλαγές ε, τους επερχόμενους μήνες στο σκέλος αυτό. Και το επόμενο έτος δηλαδή. Θα συνεχίσουμε να προωθούμε τη διαπραγματευτική μας θέση η οποία ουσιαστικά δεν επηρεάζεται σε τίποτα από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Μάλιστα, άρα η συζήτηση για την Αλία θα είναι πλέον μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου. Μάλιστα. Πρέσβη Βουελής, θέλετε να πάρετε το λόγο και να σχολιάσετε τη συζήτηση που έλαβε χώρα εδώ. Βεβαίω, Πρόεδρε. Και θα ήθελα καταρχά να ευχαριστήσω για τα σχόλια τα οποία κάνατε. Όπω είπα και στην αρχή τη παρουσίασή μου, δεν μπορώ να επισέλθω σε μεγάλο επίπεδο λεπτομερία, δεδομένου ότι τα θέματα αυτά είναι αρκετά ευαίσθητα για κάποια κράτη και είναι ακόμα σε φάση έντονων διαπραγματεύσεων και συζητήσεων. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να σχολιάσω αυτά που άκουσα από τους διάφορους ε, φορείς. Είναι σημαντικό, θεωρώ, να κοιτάξουμε την εντολή και πώς διατυπώνεται η εντολή. Μιλά για το πόσο επιζήμιες είναι οι επιδοτήσεις που δίνονται και συμβάλλουν στην υπεραλίευση. Σε ό,τι αφορά την ε, παράνομη ελευθερία και αναρχιαλία. Αυτό είναι σαφές. Όταν ε, όμως στρεφόμαστε και σε έρευνες, μελέτες, ακαδηματικά έγγραφα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να εντοπίσουμε τι είδους επιδοτήσεις είναι αυτές που προκαλούν τη μεγαλύτερη ζημιά. Και οι επιδοτήσεις αυτές επί των οποίων συμφωνούμε ότι δεν είναι επιζήμιες, μήπως τελικά θα είχαν επιζήμιες συνέπειες. Αυτές σε αυτή τη φάση βρίσκονται οι διαπραγματεύσει και οι συζητήσει επί του παρόντο. Πώ μπορούμε να ορίσουμε κατά πόσο μια επιδότηση είναι ή δεν είναι επιζήμια. Και αυτή η συζήτηση οδηγεί τι διαπραγματεύσει προ μια κατεύθυνση. Θα πρέπει να επιληθούν τα ζητήματα αυτά σύντομα. Νομίζω ότι γενικώ πώ τα δύο πρώτα σχόλια είχαν να κάνουν με τη διάκριση ακριβώ επιζήμιων και μη επιζήμιων επιδοτήσεων. Και προφανώς για τον πρώτον ε, δεν μπορούμε να δαιμονοποιήσουμε την αλλιεύση, την αλλία στο σύνολό τη. Δεν είναι ο στόχος αυτός άλλωστε για των διαπραγματεύσεων. Στον ΠΟΕ νομίζω ότι όλοι τα μέλη αναγνωρίζουν τη σημασία της ε, αλλίας ε, και έχουμε και το 14 το οποίο μας δίνει εντολή και βλέπουμε λοιπόν τον στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης αυτών σε τι αποσκοπεί στην καλή χρήση των θαλάσσιων πόρων. Θα πρέπει λοιπόν να μην ε, ξεκινήσουμε να ενεργούμε όταν είναι ήδη πολύ αργά και όταν έχουν τελειώσει τα από θέματα, Ακριβώς αυτό που προσπαθούμε να καλύψουμε στην παρούσα φάση. Να αποφύγουμε προφανώς τη δαιμονοποίηση της αλίας, αλλά να αναγνωρίσουμε τη σημασία τις, στις σωστές διαστάσεις. Γιατί είναι πολύ ο κόσμος ο οποίος εξαρτάται από την αλληλεία. Θα πρέπει να επιλύσουμε ε, ένα ζήτημα το οποίο οδεύει προς το χάος, αν δεν ενεργήσουμε τώρα. Ε, αν κάτι ξέχασα από αυτά που αναφέρθηκαν, φυσικά να μου το πείτε, αλλά στο σημείο αυτό θα βάλω τελεία. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ε, Δεν μπορείτε προφανώς να είστε και πολύ λεπτομερείς. Και ενδεχομένω κάποια από τα σχόλια σας να μην ε, μπορούσαν να ταιριάσουν με τα υπόλοιπα σχόλια. Δεν είναι ερώτηση. Θέλω να πω ότι το Διεθνές Ταμείο για τη Θάλασσα και την Αλία, το Ευρωπαϊκό Ταμείο μάλλον, εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του με, σε σχέση με την κανονιστική διάταξη υπαριθμών 14. Χαίρομαι διότι είχαμε τη συζήτηση αυτή στην Επιτροπή Ίντα. Καλό θα ήταν να εξετάσουμε το εξής ενδεχόμενο. Η DigiTrade να έρθει εδώ και να κάνει κοινή συζήτηση με εμά στην Επιτροπή Ίντα και στην Επιτροπή Αλία, η οποία έχει πολλά να μα πει για τα θέματα αυτά. Αυτά ευχαριστώ. Thank ευχαριστώ πολύ και πολλές, ε, πολλά σχόλια ακούμε για το τι θα γίνει με τις αλληλευτικές επιδοτήσεις και με το 14.6 και την υπουργική απόφαση του 2017 σε ό,τι αφορά την Ινδονησία, μια χώρα που βασίζεται στη βιωσιμότητα και στον ωκεανό. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να βρούμε δημιουργικού τρόπου για να υπάρχει μια ισόρροπη προσέγγιση. Η συμφωνία όμως για την αλληλεία πώς ε, θα συνάδει με τις περιφερειακές οργανώσεις και τους στόχους που έχουν θέσει και υπάρχουν διάφορα εργαλεία τα οποία έχουν να κάνουν με την άναρχη και παρανομική ελαφρία αλληλεία και στην ε, ε, συμφωνία σε με για τα κρατηλημένα αυτό τι συνέπειες θα είχε, θα σήμαινε επιπρόσθετες ε, υποχρεώσεις. Ευχαριστώ πολύ, ο πρέσβης Βίλης. Ευχαριστώ. Και βλέπω ότι η ερώτησή σας ε, έχει μια διτή απάντηση για τον αντίκτυπο και τη σχέση μιας ενδεχόμενης συμφωνίας με τους RFMOs. Αυτή η απάντηση ενδεχομένω να σημαίνει αποκάλυψη κάποιων από συζητήσεων που γίνονται στη φάση των διαπραγματεύσεων. Γι' αυτό λοιπόν δεν θα ήθελα να επεκταθώ. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο στοιχείο, το δεύτερο στοιχείο σε ό,τι αφορά τη σχέση μιας ε, ενδεχόμενης τέτοια συμφωνίας και το άχθος που θα συνεπαγόταν η συμφωνία για τα κράτη-μέλη και τη διάδραση με άλλες συμφωνίες διεθνών οργανισμών. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να επισημάνω το εξή. Οι πιο πολλές συζητήσεις επί της ουσίας επί των πιλότων αυτών που εξήγησε η Alice Tipping Δεν έχουμε στην παρούσα φάση κάτι το οποίο να μας καταδεικνύει σαφώ ότι θα υπάρξουν πιο πολλά δικαιώματα, πιο πολλές υποχρεώσεις για τα μέλη του ΠΟΕ σε σχέση με το διεθνέ δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Δεν μπορούμε να καθορίσουμε τώρα τι αντίκτυπο θα είχε μια τελική συμφωνία, γιατί ακόμα δεν υπάρχει σαφής ε, διάκριση και σχεδιασμός των τομέων της συμφωνίας για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα. Θα ήθελα να ακούσω όμως την πιστεύει και άλλες από αυτόν. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρέσβη. Με τα μεγάλη χαρά σας ακούσαμε και καλή τύχη στις διαπραγματεύσεις. Καλή επιτυχία. Η κυρία Τίπινγκ. Μπορείτε να ανακεφαλαιώσετε ενδεχομένω. Και πάλι η τελευταία ερώτηση είναι η πιο άδικη. Δεν θα προσπαθήσω να ανακεφαλαιώσω τη συζήτηση. Θα απαντήσω όμως στην πρόσκληση να δώσω περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες στην ερώτηση του Συμπροέδρου για το πώς ε, ποια είναι η σχέση της παρούσας συμφωνίας με τις υφιστάμενες υποχρεώσεις βάσει του δικαίου της θάλασσας. Παράδειγμα, το πρώτο γενικό θέμα είναι ότι τα μέλη έχουν απόλυτη συνέστηση ότι εδώ δημιουργούν κανόνες για επιδοτήσεις στο πλαίσιο του ΠΟΕ πέραν του μεγάλου αριθμού κανόνων και υποχρεώσεων του δικαίου της θάλασσας και άλλων περιφερειακών συμφωνιών. Άρα λοιπόν όταν μιλάμε για ε, επιδοτήσεις στο πλαίσιο της παράνομης λαθρέας και αναρχής Υπάρχει ένα πλαίσιο που έχει θεσπιστεί από περιφερειακούς οργανισμούς διαχείρισης αλίας και ένα από τα ερωτήματα που τίθενται, που δείχνουν την ε, ευαισθησία είναι είναι σωστό να ε, επιβάλλει κανείς ε, κανόνες ορθής διαδικασίας σε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν θέλω να επισέλθω ιδιαίτερα στην αμφισβήτηση αυτών των καθορισμών, των προσδιορισμών, με συγχωρείτε, Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα. Υπάρχει ένας τρόπος που μπορεί να προσδιοριστεί η κατάσταση ενός αποθέματος είναι μέσω των περιφερειακών ε, ε, οργανισμών και κάποιοι, οργανώσει κάποιες οργανώσεις έχουν μηχανισμούς. Τα μέλη θέλουν τις αποφάσεις αυτές να τις χρησιμοποιήσουν, να να τις χρησιμοποιήσουν, αλλά υπάρχει πάντοτε το θέμα του να εξασφαλιστεί ότι είναι σωστά διατυπωμένες και ορθά ε, έχουν ληφθεί οι περιφερειακές αποφάσεις και των κανόνων του ε, ΠΟΕ. Υπάρχει λοιπόν μια μεγάλη ένταση ε, στις διαπραγματεύσεις. Και μια τελευταία παρατήρηση, να υπογραμμίσω κάτι που πολλοί το έθεσαν δεν είμαι ειδική στις εσωτερικές διαδικασίες της Ένωσης, εξ όσων αντιλαμβάνομαι όμως το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο βρίσκεται στη φάση του σχεδιασμού του ακόμα και άρα ίσως η Επιτροπή σας έχει την ευκαιρία να συνεργαστεί στενά με την Επιτροπή Αλίας για να υπάρξει κάποια συνοχή ανάμεσα στα ε, αυτά που επιτυγχάνουμε στον ΠΟΕ και στα εσωτερικά μέτρα. Ε, ο ΠΟΕ είναι μια ευρύτερη κοινότητα και μετά τις διαπραγματεύσεις έχει στραφεί ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση για ε, καθοδήγηση. Είναι από τους μεγαλύτερους αλληλευτικούς οργανισμούς και η θέση που αλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τους άλλους μεγάλους μεγάλες αλληλευτικές δυνάμεις θα καθορίσει το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πάντοτε ε, προσπαθούμε να ξεφύγουμε από την κλειστή αντιμετώπιση και η Επιτροπή Αλίας είχε προσκληθεί στη σημερινή συζήτηση. Βεβαίως υπάρχει πάντα περιθώριο βελτίωσης, αλλά ε, το δεχόμαστε. Λοιπόν, και πάλι ευχαριστούμε κύριε Βουίλης, ευχαριστούμε κυρία Τίπινγκ και ας ελπίσουμε ότι ε, θα έχουμε επιτυχημένη υπουργική τον Ιούνιο. Στο σημείο αυτό Ολοκληρώνεται η συζήτηση για το θέμα 19. Περνάμε κατευθείαν στο 20. Το σημερινό τελευταίο θέμα είναι το θέμα της τριμερούς ε, συνάντησης ε, στην προσπάθεια εξυγχρονισμού των κανόνων που αφορούν συγκεκριμένα τις βιομηχανικές επιδοτήσεις. Ο Ντένις θα μιλήσει για αυτά σε σχέση με την ε, συζήτηση Ιαπωνίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να σας ενημερώσω για τη διαδικασία αυτή, η οποία ε, ξεκίνησε στις 14 Φεβρουαρίου και είναι χρήσιμο για μας να σας ενημερώνουμε για το τι καλύφθηκε από τις συζητήσεις και προς τα που ε, κινούμαστε. Ευθύς εξ αρχής θα πω ότι στόχος ε, της Ένωσης, ε, ε, η οποία είναι πλάκη σε μια υπουργική τριμερή συνάντηση, υπουργική συνάντηση Υπουργών Εμπορίου με τον Επίτροπο, είναι να συνεργαστούμε με τους δύο αυτούς εταίρους μας, ώστε να καμφθούν οι παρεμπίπτουσες επιπτώσεις διαφόρων ε, πρακτικών στρέβλωσης της αγοράς που παρατηρούμε στο εμπόριο και αυτό να το επιτύχουμε με βάση λύσεις που θα στηρίζονται σε κανόνες στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Δηλαδή, εμείς ε, θεωρούμε ότι εδώ έχουμε μια ε, ένα φυτόριο για τους μελλοντικούς κανόνες του ΠΟΕ και έχουμε τρεις βασικές τάσεις ε, γραμμές εργασίας, πολλή δουλειά ανάμεσα στις ε, ε, υπουργικές συναντήσεις, τρεις ε, τομείς δουλειάς. Πρώτον, το θέμα, το, τα βιομηχανικές επιδοτήσεις, το φαινόμενο της, ψευ, της αναγκαστικής μεταφοράς τεχνολογίας και εν γέννη στην ανάγκη να ενισχυθούν ε, οι συνθήκες που θα ε, καθοδηγούν την αγορά. Έτσι στις 14 Ιανουαρίου συναντήθηκαν οι τρεις υπουργοί στη Ουάσιγκτον και εξέδωσαν κι άλλη μία κοινή δήλωση η οποία ανακεφαλαιώνει μάλλον ε, λεπτομερώς ε, τις συζητήσεις. Μία από, ένας από τους τομείς όπως είπαμε είναι οι βιομηχανικές ε, επιδοτήσεις και βεβαίως τίθενται και άλλα θέματα στα οποία υπάρχει σύγκληση και συνεργασία στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Αυτό έχει άμεση σχέση κατά την άποψή μας με την γενικότερη προσπάθεια μεταρρύθμισης του ΠΟΕ που συζητήθηκε προηγουμένως κυρίως με σκοπό να επιτευχθεί ο στόχος της επανισορρόπησης του συστήματος ε, υποχρεώσεων και δικαιωμάτων και την προσπάθεια μεταρρύθμισης. Όσον αφορά τις βιομηχανικές επιδοτήσεις, θέλω να εξηγήσω πώς, ε, πώς, πού βρίσκεται η διαδικασία ως εξής. Η τριμερής διαδικασία έχει κατανοήσει ότι αυτή τη στιγμή το εργαλείο που έχουμε για να ε, υπάρχει ισοτιμία ε, στο Διεθνές Εμπορικό Σύστημα που είναι το σύστημα επιδοτήσεων και αντισταθμιστικών μέτρων δεν είναι αποτελεσματικό πλέον. Έχει φτάσει τα όρια του. Ως εκ τούτου είναι ε, αποτελεσματικό μεν για την αντιμετώπιση κάποιου είδους επιδοτήσεων, κυρίως αυτές που έχουν σχέση με τις εξαγωγές και αυτές που αφορούν το χαμηλό περιεχόμενο, δηλαδή αυτές που εμπίπτουν στις τρέχουσες κατηγορίες απαγορευμένων επιδοτήσεων. Πιστεύουμε όμως ε, ότι υπάρχει ανάγκη να κατέβει ο πύχης ε, στον τομέα των εμπορικών επιδοτήσεων λόγω του βάθους και του εύρους του προβλήματος. Αυτό λαμβάνει η χώρα σε ένα περιβάλλον όπου διαπιστώνουμε πολλές μορφές ε, βιομηχανικής ε, επιδότησης σε κάποιους ε, χώρους και επίσης την περιορισμένη ικανότητα της διεθνούς κοινότητας να πειθαρχήσει εδώ. Ποια είναι η κατάσταση. Η δήλωση εντοπίζει έξι συγκεκριμένους τρόπους με τους οποίους οι τρεις εταίροι θεωρούν ότι θα πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω αργότερα από τον ΠΟΕ ως νόμους. Πρώτον, με τον αποκλεισμό των άνευ όρων ε, επιδοτήσεων. Δεύτερον, με τον εντοπισμό διάφορων επιβλαβών επιδοτήσεων που είναι επιβλαβή σε τέτοιο βαθμό ώστε να επιδοτούν, ε, να δικαιολογεί την ανάγκη ε, αναστροφής του ε, βάρους της απόδειξης από τους εταίρους, δηλαδή να, ε, ε, να αντιστραφεί το ε, τεκμήριο απόδειξης. Κατά την άποψή μας είναι ένα πολύ ισχυρό πειθαρχικό μέσο στο σύστημα και ένα, μια, βεβαίως τα κράτη πρέπει να αποδείξουν τι κάνουν και οι επιδοτήσεις πρέπει να είναι διαφανείς. Η τρίτη σειρά, το τρίτο κουτί αν θέλετε που εντοπίστηκε είναι η διεύρυνση του καταλόγου των ε, αρνητικών εμπορικών επιπτώσεων. Αυτό σημαίνει ότι θα εισαχθούν νέες κατηγορίες σοβαρών ε, βλαβών που οδηγούν σε στρέβλωση η τριμερής διαδικασία έχει εντοπίσει τρόπους με τους οποίους θα καταστεί δυνατόν να βελτιωθεί ο μηχανισμός κοινοποίησης της διαδικασίας ASCM και έχει εντοπίσει τρόπου ε, τρόπους με τους οποίους η χρήση ε, ενός δίκτυ εκτός χώρας για για τις αντισταθμιστικές επιδοτήσεις να διευκολυνθεί. Η έκτη παράγραφος του, ε, της δήλωσης ασχολείται με το, θέμα του δημόσιου φορέα που είναι ένας ε, τομέας που υφίσταται ήδη. Οι τρεις εταίροι συμφώνησαν ότι ο παρόν ορισμός δεν επιτρέπει ε, επαρκή στόχευση διαφόρων επιδοτήσεων που χορηγούνται από δημόσιους οργανισμούς ε, όπως που καλύπτονται από τον τρέχοντα ορισμό. Και όσον αφορά την αναγκαστική μεταφορά τεχνολογίας, υπάρχει η διατύπωση ότι η ανάγκη να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, γίνονται τεχνικές συζητήσεις ώστε και πάλι να μπορέσει να εποαστεί, ε, να εποαστούν κανόνες ε, στο μέλλον για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Ε, προχωρούμε με το προϊόν αυτής της προσπάθειας. Πρώτον, όπως είπε και ο κύριος Μπορ σήμερα, Έχουμε περάσει ένα κατόφλιο ε, στην οριμότητα της τριμερούς αυτής συζήτησης και οι εταίροι αποφάσισαν να διευρύνουν ε, την ε, συμμετοχή και με άλλα μέλη που θα ήθελαν ίσως να ενταχθούν. Αυτή η προσπάθεια έχει ήδη ξεκινήσει. Πρώτον, με μια ομάδα πιθανώς ομοειδεατών, άλλες χώρες δηλαδή, που θα έχουν την ίδια άποψη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπε και ο Επίτροπος, σκοπό έχει να συνεργαστεί με κάποιους συμμετέχοντες για να κάνει διερευνητικές συζητήσεις ενώπιση των διαπραγματεύσεων. Ελπίζουμε ότι αυτό θα γίνει ε, ε, στην περίοδο της 12ης Υπουργικής περίπου. Κατά την άποψή μας, η δια η διάρθρωση αυτής της προσφάδειας ε, ε στα πλαίσια μιας αρχιτεκτονικής με τη συμμετοχή του ACM, ASCM υπάρχουν παράλληλες συζητήσεις και με άλλα μέλη του ΠΟΕ. Έχουμε διμερείς συζητήσεις με την Κίνα ε, δεδομένου του βάρους της στην παγκόσμια οικονομία. Αυτό γίνεται στο πλαίσιο της συζήτησης διμερούς ομάδας εργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνα για, Κίνας για την μεταρρύθμιση του ΠΟΕ. Είναι μια από τις ομάδες συζητήσεις όπου ε, υλοποιείται η, διά, η δήλωση διάσκεψης κορυφής που έγινε πέρυσι που δεσμεύτηκαν οι ηγέτες να ε, ε, εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους Γι' αυτό το θέμα των ε, ε, βιομηχανικών επιδοτήσεων, μια διαδικασία που είναι παράλληλη και συμπληρωματική με την τριμερή ε, διαδικασία και θα συνεχιστεί μέχρι και το Μάρτιο. Έτσι έχουν τα πράγματα όσον αφορά την τρέχουσα κατάσταση και τι ε, υπάρχει πίσω από την κατάσταση των ε, επιδοτήσεων και την πολιτική δήλωση των τριών υπουργών και πώς σκοπεύουν να προτείνουν να προχωρήσουμε σε συνεργασία με άλλα μέλη, ευρύτερα δηλαδή για τους επόμενους μήνες. Thanks a lot. Ευχαριστούμε πολύ. Η Κάθεν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να πω ότι είναι καλό το γεγονός ότι έχουμε κοινή δήλωση με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Πρέπει να θεωρείται πρόοδος η ύπαρξη αυτής της κοινή δήλωσης. Ωστόσο ανησυχώ και οφείλω να το πω. Για ορισμένες από τις παραχωρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πορευόμενοι προς αυτή την κοινή δήλωση και θέλω να σας υπογραμμίσω δύο παραχωρήσεις. Σημείο 1,β. Οι ενισχύσεις αφαιρέγγιες ή προβληματικές επιχειρήσεις απουσία ε, σχεδίου αναδιάρθρωσης απαγορεύεται. Η Επιτροπή έχει παρουσιάσει βιομηχανική στρατηγική Γνωρίζουμε ότι στη νέα πράσινη συμφωνία θα ε, υποστείτουν τεράστια μετάβαση οι οικονομίες μας και αυτό θα έχει τεράστιο αντίκτυπο σε ορισμένε από τις βιομηχανίες μας και τις, ε, τους παραγωγικούς μας κλάδους. Δηλαδή δεν επιτρέπονται ενισχύσει όταν σε περίπτωση αναποφεύκτου κλεισίματος μιας επιχείρησης, παύσης, δραστηριότητες, δεν πρέπει να ε, ληφθούν καθόλου μέτρα. Δεν πρέπει να υπάρχουν καθόλου ενισχύσεις. Δεύτερον, ο ορισμός του δημόσιου φορέα. Με αυτή τη θέση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει στροφή 180 μοιρών. Πάντοτε στηρίζαμε ότι οι κρατικές επιχειρήσεις είναι δημόσιοι φορείς. Και η ερμηνεία αυτού του σώματος προσφυγών υπονομεύει την αποτελεσματικότητα των κανόνων ε, των ενισχύσεων. Γιατί κάνατε αυτή την κολοτούμπα. Μπορείτε να το, μας το εξηγήσετε. Θα επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο ε, εμείς στην Ευρώπη ε, αντιλαμβανόμαστε το δημόσιο φορέα και την ε, παροχή υπηρεσιών δημοσίου συμφέροντος, κοινή ωφελία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Μπιούτικοφερ παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για τις εξηγήσει και τις, την ενημέρωση που είχαμε. Καταρχάς θέλω να τονίσω αυτό που είπε ο κύριος Γεντονέ τελευταίο. Δηλαδή προσπάθειες επικοινωνίας, να έχουμε πρόσβαση σε όλους. Ασκούμε πίεση για μεταρρυθμίσεις. Το κατά πόσο θα πετύχουμε εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το πώς θα το προβάλλουμε αυτό, πώς θα το παρουσιάσουμε. Εάν αυτό το παρουσιάσουμε ως τρεις χώρες οι οποίες ε, συμμαχούν για να αντιμετωπίσουν την Κίνα και να εμποδίσουν την άνοδό της, πολύ φοβούμαι ότι θα δημιουργήσουμε περισσότερα προσκόμματα και δεν θα τύχουμε Αν όμω μπορούμε να το προβάλλουμε, ε, να προβάλλουμε αυτή τη μεταρρυθμιστική ατζέντα με έναν τρόπο ο οποίος ε, θα εξηγεί ότι είναι μια ατζέντα μεταρρυθμίσεων που θα ωφελήσει μια αναπτυξιακή διαδικασία η οποία θα δώσει δυνατότητα στον οποιονδήποτε να ανέβει ακριβώ διότι θα απαγορεύουμε τα μονοπόλια ή τις αθέμητες πρακτικέ, Εάν έτσι το πλασάρουμε, τότε θα κάνουμε τη διαφορά. Και Παρόλο που κατανοώ πλήρως ότι θέλουμε να έχουμε πρόσβαση στις ομονοούσες χώρες, το σημαντικότερο είναι να έχουμε πρόσβαση και να απευθυνθούμε στις μη ομονοούσες χώρες ε, για να τις παρεμποδίσουμε από το να σφύριλατήσουν τη δική τους συμμαχία. Θεωρώ ότι το πλαίσιο για αυτές τις μεταρρυθμίσεις είναι σχετικά αδύναμο. Από τη στιγμή που ο πρόεδρος Τραμπ αποφάσισε να υπογράψει την ε, συμφωνία φάσης 1, γιατί τελικά δεν πέτυχε τίποτα το οποίο θα μας αφορούσε εδώ, σε αυτούς εδώ τους χώρους και σε αυτό εδώ το βήμα, υπό αυτή την παραδοχή. Ίσως είναι καλό για τους Αμερικανούς γεωργούς να πουλάνε περισσότερα φασόλια, όμως οι σχετικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις έχουν αναβληθεί ε, και έχουν ε, ε, αποσταλεί στις καλένδες, έχουν μετατεθεί επαόριστον, μάλλον γιατί οι Κινέζοι δεν έχουν καθόλου όρεξη να διαπραγματευτούν συμφωνία φάσης 2 και αυτό μας το έχουν ήδη αναφέρει και μας έχουν ενημερώσει σχετικά. Άρα μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον ένα μέρος του περιεχομένου του κειμένου θα γίνει αντικείμενο σκληρής μάχης της διαπραγματεύσεις για τη δική μας συμφωνία η NCI. Και πιο συγκεκριμένα, για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τις κυρώσεις. Θα θυμάστε κύριε Πρόεδρε, ότι την τελευταία φορά που μας επισκέφθηκε το NPC στην ε, Διακοινοβουλευτική Επιτροπή μας είπαν οι Κινέζοι ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα ως τεχνο... για μεταφορά τεχνολογίας, γιατί κανέναν δεν αναγκάζουμε να κάνει business στην Κίνα και άμα θέλει τόσο πολύ κάποιος να κάνει business στην Κίνα, ε, τότε θα πρέπει να μας παραδώσει την τεχνολογία. Θα επιμείνουμε λοιπόν σε αυτά. Θα επιμείνουμε στις κυρώσεις για τους δημόσιους φορείς με βάση το CAI. Πόρο απέχουμε από οποιαδήποτε ε, συμφωνία αυτή τη στιγμή για τα SOE. Και επίσης, μέτρα κατά των ενισχύσεων. Αυτό είναι το τρίτο μου ερώτημα. Είναι έτοιμη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πει ναι. Θα ήταν καλή ιδέα να αντιστραφεί το βάρος της απόδειξης. Όσον αφορά στα μέτρα κατά των ενισχύσεων. Είναι έτοιμη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάει το κεφάλαιο 22β ε, του πρωτοκόλου του Κινέζικου και να το προβάλλει στον ΠΟΕ για να υπάρξουν κυρώσεις. Πόσα θέματα έχουν τεθεί συγκεκριμένα με την κινέζικη πλευρά για τη μεταρρύθμιση στον ΠΟΕ και ποια ήταν η απάντηση που έχουν δώσει. Ευχαριστούμε. Η Μαγή παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίαση και για την πρόοδο που έχει σημειωθεί. Είναι καλό αυτό, είναι θετικό. Μπορούμε να αποκαταστήσουμε την ισορροπία των ανταλλαγών μας ως προς τη μεταφορά τεχνολογίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας έδωσε τους στόχους. Ποια είναι όμως τα στάδια, πιο συγκεκριμένα, πώς έχει το χρονοδιάγραμμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι είναι θετική η υποδοχή όλων αυτών με από τα άλλα μέλη του ΠΟΕ και χαίρομαι γι' αυτό. Όμως ο τριμερής διάλογος ε, θα έχει αυτό το πλαίσιο ή το πλαίσιό του θα εξελιχθεί και θα υπάρξουν αλλαγές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ συνάδελφος από τη Σενεγάλη παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να μιλήσω για την ομάδα τριών υπουργών, τριών χωρών που θέλουν να κυριαρχήσουν στη βιομηχανία παγκοσμίω. Είναι μια ομάδα η οποία εργάζεται σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Έχουμε διεθνείς κανόνες στον ΠΟΕ. Αλήθεια. Κάποιοι συμμετέχοντες μίλησαν για ένα συγκεκριμένο αρχηγό κράτος. έγγραφα τα φυλάδια για ορισμένες χώρες και όχι για άλλες. Συνυπευθυνότητα υπάρχει και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Νομίζω ότι οι βιομήχανοι σε ορισμένε χώρε δεν θα πρέπει με τι πράξει του τελικά να αμεροληπτούν και να αποβαίνει αυτό σε βάρο άλλων χωρών και οι πολιτικοί του να το στηρίζουν και τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Μπόνταν παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να πω καταρχάς ότι χαίρομαι για την πρόοδο που έχει σημειωθεί για το θέμα της μεταφοράς τεχνολογίας. Αναρωτιέμαι για την προσέγγιση που θετούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας. Υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε ίσους κανόνες για όλους. Είναι ένα θέμα που αφορά όλες τις χώρες μέλη του ΠΟΕ. Ευχαριστώ. Ντένις παρακαλώ. Έχουμε κάποιες ερωτήσεις από ό,τι ακούσατε. Ναι, πολλές ερωτήσεις, πολλά σχόλια. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε κάποια εξ αυτών τουλάχιστον. Καταρχάς, για το θέμα του πεδίου εφαρμογής ε, και τη σωστή ισορροπία μεταξύ ε, αμυντική και επιθετική τάση. Προφανώ, ε, πολλέ επικράτειε έχουν διάφορε μορφέ ενισχύσεων και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΕΠΑ και η Ιαπωνία. Πώ λοιπόν όλα αυτά θα συνδυαστούν. Να πω και πάλι ότι η προσπάθεια γίνεται για να υπάρχει καλύτερη πειθαρχία μέσω διαφορετικής ε, μεταχείρισης διάφορων μέσων ενός αριθμού ιδιαίτερα επιζήμιων επιτοτήσεων που διαπιστώνουμε σε κάποιες χώρες. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλες ε, οι μορφές υποστήριξης κρατικής ε, είναι κακές ε, ή θα απαγορευτούν από επιπροσθετούς κανόνες. Στην παρούσα φάση το ESM είναι περίεργο, γιατί δεν υπάρχει το πράσινο κουτί, όλες οι μορφές επινίσχυσης είναι ίδιες, αλλά για να μπορέσουμε να αμφισβητήσουμε κάποιες Επιδοτήσει θα πρέπει να είναι σε χαμηλότερο ποσοστό, γιατί το σύστημα είναι μη αποτελεσματικό σε ό,τι αφορά την πειθαρχία που επικρατεί τελικά και γι' αυτό λοιπόν προσπαθούμε να βρούμε τη λύση σε ό,τι αφορά την πολιτική, σε ό,τι αφορά την κατάρτιση των σχετικών κανόνων. Κάνουμε υποχωρήσεις ε, αν θέλουμε να μεταφράσουμε τις δηλώσεις που γίνονται σε δεσμευτικούς κανόνες δεν μπορούμε να πούμε ότι ε, οι κατηγορίες ε, επιζήμιων επιδοτήσεων τα είδη των επιδοτήσεων που προβλέπονται στο 1β είναι είδη επιδοτήσεων τα οποία ήδη καλύπτονται από τι συμφωνίε ελευθέρου εμπορίου. Αυτό ισχύει και για εμά και για του εμπορικού μα εταίρου. Άρα, αυτή η κατηγορία των επιδοτήσεων καλύπτεται, γιατί είναι ήδη αποτελούν ήδη ένωμη τάξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα επιβάλλουν επιπλέον υποχρεώσει. Αλλά υπάρχουν, θεωρούμε, ήδη επιδοτήσεων που είναι ιδιαίτερα απαράδεκτε και επιβλαβείς και δεν θα ε, πρέπει να επιτραπούν στο διεθνές σύστημα. Και πιστεύουμε ότι συνεχίζουν να υφίστανται σε κάποια κράτη. Αυτή λοιπόν είναι μια απαγόρευση που για πρώτη φορά την ε, θέσαμε σε ό,τι φορά την Κορέα για το σώμα προσφυγών. Το δημοσίου, συγγνώμη, ε, σώματος του δημοσίου φορέα. Όσο έχουν τα πράγματα, ο δημόσιος φορέας ε, ορίζεται και ερμηνεύεται ως εξής. Δημόσιο σώμα, λοιπόν. Είναι πολύ δύσκολο να καταδείξουμε ότι μία σειρά οντοτήτων που δεν είναι η κυβέρνηση μεν, αλλά συνδέονται συχνά, στιχνά και στενά με την ε, κυβέρνηση μπορούν να παρέχουν επιδοτήσει. Ε, και για να είμαστε ξεκάθαροι, αυτό ισχύει για παράδειγμα σε ό,τι αφορά τι ε, κινέζικε τράπεζε κρατική ιδιοκτησία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο λοιπόν να αποδειχτεί ότι υπάρχει σχέση με, τις με την κυβέρνηση. Και μάλιστα τόσο στενή που θα μπορούσαν να είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής α, της συμφωνίας. αν θεωρήσουμε ότι πρέπει να αμφισβητήσουμε την παροχή των επιδοτήσεων αυτών. Αλλά ο νέος ορισμός του δημοσίου σώματος στο πλαίσιο αυτό δεν θα άλλαζε το οτιδήποτε σε ό,τι αφορά το πεδίο κάλυψης, το πεδίο εφαρμογής, ε, σε ό,τι αφορά τον ορισμό τώρα της επιδότησης, κατά δεν πρόκειται για προνόμια, η οικονομική ενίσχυση ή κάτι πιο συγκεκριμένο. Αυτό λοιπόν δεν αλλάζει στα πρόταση στο πλαίσιο του ASEM. Και γι' αυτό λοιπόν θεωρούμε ότι οι φορείς, οι δημόσιοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα κρατικές υπηρεσίες ηλεκτροδότησης και αερίου, θα είναι, θα πιο πολύ στα μέτρα πειθαρχίας από σε σχέση με το ESM, γιατί δεν πιστεύουμε ότι παρέχουν τέτοιες ε, επιδοτήσεις. Για τα ζητήματα που έθεσε ο κύριος Μπουτικόφερ, τα ερωτήματα. Εδώ η ιδέα είναι η εξή. Αν γίνει μια προσπάθεια για να αυξηθεί η πειθαρχία στο πλαίσιο του ΠΟΕ, του Διεθνούς ε, εμπορικού συστήματος για τις ε, επιδοτήσεις θα πρέπει να υπάρχει μια πειθαρχία που θα ισχύει οριζόντια σε όλες τις μεγάλες οικονομίες. Αυτό είναι το μοναδικό που θα έχει νόημα. Αυτό σημαίνει ότι στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων θα πρέπει ουσιαστικά να έχουμε τις μεγάλες ε, οικονομίες γιατί φυσικά μιλάμε για θέμα κλίμακας. Αν θέλουμε λοιπόν να υπάρχουν κεντρικοί, κεντρικοί κύκλοι, ομοκεντρικοί κύκλοι, έχουμε κάποιες χώρες οι οποίες είναι οι χώρες οι οποίες λίγο πολύ έχουν την ίδια αντίληψη και από αυτές θα ξεκινήσουμε. Αυτό δεν πρέπει να σημαίνει φυσικά ότι θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες και πέρα από τον στον αυτό των χωρών που είναι στο ίδιο επίπεδο και δεν θα πρέπει να συμπεριληφθούν και άλλες χώρες. Κατά πόσο η συμφωνία πρώτης φάσης ε, που προτάθηκε από τη ΣΥΠΑ και από την Κίνα κινείται προς την κατεύθυνση αυτή, δεν ξέρουμε ακόμα. Θα φανεί στο μέλλον. Είναι σαφές ότι η ΙΠΑ και η Κίνα δεν ε, έχουν ενσωματώσει τίποτα σε ό,τι αφορά τις βιομηχανικές αυτές επιδοτήσεις μέσα στη συμφωνία αυτή. Και ούτω το θέμα των βιομηχανικών επιδοτήσεων και της πειθαρχίας της σχετικής είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί σε διμερές επίπεδο, γιατί προφανώς όταν κάποιος πειθαρχεί, επιβάλλει πειθαρχία στον εαυτό του, σε ό,τι αφορά τις κρατητικές επιδοτήσεις που παρέχει στη χώρα του, αυτό ισχύει για όλες τις χώρες στο παγκόσμιο προσκήνιο, όχι μόνο για μια χώρα. Άρα λειτουργεί πολύ καλύτερα σε πολυμερές επίπεδο αυτή η ρύθμιση. Και σε ό,τι αφορά και όσα έχουν συμβεί στις ε, συμφωνίες ελευθερίου σε ό,τι αφορά το θέμα των επιδοτήσεων. Όλα αυτά λειτουργούν λοιπόν καλύτερα σε παγκόσμιο προσκήνιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα αυτά δεν μπορούν να καθοριστούν και σε διμερές επίπεδο. Άλλα στοιχεία πειθαρχία, τα οποία όμω ενδεχομένω να μην συνδέονται απαραίτητα με τι επιδοτήσει σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, το κανονιστικό πλαίσιο για τι ε, εταιρείε, ε, τι κρατικέ. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ρυθμίζεται πιο εύκολα σε διμερές επίπεδο, γιατί είναι όντω ε, ένα φαινόμενο. Το ότι όταν υπάρχουν κρατικέ επιχειρήσει στα σύνορα κοντά τα συνοριακά, αυτό έχει συνέπειε για τι κοντινέ χώρε. Σε ό,τι αφορά τι τεχνολογικέ μεταφορέ τώρα, μπορεί να σκεφτούμε διαφορετικού κανόνε είτε σε διμερέ επίπεδο είτε σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό το θέμα είναι πολύ περίπλοκο γιατί έχει να κάνει και με τι ε, όρου πρόσβαση στην αγορά και διάφορα στοιχεία τα οποία μπορεί να τύχουν διαπραγμάτευση σε μια καθολική και σε βάθος συμφωνία για τις επενδύσεις, σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τις απαιτήσει και τις κοινοπραξίες ιδιωτικού και δημοσίου κλάδου και άλλα είδη πειθαρχία σε ό,τι αφορά την πιστοποίηση, την αντιδότηση κτλ. Και αυτό αναφέρεται και σε αυτά που είπε η συνάδελφος η κυρία Βεντρέν. Τα επόμενα βήματα θα είναι δύσκολα, γιατί προφανώς θα χρειαστεί να συνδυαστούν διάφοροι παράγοντες από διάφορα είδη διεθνών κανόνων. Αυτό δεν ισχύει για τις, βιοσυ... για τις ε, βιομηχανικές επιδοτήσεις, γιατί στις βιομηχανικές επιδοτήσεις καταφέραμε να, σημειώσουμε σημαντική πρόοδο σε ό,τι αφορά τους πιο εκτενείς κανόνες, γιατί έχουμε μία βάση εκκίνηση σε ό,τι αφορά τον ΠΟΕ. Όταν υπάρχει λοιπόν μία ενιαία γραμμή μπορούμε να βασιζούμε σε αυτή. Σε ό,τι αφορά τη μεταφορά τεχνολογίας, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα. Ε, εδώ λοιπόν θα υπάρξει συνέχιση των προσπαθειών. Για να δούμε τι έχει γίνει ήδη στον τομέα των επιδοτήσεων και να δούμε ποιες, ε, ποιες θα ήταν οι τομείς που θα μπορούσαμε να εργαστούμε. Νομίζω και ελπίζω να κάλυψα τις πιο πολλές ερωτήσεις. Όπως σας είπα για το θέμα της ε, εξέλιξης του μορφότυπου, τελευταίο σημείο. Θέλουμε να ξεκινήσουμε με ομόκεντρους κύκλους. Πιστεύουμε ότι στην τελική ανάλυση όλοι οι βασικοί φορείς παροχή επιδοτήσεων θα πρέπει να βρεθούν στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων, αν θέλουμε να πετύχουμε κάτι. Αλλά βαθμιαία μπορούμε να λειτουργήσουμε. Καταρχάς, να ξεκινήσουν κάποιε διαπραγματεύσει διεθνεί για την πειθαρχία αυτή, για τις επιδοτήσει. Στη συνέχεια θα πρέπει να αποφασίσουμε με επαρκή ομάδα διαπραγματευτών πώ θα διαπραγματευτούμε τις μεμονωμένες διατάξεις βάσει και της ε, τρέχου, του τρέχοντος συστήματος ε, πιστοποίησης και διαδότησης. Πρόκειται λοιπόν για το επόμενο βήμα. Δεν έχουμε, δεν είμαστε ακόμα στη φάση αυτή, αλλά θέλουμε στους επόμενους μήνες να αναπτύξουμε τη διαδικασία αυτή, να κινηθούμε προς την κατεύθυνση αυτή και σταδιακά να διευρύνουμε αυτό το ομόκεντρο κύκλο, όπως σας είπα, ομοειδεατών. Ελπίζω να κάλυψα έτσι τα διάφορα στοιχεία που αναφέρατε. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι βέβαιος ότι δεν είναι η τελευταία φορά που θα συζητηθεί αυτό το θέμα. Την μετα... Ε, ε, αναγκαστική μεταφορά τεχνολογίας κλπ. Λοιπόν, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η συζήτηση ε, επί του 20. Το 21 διάφορα. Τίποτα. Η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει στις 10.